Σχέδιο λοιπόν ημερήσιας διάταξης ε, στα αγγλικά σας έχει σταλεί στις 22 Νοεμβρίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Έγκριση των πρακτικών. Φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που δεν βλέπω κανέναν να, ε, να αντιδρά, θεωρούνται εγκεκριμένα. Την ε, έδειξη <clears throat> για σήμερα και αύριο θα τη βρείτε και ε, στο ε, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σήμερα στις 6.30 θα έχουμε ένα κοκτέιλ για τις χριστουγεννιάτικες ευχές. Πριν περάσουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας ε, διάταξης, θέλω να σας πω, για όποιον ενδιαφέρεται, ότι αύριο στην Επιτροπή Προπολογισμών στο σημείο 8 της Υπηρεσία διατάξεως έχει προβλέψει ανταλλαγή απόψεων για την τροποποίηση των δημοσιονομικών προοπτικών. Και η ε, κυρία Ριβελίνη, σαν εισηγήτρια, ε, θα είναι παρούσα βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού. Περνάμε στο σημείο 4 του, ε, Σχεδίου Ημερησίας Διατάξεως, απαλλαγή 2009, Γενικός Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκή Ένωση, τμήμα 3, Επιτροπή. Να σας πω λοιπόν ότι πρώτα θα μιλήσει ο υπεύθυνος ε, του ελεγκτικού ε, συνεδρίου, συγγνώμη, η κυρία Κάριο Λάινε, και μετά θα δώσουμε τον λόγο ε, στον Επίτροπο Χαν για πέντε λεπτά ε, και ε, μετά στον επόμενο Επίτροπο Άντορ για άλλα πέντε λεπτά. Μετά, αφού πάρει το λόγο ο κύριος Χατζημαρκάκης, θα ξεκινήσουμε να δίνουμε το λόγο στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων, με πρώτο τον εκπρόσωπο του ΕΛΚ, λόγο μεγέθους. Θα δώσουμε πρώτα το λόγο λοιπόν στην κυρία Κάλιο Λάιν. Thank Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αξιότιμοι κυρίε και κύριοι βουλευτέ, κύριοι επίτροποι. Θα ήθελα να σα παρουσιάσω την ειδική αξιολόγηση της πολιτικής συνοχής Το δημοσιονομικό έτο 2009 ήταν το πρώτο κατά το οποίο το δείγμα του συνεδρίου, του ελεκτικού συνεδρίου, σχετιζόταν με τις ε, αποζημιώσεις για την περίοδο 2007-2013. Για το 2009 λοιπόν το τελευταίο έτος κατά το οποίο μπορούσαν να κατεβληθούν από ζημιώσεις για την περίοδο μέχρι το 2006 πριν από το οριστικό κλείσιμο των προγραμμάτων. Το 2009 η χρηματοδότηση πολιτικής συνοχής από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανερχόταν σε 35,5 ε, δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 14,1 δισεκατομμύρια ευρώ τις δικούσαν σε αποζημιώσεις που καταβάλλονται στα κράτη-μέλη ε, για την, προγραμματική, για την νέα προγραμματική περίοδο και 11,3 δισεκατομμύρια για την περίοδο 2000-2006 δηλαδή ε, προχρηματοδότηση στο πλαίσιο της περίοδου 2007-2013 ήταν τα υπόλοιπα 11,3 ευρώ. Ο έλεγχος λοιπόν ο νομικού του Εθνικού Συνεδρίου ε, για τη συνοχή του 2006, ε, το 2009 εξέτασε την νομιμότητα και ε, κανονικότητα των προσωρινών και οριστικών πληρωμών για, το, για τα ταμεία το 2009 την ε, συμμόρφωση με κύριες προδιαγραφές για, τη διαχείριση και τα, συστήματα, για τα συστήματα ελέγχου και διαχείριση για το 2007-2013 και την ε, επεξεργασία και κατάθεση των σχετικών πορισμάτων για απόδοση καταβληθέντων και δημοσιονομικές διορθώσεις από τα κράτη-μέλη, 180 μεσοπρόθεσμες ε, πληρωμές ε, επικυρώθηκαν, 64% των πληρωμών σε σχέδια ε, αποδείχθηκε ότι δεν είχαν κανένα σφάλμα. Για το 2008 και 2007 αντίστοιχα τα ποσοστά ήταν 57% και 46%. 36% των σχεδίων είχαν ένα ή περισσότερα σφάλματα. 47% του συνολικού αριθμού ε, σφαλμάτων μπορούσαν να υπολογιστούν ποσοτικά και έτσι υπολόγισε το συνέδριο το ε, πιθανότερο ποσοστό σφάλματος κάπου στο 5%, λίγο πάνω από το 5%, δηλαδή αντίστοιχα με αυτό του έτους 2008. Ε, ταυτόχρονα η υπεραπόδοση ποσών ήταν περίπου στο 3% για την ομάδα της συνοχής. Πρόκειται για στατιστικά στοιχεία τα οποία προκύπτουν από το μάλλον πιθανό σφάλμα και μας επιτρέπουν να πούμε ότι 95% ε, των πληρωμών είχαν γίνει ικανοποιητικά. Αυτό είναι το λεγόμενο κατώτατο ποσοστό, η όριο φάλματος. Το οποίο έτσι ε, υπολογίζεται όπως είπα σε 5% ενώ για το 2008 ήταν στο 11% τουλάχιστον. Εάν τώρα υπάρχει πραγματική βελτίωση ως προς τη συνοχή στις δαπάνες συνοχής ε, και κατά πόσον αυτό προκύπτει από, ε, ως αποτέλεσμα του πληθυσμού ή των μεσοπρόθεσμων ε, πληρωμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιθανόν να συμβάλλουν και οι δύο αυτοί παράγοντες. Οι περισσότερες επιστροφές ποσών έγιναν το 2009 σε σχέση με το 2007-2013 σχετίζονταν δηλαδή με την περίοδο 2007-2013, ο έλεγχος και οι προβλέψεις ελέγχου για τη νέα περίοδο ε, από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχαν ενισχυθεί και αντίστοιχη είχε ενισχυθεί και η περιγραφή του συστήματος και οι δηλώσει συμμόρφωση των κρατών μελών. Οι δε προληπτικοί έλεγχοι αποτελούν το κύριο και ουσιαστικό στοιχείο του συνολικού πλαισίου ελέγχου. Έτσι λοιπόν, είχαμε καλή, ε, καλά αποτελέσματα και οι πληρωμές ε, του 2009 μπορούμε να πούμε ότι είχαν αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Επιπλέον, μεγάλο ποσό των επιστροφών για το 2009 σχετιζόταν με τις δημοσιονομικές με τα μέσα μάλλον δημοσιονομικής μηχανικής που σημαίνουν περιορισμένες ε, απαιτήσει πληρωμών και ως εκ τούτου χαμηλότερο ποσοστό σφάλματος ή χαμηλότερο κίνδυνο σφάλματος. Ο όγκο λοιπόν των πληρωμών μέσω των συστημάτων είναι σχετικά χαμηλός και έτσι η διαχείριση και ο έλεγχος για τα προσεχή χρόνια παραμένει ικανοποιητικό, καλύτερος. Και συνολικά βλέπουμε ότι και τα κράτη-μέλη είχαν συνείδηση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων για την περιοδο 2006 2000-2006. Και έτσι είχαμε και το κόστος το οποίο δεν ήταν πιθανόν ε, να ενταχθεί στην αποζημίωση και τις ε, εσφαλμένες καταγραφές της δημόσιας προμήθειας ως κύρια σφάλματα. Η μη τήρηση λοιπόν των κύριων προδιαγραφών ε, για ε, τις δημόσιες ήταν το 43% όλων των ποσοτικά υπολογίσιμων σφαλμάτων, δηλαδή 3 τέταρτα των κατεκτήμησιν ποσοστών σφάλματος το 30 περίπου των σφαλμάτων που διαπιστώνει στο, στο ελεγκτικό του δείγμα το ελεγκτικό συνέδριο θα μπορούσαν να διορθωθούν από τα κράτη-μέλη, από τις αρχές τους δηλαδή, πριν από την πιστοποίηση της σχετικής δαπάνης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ελεγκτικό συνέδριο σημειώνει ότι 16 ε, συστήματα τήρησης και ελέγχου στα κράτη-μέλη συμφωνούν με τις προδιαγραφές του ρυθμιστικού πλαισίου του 2007-2013. Αυτά τα 16 λοιπόν συστήματα διαχείρισης και ελέγχου έχουν ήδη πάρει τη σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο έλεγχο του ηλεκτρικού συνεδρίου δείχνει ότι 11 εκ των 16 αυτών των συστημάτων που ελέγχθηκαν αποδεικνύουν πως οι επαληθεύσει από τις αρχές διαχείρισης εν μέρη μόνο συμμορφώνονται με τι ε, προδιαγραφέ του κανονισμού. Επιπλέον σημειώνει το ελεγκτικό συνέδριο ορισμένε καθυστερήσει ω προ την υλοποίηση τη εθνική στρατηγική ελέγχου και στρατηγικέ διαφορέ στο βαθμό με τον οποίο πραγματοποιούνται αυτέ οι δραστηριότητε δημοσιονομικού ελέγχου από τι αρχέ μέχρι το 2000, 2009. Συνολικά, τα συστήματα εποπτεία και ελέγχου για την περίοδο 2007-2013 εν μέρη ήταν ε, σύμφωνες με τις κύριες προδιαγραφές ε, του ελεκτικού κανονισμού. Όπως και στα προηγούμενα χρόνια ε, το ελεκτικό συνέδριο εξέτασε τα συστήματα των κρατών μελών 2000-2006 για να επαληθεύσει και να επεξεργαστεί σφάλματα που είχαν ήδη εντοπίσει οι ελεγκτικέ αρχέ των κρατών μελών και αντίστοιχα κατέθεσαν τι προτάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι λοιπόν τα συστήματα εντοπισμού και διόρθωσης φαλμάτων ε, που χρησιμοποίησαν τα κράτη-μέλη την περίοδο 2000-2006 φαίνεται να ήταν αποτελεσματικά. Τα συστήματα για την ε, καταγραφή των ε, επιστροφών, τη απόδοση των χρημάτων και τη σχετική διόρθωση των χρημάτων που ε, υποβάλλονταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν εν μέρη ικανοποιητικά. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν λάμφανε πάντοτε τι επαρκεί πληροφορίε ή αξιόπιστε πληροφορίε για τη σχετική διόρθωση και απόδοση των κονδυλίων από τα κράτη-μέλη. Και εν τέλει ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενθαρρύνει τι εθνικέ αρχέ σε μια πιο πιστή τήρηση αυτών των μηχανισμών πριν από την πιστοποίηση των σχετικών δαπανών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η υποκατάσταση των δαπανών από τις μη δικαιούχες σε δικαιούχες δεν μπορεί να είναι αυτόματη, δεν μπορεί αυτόματα δηλαδή να χορηγηθεί η έγκριση για δικαιούχες, οι επιλέξιμες πιστώσεις και τα κράτη-μέλη. Και στα επόμενα χρόνια που θα αυξηθούν τα σχετικά κονδύλια, η κατάσταση είναι πιθανόν να καταστεί ακόμη πιο δύσκολη. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε την εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου για το εισαγωγικό της σημείωμα. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής, κύριο Χάν, για πέντε λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, του Ελεκτικού Συνεδρίου. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα καταρχά να ευχαριστώ την κυρία Καρολάιτ αλλά και τα άλλα μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου και του προσωπικού του και το προσωπικό του για την συνεργασία και την επικοινωνία σχετικά με την πολιτική συνοχή θα ήθελα <clears throat> να πω ότι για την έκθεση και γενικότερα το πρόγραμμα δράσης για το 2008 ε, που παρακολουθήσαμε, είχα πει ήδη από την αρχή ότι ήμουν αισιόδοξο ότι η κατάσταση σε σχέση με την πολιτική της συνοχής θα είναι θετική. Η σημερινή συζήτηση αποδεικνύει και η έκθεση βέβαια αποδεικνύει ότι έχουμε μπει στο δρόμο. Η σημαντικότερη βελτίωση σημειώνεται ακριβώς στην ποσοτική μέτρηση, τα ποσοτικά μετρήσιμα ποσοστά ασφάλματος. Εδώ νομίζω μπορούμε να πούμε ότι και η Επιτροπή αλλά και το Ελεκτικό Συνέδριο όπως ε, και η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού μπόρεσαν χάρη στη συνεργασία την αντιπαράθεση απόψεων, την αμοιβαία ενημέρωση να διαδραματίσουν το ρόλο που τους αρμόζει για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης. Και χωρίς να μπορώ να μιλήσω ακόμη για συγκεκριμένη τάση, είμαι αισιόδοξο ότι όντω στα επόμενα χρόνια θα συνεχιστεί αυτή η θετική εξέλιξη. Έχουμε επίση σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με την ε, μείωση, περαιτέρω μείωση του ποσοστού σφάλματος στο δείγμα, δύο τρίτα δηλαδή των ε, ε, ελεγχθησών συναλλαγών δεν έχουν κανένα είτε ποσοτικά είτε μη ποσοτικά μετρήσιμο σφάλμα. Νομίζω ότι αυτό δείχνει πως μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματική πλέον αυτή η διαδικασία του, της συνοχής, λειτουργεί δηλαδή πολύ αποτελεσματικά η συνοχή χωρίς φάλματα και θα ήθελα να πω, δεδομένων και των διαφόρων ε, δημοσίων συζητήσεων, αναφορών στον τύπο κτλ, ότι μπορεί να μην ήταν πάντα επιτυχημένη η επιλογή των δειγμάτων στο παρελθόν. Τα δείγματα μερικές φορές ε, τα όριζαν τα κράτη ή οι περιφέρειες και ήταν ε, μερικές φορές και ε, λόγος ανησυχίας η επιλογή δειγμάτων ε, Φερρυπίν από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, τον Εμένο Βασίλειο σε έναν βαθμό, την Πολωνία, την Τσεχία, την Εστονία, την Φινλανδία, τη Γαλλία, την Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, δηλαδή σχεδόν όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου βλέπουμε πως η ετήσια έκθεση για τη λειτουργία της ε, πολιτικής συνοχής αποδίδει στην σχετική γενική διεύθυνση το βαθμό α κεφαλαίο. Επίσης δεν πρέπει να λησμονούμε ότι το ελεκτικό συνέδριο έχει δώσει σαφείς υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επεξεργάζεται τις εκθέσεις για τα επόμενα χρόνια και αξιολογήσει το πρόγραμμα δράσης θετικά. Ε, λόγοι τη σχετική βελτίωση. Νομίζω ότι μπορούμε να αναπτύξουμε λίγο περισσότερο το τομέα αυτό, το κεφάλαιο αυτό των λόγων. Ναι, βλέπουμε ότι οι δράσεις έφεραν αποτελέσματα. Έχουμε μια καλή αξιολόγηση και επαλήθευση των ε, στρατηγικών που έχουν επιλεγεί, ιδιαίτερος δηλαδή την ε, επαλήθευση πριν από την εκκίνηση των προγραμμάτων. Αυτή η μέθοδος βλέπουμε ότι αποδεικνύεται πολύ ε, αποδοτική και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίμησε προληπτικά να δρά, να ενημερώνει, να καταρτίζει τις αντίστοιχες αρχές των κρατών μελών, ε, πράγμα το οποίο τηρήσαμε αυστηρά. όπως άλλωστε τηρήσαμε πολύ αυστηρά και τον κανόνα της άμεσης διακοπής διάθεση των κονδυλίων, όπου παρουσιάζονταν, διαπιστώνονταν παρατυπίες ή ε, όχι ικανοποιητική ε, λειτουργία των προγραμμάτων. 43 ήταν για το έτος 2010 οι διακοπές ροής των κονδυλίων. Όχι παύσεις, αλλά μόνο διακοπές. Και νομίζω ότι αποδεικνύεται πως ήταν αποτελεσματικό το σύστημα αυτό δεδομένων των στοιχείων που έχουμε να διαπιστώσουμε σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν θα σα αναφέρω τώρα αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία, αν χρειαστεί θα επανέλθουμε στη συζήτηση. Και χωρί να θέλω βέβαια να ε, πενεύω το σπίτι μου, θα έλεγα ότι είμαστε ικανοποιημένοι, θα έλεγα ότι μπορούμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο, ε, να μειώσουμε δηλαδή ακόμη περισσότερο το ποσοστό αυτού του σφάλματο. Έχουμε ε, μια στρατηγική ε, για την περίοδο 2000, 2006 την οποία εξετάζουμε και αξιολογούμε Προφανώς και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων θα προκύψουν και άλλες παρατηρήσεις. Ε, και για να ολοκληρώσω κύριε και κύριοι, για την προσεχή περίοδο προτείνουμε έχουμε προτείνει ήδη μια μεταρρύθμιση η οποία πιστεύω ε, αποστέλει και σαφή μηνύματα για το πώς θέλουμε να προχωρήσουμε στο μέλλον. Θα ήθελα επίσης να πω ότι από τις αντιδράσεις που βλέπουμε στον τύπο ήδη σήμερα ε, θεωρώ ότι αποδεικνύεται πως μπορούμε να δείξουμε πώς η Ευρώπη μπορεί να αναπτύσσεται με τα κοινά προγράμματα, με την βελτίωση των προδιαγραφών, την ανύψωση σε, όλα, σε όλη την επικράτεια της Ένωσης του επίπεδου και αυτοί οι έλεγχοι αποδεικνύουν πως η ε, τήρηση των προδιαγραφών σημαίνει ότι και τα κράτη-μέλη μπορούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον ε, Επίτροπο Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, Λάσλο Άντορ. Παρακαλώ, κύριε Άντορ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου και εκπρόσωποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κυρίες και κύριοι, όπως και ο συνάδελφός μου, ο τύπος Γιωχάννης Σεχάνα, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην κυρία ε, Κάλιου Λάιτ, καθώς επίσης ε, και στον κύριο Καλδέρα για την ε, σαφή παρουσίαση της ετησία εκθέσεως για το 2009. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την πραγματογνωμοσύνη την οποία έδειξαν στην προετοιμασία της έκθεσης αυτής. Όσον αφορά λοιπόν την εφαρμογή του προϋπολογισμού, λάβαμε υπόψη μας ε, πάρα πολύ σοβαρά και τις προτάσεις ε, του ε, Ελεκτικού Συνεδρίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο σύνολό της η έκθεση 2009 καταδεικνύει, καταδεικνύει βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, σε διάφορους δείκτες μάλιστα, ας πούμε μέσω ε, της ε, ετήσιας έκθεσης δραστηριότητας των γενικών διευθύνσεων που πλέον έχουν βαθό α, επίσης τα οικοσυστήματα, επίσης όπως σαφώς αναφέρονται στους εγχρώμους κανόνες, ε, συγγνώμη, πίνακες. Ε, οι τυχαίες δειγματοληψίες βεβαίως ε, μπορεί να δώσουν και κάποια ε, μικρή διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων και τα επόμενα χρόνια. Αλλά ούτως ή άλλως είναι αναμφισβήτητα τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Λίγο πριν το 2010 ε, είχα την δυνατότητα να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα του σχέδιου δράσης του 2008. Ε, ευελπιστούμε και βασιζόμαστε σε συγκεκριμένες συγκεκριμένα αποτελέσματα και ενδείξεις ε, ευελπιστούμε λέγω ότι ήδη το 2013 θα δούμε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως δε όσον αφορά το κοινωνικό ταμείο έχει εφαρμόσει αυστηρότερη πολιτική όσον αφορά ε, την ε, πάυση πληρωμών για οποιαδήποτε προγράμματα ε, κατέδειξαν ασθενή διαχείριση. Επίσης είναι γεγονός ότι κάποιες χώρες δεν έχουν επιλογή, επιλεγεί από το ελεγκτικό συνέδριο ε, και αυτό γιατί λόγω σαφών αδυναμιών και για να προστατέψουμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων φορολογουμένων εμείς εξ αρχής ε, σταματήσαμε τις πληρωμές. Ευελπιστούμε ότι βασιζόμενοι και στις προτάσεις ε, του ελεγκτικού συνεδρίου θα βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την αποτελεσματικότητά μας και θα μειώσουμε το περιθώριο λάθους. Αυτό δεν σημαίνει ότι ε, θα αυξήσουμε υπερβολικά τον αριθμό των ελέγχων, αλλά θέλουμε η έλεγχη να είναι πιο αποτελεσματική. Το σημαντικό είναι ε, να εφαρμοστεί πλήρως ε, η προσέγγιση του ενιαίου και ε, μοναδικού ελέγχου, οικονομικού ελέγχου. Τα χρήματα τα οποία δαπανώνται προς αυτό το σκοπό έχουν αυξηθεί. Όσον αφορά το κοινωνικό ταμείο, το μεγαλύτερο πρόβλημα, η μεγαλύτερη αδυναμία είναι η επιλεξιμότητα έχουμε ήδη ε, εφαρμόσει μέτρα ε, απλούστευσης τα οποία θα βοηθήσουν να μειωθεί ακόμα περισσότερο το περιθώριο λάθους αλλά βεβαίως ταυτοχρόνως θα πρέπει να απλουστευθούν ε, και σε εθνικό επίπεδο οι κανόνες επιλεξιμότητας. Κατά την άποψή μου όμως η απλούστευση δεν ταυτίζεται με την επιλεξιμότητα. Ας πούμε, εγώ θα ήθελα και με τη δικιά σας βοήθεια να ε, δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να έχουμε περαιτέρω απλούστευση του, των κανόνων ε, στο μέλλον. Αλλά φυσικά ε, με την, μείωση, με την αύξηση της αποτελεσματικότητας δεν μειώνονται αυτόματα τα λάθη. Οπωσδήποτε θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αυστηρότητα τους υπάρχοντες ελέγχους. Τέλος, το ελεγκτικό συνέδριο αναφέρθηκε στις ε, δημοσιονομικές διορθώσεις ε, και στα προβλήματα σε εθνικό επίπεδο. Ε, φαντάζομαι και ορθώς ότι πολλοί μεταξύ ημών θεωρούν το πρόβλημα αυτό πολύ μεγάλο. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να σας πω, παρότι δηλαδή έχουν ήδη βελτιωθεί τα πράγματα, δεν είμαστε ακόμα ικανοποιημένοι. Επομένως εστιάζουμε την προσοχή μας και τις προσπάθειές μας προς την κατεύθυνση αυτή έτσι ώστε να έχουμε απολύτως αξιόπιτα στοιχεία. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η εκτέλεση του προϋπολογισμού προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συμμόρφωση με τους κανόνες εφαρμογής είναι οπωσδήποτε απαραίτητη αλλά δεν είναι επαρκής. Τα χρήματα των πολιτών, των φορολογουμένων θα πρέπει να τα διαχειριζόμαστε σωστά αλλά ταυτοχρόνως και με την μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. Επομένως θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας ε, στην μεγιστοποίηση της προστιθέμενης ευρωπαϊκής ε, ε, αξίας και κυρίως όσον αφορά την πολιτική συνοχή. Κατά αυτή την έννοια θα ε, πρέπει να κάνουμε περισσότερες ε, προσπάθειες βελτίωσης όσον αφορά την ποιότητα των δαπανών καθώς επίσης και όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος 2020. Εγώ βεβαίως είμαι απολύτως διαδεθειμένος να ε, συζητήσω οποιασδήποτε μεθόδου βελτίωσης της ε, ε, χρήσης του Ταμείου και αυτό για τους επόμενους μήνες ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία νομοθετικής ε, τροποποίησης ε, του δημοσιονομικού πλαισίου και το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει ε, και την πρότασή της για την επόμενη γενιά των διευθυντικών ταμείων. Νομίζω ότι αυτή θα είναι μια καλή ευκαιρία για να προωθήσουμε έτσι περαιτέρω τα στοιχεία τα οποία ανέφερε το ελεγκτικό συνέδριο και βεβαίως ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμβάλλει τα μάλα ε, στην ε, διαδικασία αυτή και περιμένω και τη δική σας άποψη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Χατζημαρκάκη ως εισηγητή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστώ την κυρία Κανουλάιτα για την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και να ευχαριστήσω επίσης και για το πρώτο κεφάλαιο ιδιαίτερος είναι το καθοριστικό εκείνο το οποίο μας λέει εάν η πολιτική των ε, πληρωμών των δαπανών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αξιόπιστη, δεν μπορούμε να την εμπιστευόμαστε δηλαδή ως εμείς, εμείς ως αρμόδια αρχή για τον προπολογισμό. Είμαστε ευγνώμονε λοιπόν για αυτό το συγκεκριμένο κεφάλαιο στην, ε, στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Για τη συνοχή και οι δύο επίτροποι, οι οποίοι είναι αρμόδιοι, συναρμόδιοι στο θέμα αυτό, βλέπουμε ότι έχουν εργαστεί στενά, σε στενή συνεργασία με το Ελεγκτικό Συνέδριο και άρα μπορούμε να είμαστε πολύ πιο βέβαιοι για την αποτελεσματικότητα αυτή τη δράση, ε, γιατί βέβαια είναι πολύ καλύτερο να υπάρχει η συνεργασία, στενή συνεργασία κατά τον προσδιορισμό του δείγματος από μια απλή επικοινωνία. Θα ήθελα επίσης καταρχάς να ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την αναδρομικότητα που ε, ανέπτυξε για, την, ε, για τον υπολογισμό των προβλημάτων δεν ξέρω εάν αυτή η ευτυχή σύμπτωση που αναφέρατε νωρίτερα είναι σύμπτωση ή αν είναι αποτέλεσμα μια συγκεκριμένη πολιτική, αλλά πάντω εμεί βλέπουμε από πλευρά του Κοινοβουλίου ότι όντω οι προσπάθειε τι οποίε ανέλαβε να υλοποιήσει ο επίτροπο Κάλλα συνεχίζονται και τώρα και φέρνουν αποτέλεσμα και από τον Επίτροπο Σεμέτα επίση. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση για το ότι αναφέρει ονόματα συγκεκριμένα. Στο Annual Accounts of the European Union για πρώτη φορά στου ετήσιου λογαριασμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση λέει συγκεκριμένα ποιο κράτο μέλο ε, παραβιάζει ποια αρχή ή υστερεί έναντι τίνο κανόνα. Αυτό είναι μια νέα βάση για μα. Μπορούμε έτσι καλύτερα να καταλάβουμε τη δουλειά σα και επίση μπορούμε να εντοπίσουμε πολύ πιο ξεκάθαρα τι παραλήψει των κρατών μελών. Στον τομέα τη συνοχή έχουμε ένα στοιχείο, και εδώ δυστυχώ θα πρέπει να περάσω στα αρνητικά στοιχεία. Ένα στοιχείο λοιπόν, ένα νούμερο, το οποίο δημοσιεύεται εδώ στους ετήσιους λογαριασμούς, μεγάλο νούμερο για την περίοδο 94 με 2006, μεγάλο όπως είπα νούμερο, ότι εσφαλμένα διατέθηκαν 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το συγκεντρωτικό ποσό. Το ποσό δηλαδή των κονδυλίων που έλαβαν αδικαιολόγητα τα κράτη-μέλη. Από αυτά, μόνο 709 εκατομμύρια ευρώ επεστράφησαν. Και εδώ ακριβώς εντοπίζεται το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλες δαπάνες, μεγάλα ποσά, ποσά τα οποία προέρχονται από τον φόρο που πληρώνει ο Ευρωπαίος φορολογούμενος, που μοχθεί, που εργάζεται σκληρά και που αποδεικνύεται ότι τα χρήματα αυτά πήγαν αδικαιολόγητα σε κάποιον εθνικό κορβανά και επιστρέφει και μόνο μικρό ποσοστό από αυτά στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αυτό το πρέπει να το εντοπίσουμε τώρα. Δυστυχώ αυτό συνεχίζεται. Σημαντική αλλαγή δεν βλέπουμε. Η τάση μπορεί να παρουσιάσει κάποια εξέλιξη, αλλά στη λογική δεν βλέπουμε αλλαγή. Και γι' αυτό χαίρομαι που βλέπω ότι και οι δύο επιτροποί, αλλά ιδιαίτερα θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Άντορ για την ε, πρακτική που έχει εισαγάγει, δηλαδή την διακοπή των πληρωμών που επέλεξε ως λύση. Είπατε ότι δεν είναι διακοπή αλλά είναι πάυση. Ε, δεν είναι πάυση είναι διακοπή. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει το ότι δεν καταβάλλονται τα ποσά αυτά. Είναι νομικό ζήτημα το αν πρόκειται για διακοπή ή για πάυση. Πάντως έχει πρόβλημα ως προς τις πληρωμές ένα κράτος μέλος. Και αυτό ακριβώς ήθελα να ε, επισημάνω κύριε Άντος. Ότι δηλαδή προγράμματα, τα σχέδια μάλλον τα οποία είναι ελλειπή, ότι, που δεν είναι αξιόπιστα, σταματούν να χρηματοδοτούνται άπαξ και δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Και άμα δεν ε, χρηματοδοτηθούν όπως πρέπει δεν μπορούν να μπουν και στο δείγμα κλπ. Σα συγχαίρουμε λοιπόν γι' αυτό. Ακόμα όμως δεν βλέπουμε ακριβώς πρόγραμμα δράσης. Πότε θα αρχίσετε να υλοποιείτε αυτές τις διακοπέ. Δηλαδή ε, υπάρχουν αυτοματισμοί στο παρελθόν ξέραμε, επί παραδείγματι, ότι σε μεγάλες ε, περιπτώσεις προβλημάτων στην ε, ε, ενίσχυση της υπαίθρου, τις περιφερειακές πληρωμές, στην συνοχή γενικά, υπήρχε μια προσπάθεια από τις πολιτικές αρχές της περιφέρειας που έρχονταν στις Βρυξέλλες, που προσπαθούσαν με τον Επίτροπο, να προσπαθήσουν να διεκδικήσουν ένα μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο, να μην διακοπούν οι πληρωμές. Τώρα όμως Ίσως θα έπρεπε να υπάρχουν αυτοματοποιημένες διαδικασίες διακοπής των πληρωμών. διακοπής των πληρωμών. Γι' αυτό θα ήθελα να έχουμε μια πιο συγκεκριμένη, ε, ένα πιο συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης, ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και μεταξύ μας, ε, θα επέβαλε αυτόματα τη διακοπή αυτών πληρωμών. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να σα ζητήσω, θα ήταν να επιδείξετε μεγαλύτερη απευθυνότητα απέναντι στι δικέ μα ευθύνε και αρμοδιότητε στο Κοινοβούλιο. Και θα ήθελα εδώ πάλι να καλωσορίσω εδώ να χαιρέτησω τον συνάδελφο Γιάνν Μίλτζερ, ο οποίο χρόνια τώρα και δεν ήταν ο μόνο, αλλά ήταν ε, μεταξύ των πρωτοπόρων που αγωνίστηκαν από πλευρά τη ομάδα μου έναντι των εθνικών αρχών για την εθνική διακήρυξη διαχείριση ε, που πίεσε λοιπόν να εξασφαλιστεί αυτό το, αυτή η υποχρέωση για τα κράτη-μέλη να δηλώνουν τι ακριβώς έχουν κάνει. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω κύριε Άντορ, κύριε Άνερ, να βοηθήσετε ώστε αυτή η διακήρυξη διαχείριση, την οποία διεκδικούμε εμείς, να συνεχίσει να υποβάλλεται από τα κράτη-μέλη και να βελτιωθεί η καταγραφή ώστε να μπορούμε και στο λογαριασμό να βλέπουμε καλά και να επαληθεύουμε τι έχει ε, δαπανηθεί. Και να σας πω γιατί. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να μπούμε σε αλλού τα χωράφια. Εσείς έχετε την ευθύνη να επαληθεύετε το ότι πράγματι καταβάλλετε, κατατίθεται μάλλον η σχετική διακήρυξη από τα κράτη-μέλη και ότι είναι πλήρης κτλ. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε αυτή τη δουλειά στη θέση σας. Εσείς έχετε το καθήκον όπως πάντα κατάξετε. Γι' αυτό σας ζητούμε και όταν υπάρχουν κάποια κράτη τα οποία ενδεχομένω έχετε και κατονομάσει ε, που δεν τηρούν αυτή την προδιαγραφή να μας πείτε τι μπορείτε να κάνετε επιπλέον. Τρίτο, οι δικέ σα εκθέσει, τρίτο τομέα προβλήματο. Εδώ έχω τι αιτήσει εκθέσει δραστηριοτήτων, annual activity reports. Είναι ενδιαφέρουσε, ενδιαφέρουσα ανάγνωση. Ειλικρινεί, ανοιχτά λένε που έχετε κάποιε επιφυλάξει, ε, που δεν έχετε καταβάλει τα ποσά, δεν έχετε αποδεσμεύσει τα ποσά και θα ήθελα αν μου επιτρέπετε κύριε Άνερ, μια είστε εδώ και το είπα και νωρίτερα για τη δική σας δήλωση, αυτή που έχετε εσείς υπογράψει ως ε, Επίτροπος. Παραθέτω λοιπόν από το δικό σας κείμενο. Επιβεβαιώνω ότι δεν τελώ εν γνώση παραλήψεως ή ασδήποτε δήλωση η οποία θα μπορούσε να αποβεί εις του οργάνου. Μέχρι εδώ καλά. Και μετά έχει το however. Πλην όμως, 38 εκ των 79 προγραμμάτων που μας απασχόλησαν δεν έδωσαν επαρκείς βεβαιώσεις νομιμότητας και κανονικότητας των υφισταμένων δράσεων στις υπηρεσίες Γενικής Διεύθυνσης. Από τα, 38, 79, από τα 79 τα 38 προγράμματα δεν δίνουν επαρκείς πληροφορίες. Αλλά μας λέτε ότι θεωρείτε αυτονόητο πως είναι όλα κανονικά και ε, άμεμπτα. Συνεχίζεται μάλιστα. Εκ των 79, ε, τα 41 προγράμματα έχουν σημαντικές ελλείψεις παρουσιάσει πριν ακόμη από την εκκίνηση των κονδυλίων. Δηλαδή, για κάποιον που ξέρει καλά αγγλικά, μας λέτε ότι τα μισά προγράμματα ε, θεωρείται ότι ήταν ε, ικανοποιητικά παρότι βλέπετε ότι υπάρχουν προβλήματα ή δεν, δεν έχετε απόδειξη ότι δεν υπάρχουν προβλήματα και τα άλλα μισά είναι προβληματικά, έχουν προβλήματα και δεν είναι πλήρη. Δηλαδή αναλαμβάνετε ευθύνη για πράγματα τα οποία δεν μπορείτε κανονικά να αναλάβετε υπό την ευθύνη σας. Να δώσετε αυτή την ε, βεβαίωση ότι καλώς εκτελέστηκαν τα προγράμματα. Αυτό λοιπόν προσωρινά μπορώ να το δεχθώ ως μέθοδο εργασία, αλλά όχι μακροπρόθεσμα. Και γι' αυτό περνάω τώρα σε αυτό το οποίο λέει το ελεγκτικό συνέδριο. Η κυρία Κάλιου Λάιτ ανέφερε τα ποσοστά. 30% των περιπτώσεων είναι αυτέ οι οποίε γνωρίζουμε ότι έχουν, ενέχουν υψηλό ποσοστό κινδύνου. Και άρα δεν θα, έπρεπε να έχουν υψηλέ πληρωμέ αυτό είναι ακριβώ το πρόβλημα. Εκεί όπου γνωρίζουμε δηλαδή προκαταβολικά ότι είναι κράτη-μέλη, ότι είναι περιφέρειε στι οποίε μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα, καταθέτουμε προκαταβολικά τα ποσά, τα διαθέτουμε και μετά μα λέτε εκ των υστέρων ότι δεν μπορείτε να υπαλληθεύσετε ότι πράγματι εκτελέστηκαν σωστά. Μα ακριβώ εκεί είναι το πρόβλημα. Με τι τεράστιε προκαταβολέ είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το οποίο εμεί ε, ε, ε, βλέπουμε ω μεγάλη δυσκολία από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό που μα ενοχλεί πιο πολύ από όλα και αυτή είναι και η μόνη δυνατότητα που έχουμε ω Κοινοβούλιο να ελέγξουμε την κατάσταση στην απαλλαγή. Ξέρουμε πολύ καλά πώ να το χειριστούμε το πράγμα. Εσεί επίση γνωρίζετε τι εννοώ. Νομικά είναι δύσκολο, αλλά πολιτικά είναι πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο αυτό τη απαλλαγή. Και βλέπω ότι για το 2009 έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου η δημοσίευση των ονομάτων των κρατών μελών, όπου και έτσι με τη νέα συνθήκη τη Λισαβόνα έχουμε μια διαφορετική νομική βάση, έχουμε μια νέα νομική βάση. Έχει φτάσει πια το χρονικό σημείο να σα πούμε ξεκάθαρα ότι βλέπουμε μεγάλο πρόβλημα. Παρά τις θετικές τάσει που αναφέρατε, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να δεχθούμε προκαταβολές ποσών σε κράτη-μέλη στα οποία δεν έπρεπε να έχουν διατεθεί τα ποσά αυτά. Γιατί άλλο είναι τα ποσά του κυρίου Άντορ και του κυρίου Χάν κύριος Άντορ μιλάει για με το μέσον, έχει, έχει χρησιμοποιήσει μάλλον το μέσον της διακοπής των πληρωμών, είναι ξεκάθαρο ότι έχει χρησιμοποιήσει το μέσο αυτόν. Βεβαίω έχουμε να κάνουμε μικρότερο αριθμό προγραμμάτων ή σχεδίων καλύτερα. Αλλά πάντως πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό και αποφασιστική σημασία μέσο το οποίο πιστεύω, πιστεύω και εσείς να χρησιμοποιήσετε, διακοπή των πληρωμών. Για δε τη Λισαβόνα και την ε, έκθεση αξιολόγηση. Κύριε Καλουλάιτε, φαντάζομαι θα το επαληθεύσετε και εσείς αυτό, θα το επιβεβαιώσετε και εσείς. Εδώ δεν κοιτάμε μόνο την νομιμο, μάλλον την τήρηση των κανόνων ως προς τις πληρωμές, αυτό το κοιτάει το ελεγκτικό συνέδριο. Εμείς κοιτάμε με βάση και τη Λισαβόνα την αποτελεσματικότητα, την αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων, όχι τον τρόπο διάθεσης τους. Και γι' αυτό, μια και μιλούμε για μεγάλη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που έχει πλήξει πολλά μεγάλα κράτη-μέλη, μιλάμε για πολύ δύσκολα οικονομικά ε, δημοσιονομικά. Μιλούμε για δύσκολε διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο για τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό που έχουν βρεθεί σε μεγάλο αδιέξοδο και που δεν ξέρουμε αν θα βγουν από το αδιέξοδο. Μπορεί να καταλήξουμε να μην έχουμε προπολογισμό για του χρόνου. Έχουμε λοιπόν τώρα την υποχρέωση να δούμε πώ μπορούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα τη διάθεση των κονδύλιων μα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο ε, αυστηρή στους ελέγχους του τρόπου με τον οποίο ε, ε, εκτελέστηκαν αυτά τα σχέδια. Παρακαλώ λοιπόν αυτές τις εκθέσεις αξιολόγηση να μας πείτε πώς σκοπεύετε να τις αξιολογήσετε στη συνέχεια, πώς μπορείτε να μας ενημερώνετε για τις εκθέσεις αξιολόγησης. Γιατί πέραν τη εκθέσεως δραστηριότητας που δείχνει απλώ το τι δράσεις έχετε αναλάβει σε κάθε πρόγραμμα που έχετε, σε κάθε σχέδιο που έχετε προγραμματίσει. Θα ήθελα να μας πείτε και τι έχετε πράγματι εκτελέσει, ποιε δράσεις εκτελέστηκαν και μια πολιτική αξιολόγηση, τι όφελο έφεραν αυτές οι δράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να είναι κάποια συγκεκριμένα περιφερειακά προγράμματα, μπορεί να είναι κάποια εθνικά προγράμματα, δεν ξέρω. πάντως θέλω να έχω μια συγκεκριμένη και αποδεδειγμένη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα αυτών των σχεδίων. Αυτό θα ήθελα να βλέπω με τι εκθέσει σα. Και επίση, κύριε Άνες, χαίρομαι ιδιαίτερω που έχετε υπογράψει εδώ το κείμενο. Αν και θα ήθελα να έχω και την υπογραφή του κυρίου Χάν πάνω στο κείμενο αυτό. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να επιτρέψουμε την πρακτική η οποία σημαίνει πως απαλλάσσεται το συλλογικό όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ηγεσία αν θέλετε συγκεκριμένα, από την πολιτική ευθύνη. Όταν έχουμε την υποχρέωση για τους επιτρόπους να περνούν από ακρόαση για να εκλεγούν από το Κοινοβούλιο, πρέπει να αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη για τα όσα καταγράφουν στις ε, εκθέσεις τους και για την δραστηριότητα των υπηρεσιών τους. Ιδιαίτερα στην έκθεση αξιολόγησης θα ήθελα να δω τους επιτρόπους να αναλαμβάνουν την ευθύνη και τον κύριο Επίτροπο Χάν να τον δω να αναλαμβάνει γραπτός την ευθύνη, με την υπογραφή του δηλαδή. Σε αυτό επιμένω. Γιατί έτσι νομίζω θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό το σύστημα, εάν φέρει ο Επίτροπος κάθε φορά την ευθύνη. Και τώρα μου επιτρέπετε να, φτά, να περάσω στο 7,7 δις ευρώ που θα έπρεπε να έχουν αποδοθεί, εκ των οποίων μόνο τα 709 επιστράφησαν. 709 εκατομμύρια από 7,7 δί. Είναι αυτό που λέμε μηχανισμό διορθώσεως, διορθωτικό μηχανισμό. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν τα μέσα εκείνα τα οποία υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη, εάν έχουν ε, εισπράξει αδικαιολόγητα κάποια ποσά, να τα επιστρέφουν το χέτερο δυνατό. Θα ακούσουμε φυσικά και τι στάση του, Ευρωπα... του Λεκτικού Συνεδρίου, αλλά θα θέλαμε να ξέρουμε τι ιδέε μπορούν να υπάρχουν για την επιστροφή αυτών των ε, ποσών. Βεβαίω είναι πολύ περίπλοκη η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων, για την εκτέλεση των σχεδίων. Είναι περίπλοκη, είναι μεγάλη η γραφειοκρατία. Και βεβαίω ξέρω ότι η πρώτη απάντηση είναι η απλούστευση. Απλούστευση την οποία γνωρίζουμε ότι εσκεμμένα ορισμένα κράτη παρεμποδίζουν, μποϊκοτάρουν, γιατί βέβαια πίσω από ένα περίπλοκο σύστημα μπορεί να κρυφτεί κανεί ένα περίπλοκο σύστημα επιτρέπει την διάπραξη κάποιων σφαλμάτων τα οποία δεν εντοπίζονται εύκολα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και κάποιε συγκεκριμένε νοοτροπίε στην Ευρώπη σχετικά με αυτό. Ε, αλλά δεν είναι απαραδεκτή μια τέτοια κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να συνεχιστεί και να διονυστεί ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο σημαίνει ότι χάνονται λεφτά του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Τι έχετε λοιπόν να μα πείτε, τι έχετε συγκεκριμένα να μα προτείνετε για την εκτέλεση των προγραμμάτων Δυστυχώς η κατάσταση είναι αυτή ε, που καθιστά εσάς, ολόκληρη την Επιτροπή δηλαδή, μαζί με τα κράτη-μέλη συνυπεύθυνους για την εκτέλεση, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε 27 εκθέσεις, 27 σημεία μάλλον εκθέσεις εκτελέσεως, με αποτέλεσμα να μην είναι κανείς πραγματικά υπεύθυνο. Άρα θα θέλαμε μια πραγματική πρόταση, ουσιαστική πρόταση για το πώς θα σταματήσει αυτό το πρόβλημα. Καλό είναι να γνωρίζουμε ποια είναι τα κράτη τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη στην υπόθεση αυτή και ίσως θα είναι καλό η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία για την οποία πάντα μιλάμε να προβληθεί περισσότερο με τα προγράμματά μας και στην υπόθεση αυτή. Κυρίε και κύριοι, έχουν καταθέσει γραπτώ ερωτήσει οι συνάδελφοι. Ε, Ασφαλώ υπάρχουν και άλλε που ήθελαν και προφορικά να ε, υποβάλουν. Θέλω μόνο να σα προειδοποιήσω για το εξή. Είναι πολύ εξειδικευμένε οι ερωτήσει. σω θα ήταν σκόπιμο να δοθούν γραπτέ απαντήσει. Έτσι θα μα βοηθήσετε περισσότερο. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πια όπου η διαδικασία, η γραπτή, είναι πιο ενδιαφέρουσα. Δεν μπορούμε όμως να περιοριστούμε μόνο σε αυτό. Με 16ο έτος με αρνητική δήλωση αξιοπιστίας δεν επιτρέπεται. Γι' αυτό καλύτερα θα ήταν να συστήσουμε όχι επιμέρους και συγκεκριμένα μικρό αλλά πώς πρέπει να αλλάξουμε το πρόγραμμα. Ξέρω ότι έχετε κάνει πολλή δουλειά, κύριε Χάν, κύριε Άντορ. Ε, έχετε εξαιρετικό όραμα για την υπόθεση αυτή. Ήρθε η ώρα νομίζω να συζητήσουμε συγκεκριμένα πώ μπορούμε να αλλάξουμε το σύστημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πριν να ανοίξω τη συζήτηση θα δώσω το λόγο έστω για πολύ λίγο στους επιτρόπους έτσι ώστε ε, να απαντήσουν στον εισηγητή. Παρακαλώ πολύ κύριε Χάν. Ναι πρόεδρε ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαστε δυνατόν πιο σύντομο. Καταρχάς ευχαριστώ ρητά για την αναγνώριση της προσπάθειάς μας. Προσπαθούμε πράγματι να βελτιώσουμε εδώ την κατάσταση. Αυτό ήθελα να το επισημάνω και επί τη ευκαιρία, αν μου επιτρέπετε, να ευχαριστήσω όλο μας το προσωπικό που κατά κάποιο τρόπο έχω κληρονομήσει από την προηγούμενη Επιτροπή και που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην υπόθεση αυτή. Κύριε Χατζημαρκάκη, είναι ε, πολύ σωστή η επισήμανση ότι πρέπει να συζητήσουμε ε, επί της ουσίας, επί της βάσης μάλλον ε, της ε, πολιτικής συνοχής. Πέραν δηλαδή των στόχων, επένδυση στις περιφέρειες, προαγωγή των περιφερειών, αντιμετώπιση των οικονομικών δυσχεριών τους. Πρέπει να μιλήσουμε εδώ για ένα σύστημα το οποίο θα μας επιτρέπει στον έλεγχο, στο δημοσιονομικό έλεγχο, να έχουμε μέσα στη θέσή μας ε, στα κράτη-μέλη, στις περιφέρειες, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα φέρουν όλους αυτούς τους παράγοντες, επιχειρήσεις, περιφέρειες, κράτη-μέλη σε μια σε ένα κοινό ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι ώστε να είναι εξίσου καλός ο έλεγχος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπάρχει σχετική νοοτροπία, η κουλτούρα όπως τα λέγαμε, του δημοσιονομικού ελέγχου. Και αυτό νομίζω μπορεί να αποτελέσει μια επιπλέον συμβολή στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Οι επιχειρήσεις από τα κράτη-μέλη από τα διαφορετικά κράτη-μέλη θα γνωρίζουν ότι μπορούν να κινούνται σε ίδιο επίπεδο, στο ίδιο μήκο κύματο, με αντίστοιχε επιχειρήσει των άλλων κρατών μελών. Και έτσι έχουμε νομίζω και παιδαγωγικό καθήκον να επιτελέσουμε, διδακτικό καθήκον. Αυτό το εντοπίζω και εγώ ως καθήκον των υπηρεσιών μου, δηλαδή πρέπει να δείξουμε στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες τον δρόμο και δεν θεωρώ ότι είμαι πιο επιτυχημένος άμα επιβάλλω πολλές κυρώσει. Θεωρώ ότι είμαι πιο επιτυχημένος εάν στοχευμένα εξασφαλίζω καλά αποτελέσματα, ορθές επενδύσεις, καλύτερη παραγωγή αποτελέσματος. Και αυτή είναι η φιλοσοφία την οποία εγώ ακολουθώ και γι' αυτό σας παρακαλώ να αντιληφθείτε βάσει αυτής της φιλοσοφίας την ιδέα της δημοσιονομικής ε, διορθώσεως και της επιστροφής των χρημάτων. Η δημοσιονομική διόρθωση σημαίνει ορθή χρήση των κονδυλίων. Εφόσον αυτή εξασφαλίζεται, εφόσον τα κράτη-μέλη καταφέρνουν να προβαίνουν μόνα τους στη διόρθωση αυτή, τότε φρονούμε εμείς, και αυτή είναι η πρακτική που ακολουθήσαμε μέχρι τώρα και εγώ εμένω σε αυτήν γιατί θεωρώ ευφυή πρακτική, θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να έχουν το περιθώριο τα κράτη-μέλη ποσά τα οποία αρχικά δεν διατέθηκαν ορθά να τα εντάξουν σωστά μέσα στο δεδομένο πρόγραμμα για κάποιο άλλο σχέδιο και να τα αξιοποιήσουν με τρόπο νομότυπο. Δηλαδή, έχω αφενός μεν την ανάγκη για διόρθωση, ναι, αφετέρου δε έχω μια ενδεχομένως συγκριτικά ε, μικρότερης αξίας ανάγκη να καταβληθεί κάπου αλλού ένα ποσό δηλαδή, αλλά θα ήθελα να δίνω τη δυνατότητα στο κράτος μέλος να χρησιμοποιεί κάπου αλλού τα κονδύλια αυτά. Ε, η άλλη περίπτωση είναι να σταματήσει η διάθεση των ποσών σε, ε, εάν στο τέλος μιας περίοδου πια δεν υπάρχει η περίπτωση να αξιοποιηθούν τα κονδύλια αυτά. Γιατί λίγη η, περίοδος, η προγραμματική περίοδο και άρα δεν μπορούν να απορροφηθούν τα ποσά, οπότε και σταματάμε την πληρωμή. Δεν τα διαθέτουμε. Αυτή λοιπόν, ε, αυτές είναι οι, διπλές, οι δύο επιλογές. Αυτό λοιπόν είναι η επιλογή που έχουμε να κάνουμε και εδώ πρέπει να δούμε και κάτι άλλο, ότι έχουμε να κάνουμε συστημικά σφάλματα αφενός ή με ατομικά σφάλματα αφετέρου. Συστημικό σφάλμα είναι το να δούμε ότι ένα κράτος μέλος ε, εσφαλμένα μετατρέπει, μεταφέρει σε εθνικό δίκαιο τις διατάξεις του κανονισμού και ποια είναι υποχρεωμένο να τηρεί τις σχετικές εθνικές διατάξεις. Εκεί λοιπόν πρέπει να εντοπιστούν τα σφάλματα, σε συνεργασία με το κράτος μέλος να γίνει η διαπραγμάτευση για την σχετική διόρθωση, να μιλήσουμε για ένα ποσοστό διόρθωσης, για σχέδια τα οποία έχουν υπαχθεί σε αυτό το εσφαλμένο σύστημα, σε αυτήν την εσφαλμένη συστηματική προσέγγιση και μετά να εντοπιστούν τα συγκεκριμένα σχέδια για το κράτος μέλος, για τα οποία θα στήθει η απόδοση των κονδυλίων. Εδώ, όπω είπα, μιλούμε για διαπραγματεύσει. Επικοινωνούμε με διαπραγματεύσει. Γιατί, όπω θα φαντάζεστε, δεν έρχονται με μεγάλο ενθουσιασμό τα κράτη-μέλη να επιστρέψουν τα κονδύλια στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Μερικές φορές υπάρχουν καθυστερήσεις, μερικές φορές υπάρχει ακόμη και άρνηση να επιστραφούν τα χρήματα ή μερικέ φορέ υπάρχει απόκληση μεταξύ του ποσού το οποίο ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του υλικού στο οποίο καταλήγουμε με τη διόρθωση. Αυτό βλέπουμε, όπω είπα, στα συστημικά σφάλματα. Όταν έχουμε να κάνουμε με ατομικά σφάλματα, φυσικά και μπορούμε να δράσουμε πολύ πιο γρήγορα, όπω άλλωστε πράττουμε. Και θα παρακαλέσω και τον Γενικό κύριο Άνερ να σας δώσει περισσότερες ε, πληροφορίες για την επικύρωση κατά βάση για το πώς ε, χειριζόμαστε εμείς από πλευράς μας το θέμα αυτό. Ήταν, μια, ήταν αυτό ένα κομμάτι της μεταρρύθμισης του ΚΙΝΟΚ, ε, της μεταρρύθμισης δηλαδή του δημόσιου τομέα στην Επιτροπή. την ευθύνη την αναλαμβάνει η υπηρεσία, το προσωπικό της υπηρεσίας πολύ πιο σαφώς με την υπογραφή των σχετικών υπαλλήλων, των αρμοδίων υπαλλήλων. Η πολιτική ευθύνη ούτω ή άλλω ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συλλογικά. Συλλογικά έχει λάβει τι αποφάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συλλογικά έχει την πολιτική ευθύνη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και έτσι υποβάλλεται η έκθεση στην, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει η ευθύνη τη Υπηρεσία, όπω είπα, και ούτω ή άλλω η αλλω η ευθύνη της Επιτροπής. Για την απλούστευση, κύριε Πρόεδρε, θα έχουμε πιστεύω την ευκαιρία να συζητήσουμε περισσότερο. Χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες, ναι, αλλά θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να υπενθυμίσω ότι μέρος του γραφειοκρατικού φόρτου προκύπτει μέσα στο κράτος μέλος. Και βέβαια συνομιλούμε με τα κράτη-μέλη και τους ζητούμε να μειώσουν αυτό το γραφειοκρατικό φόρτο. του τα ρωτάμε εσεί τι μπορείτε να κάνετε από πλευρά σα για να μειωθεί ο γραφειοκρατικό φόρτο. Διαπιστώνω λοιπόν εγώ σε σχέση με κάποιο συγκεκριμένο κράτο μέλο ότι η, από την αίτηση, την κατάθεση τη αίτηση μέχρι την ε, οριστική ε, καταβολή των ποσών περνάνε 8 μήνε ενώ το κράτο μέλο είναι κράτο μέλο μόλι 6 μήνε. Ε, στο κράτο μέλο, μάλλον μένει η διαδικασία επί 6 μήνε. Στι Βρυξέλλε μόνο 2, αλλά ακούγεται στον τύπο ότι α, μια διαδικασία κρατάει στι Βρυξέλλε 8 μήνε, γιατί οι Βρυξέλλε έχουν μεγάλη γραφειοκρατία κτλ. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν ορισμένα πράγματα σε σχέση με το σύστημα και με το ποιο, πού εντοπίζονται οι ευθύνε ή η γραφειοκρατία. Αν μου επιτρέπει τώρα ο Γενικός Διευθυντής κ. Άνερ να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ το πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με τη δική μου έκθεση δραστηριοτήτων που περιγράψατε ως προς το έτος 2009 ήταν ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, ειδικότερα όσον αφορούσε τα 38 προγράμματα εκ των 79 που αναφέρατε. 38 προγράμματα για τα οποία δεν είχα καμία ασφάλεια, καμία πρόβλημα λοιπόν. Ήταν ότι ορισμένα κράτη-μέλη, μια σειρά κρατών μελών και περιφερειών δεν ήταν έτοιμα εγκαίρως ή ετοίμασαν πολύ καθυστερημένα την επαλήθευση ε, συμμόρφωσης. Και έτσι την δεχθήκαμε, με μεγάλη καθυστέρηση. Ωστόσο τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες πολύ συχνά για τον λόγο ακριβώς αυτών ε, διέθεσαν πολύ περιορισμένα κονδύλια και αντίστοιχα οι ελεκτικές τους αρχές πραγματοποίησαν πολύ λίγους περιορισμένους ελέγχους. Αυτό σχετίζεται τα προηγούμενα χρόνια με αυτό το οποίο αναφέρατε και εσείς, δηλαδή μετάβαση σε, ένα, ε, σε μια αλλαγή συστήματος, σε ένα διαφορετικό σύστημα. Αυτό έχουμε πραγματοποιήσει, έχουμε περάσει ένα διαφορετικό σύστημα και όπως είπα δεν είχα ασφαλίσει πληροφορίες, δεν είχα βεβαιότητα πώς τα ποσά για τα κράτη-μέλη ευσταθούν. Μάλιστα ένα από αυτά τα κράτη ε, προσήχθη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και είμαστε αναμονή της δημιουργίας. Αυτή η κατάσταση όμως δεν θα επαναληφθεί τα επόμενα χρόνια. Δεν προβλέπεται να επαναληφθεί. Κυρίες και κύριοι, λέει ο κύριο Άντερ, καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζημαρκάκη για την ανάλυση της κατάστασης. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η αξιολόγηση του και η ταυτοποίηση των βασικών προκλήσεων ε, του κυρίου Χατζημαρχάκη συνάδει με τις δικές μας απόψεις, ειδικότερα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής. Ο, ως προς το θέμα της ε, ετήσιας έκθεσης ε, και για τις δραστηριότητες, συμφωνώ με τον κύριο Χάν. Ακολουθούμε τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Γενική Διεύθυνση για τη Συνοχή ακολουθεί ε, την πεπατημένη που ακολουθούν και οι άλλες γενικές διευθύνσει. Επιτρέψτε μου τώρα να εστιάσω την προσοχή μου σε κάποια βασικά ζητήματα που έχουν τεθεί από τον εισηγητή. Οι διακοπέ και οι παύσει, Αλλά και τα καθήκοντα που θα πρέπει να φέρουμε σε πέρα στην επόμενη περίοδο. Δηλαδή, την απλούστευση. Και ίσω επεκταθώ και λίγο περαιτέρω. Τώρα, ω προ τη διακοπή και την παύση. Ε, θα ήθελα να τονίσω το εξή. Είναι μεγάλη διαφορά. Είναι ουσιαστική διαφορά ε, μεταξύ της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου και της προηγούμενης. Ε, θεωρούμε ότι έχει βελτιωθεί η ποιότητα. Δεν είναι όμως αυτοσκοπός αυτό. Είναι ένα εργαλείο, μια δυνατότητα που έχουμε για να βελτιώσουμε ε, τη διαχείριση, να κάνουμε πιο ποιοτική διοίκηση, αν θέλετε, της κατάστασης και σε δικό μας επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών. Πρέπει όμως να αξιοποιήσουμε αυτό το εργαλείο με επικοδομητικό τρόπο για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις των κρατών μελών και ποσοτικά και ποιοτικά, για να αξιοποιήσουν καλύτερα τα κράτη-μέλη τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν είναι κάτι που γίνεται αυτόματα, αλλά δεν είναι και κάτι που εξαρτάται αμυγός από μια πολιτική απόφαση. Είναι μια διοικητική, διαχειριστική απόφαση. Είναι προϊόν συνεχούς επαφής και επικοινωνίας μεταξύ γενικών διευθύνσεων από τη μία και χρηστών κονδυλίων από την άλλη. Είναι μια δυνατότητα να εντοπίσουμε σφάλματα, λάθη, τη στιγμή που αξιοποιούνται τα κονδύλια όταν εκταμιεύονται ή στη συνέχεια. Σφάλματα και λάθη που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή των διαφόρων προγραμμάτων. Προσπάθησα να σε εξηγήσω το πνεύμα αυτής της πρακτικής. Αυτό είναι το πνεύμα ε, πίσω από αυτή την δράση και ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσει να προσφέρουμε καλά αποτελέσματα. Επίσης είναι αληθές ότι η περαιτέρω απλούστευση αναπόφευκτα και κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγήσει σε μικρότερη πιθανότητα διάπραξης σφαλμάτων. Θα κάνουμε το παν, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να εντοπίσουμε τα βήματα που θα πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια για να προβούμε σε περαιτέρω απλούστευση, για να εισαγάγουμε πιο απλούς κανόνες ως προς την επιλεξιμότητα, για παράδειγμα. Μετά την, το 2013, στο τέλος δηλαδή αυτής της προγραμματικής περίοδου. Νομίζω ότι ε, η πιο ρεαλιστική προθεσμία είναι αυτή. Ότι δηλαδή ε, ουσιαστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορέσουν να γίνουν την επόμενη προγραμματική περίοδο. Δεν ε, ασχολούμαστε όμως μόνο με αυτό. Εξίσου σαφές είναι ότι πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας ως προς τις διαφόρων ειδών αξιολογήσεις για να δείξουμε ότι σωστά χρησιμοποιούνται τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου, ότι αξιοποιείται ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός προς όφελος του Ευρωπαίου πολίτη και ότι ε, αυτό συνεπάγεται προστιθέμενη αξία για τον Ευρωπαίο πολίτη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για να το αποδείξουμε αυτό θα πρέπει να έχουμε κάπως διαφορετικά συστήματα αξιολόγησης, να βασίζονται δηλαδή περισσότερο στις επιδόσεις, στην απόδοση. Και είναι κάτι το οποίο ε, θα πρέπει να γίνει. Έχουμε χρόνο μπροστά μας και χρησιμοποιούμε και τη συνεισφορά που έχουμε αποκομίσει μετά από τη διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη, μεταξύ των οποίων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γκρέσλερ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι απολύτως ε, σίγουρη για το τι θα κάνουμε με αυτή την έκθεση της, ε, του Ελληνικού Συνεδρίου για το 2009 ε, γιατί στα διαχρονικά προγράμματα για 50% των περιπτώσεων, εάν καταλαβαίνω καλά, δεν υπήρξαν πληρωμές. Επίσης, στο κοινωνικό ταμείο δεν υπήρξαν πληρωμές για σημαντικά μέρη του προγράμματος. Έχουμε λοιπόν απέναντί μας μια ιδιάζουσα κατάσταση ε, μαζικές αρνήσεις πληρωμών. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν να δουλεύουμε πάνω σε αριθμούς οι οποίοι δεν είναι αποκαλυπτικοί. Θα ήθελα επίσης να μάθω Ε, ε, τι υπόλοιπα υπάρχουν για το 2009. Ε, προφανώς υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες δεν έχουν διαχειριστεί τα προγράμματα ως όφυλαν. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που τα πράγματα πήγαν καλά, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι πρέπει να αναρωτηθούμε τι θα κάνει η Επιτροπή πέρα από τα ωραία λόγια και σε περιπτώσεις αμφιβολίας τι κάνει ε, θα ήθελα λοιπόν λίγο να σκέψουμε πάνω σε αυτό το ε, ζήτημα. Επίσης, ε, σχετικά με τις απαντήσεις, γραπτές απαντήσεις ερωτήσεις μας να πω ότι επανειλημμένα έγινε λόγος στον κανονισμό και στην ουσία δηλαδή λείπει η βάση για, για τις απαντήσεις που μας δόθηκαν. Ας πούμε 30% ή 70% μάλλον αυτών των ερωτήσεων ε, θα έπρεπε να είχαν απαντηθεί ήδη από το ελεγκτικό συνέδριο ε, σχετικά με τους εκ των προτέρων ελέγχους. Φαίνεται ότι βάσει των εξάντε ελέγχων 70% των λαθών δεν είχαν ανοιχνευτεί. Επομένως θα πρέπει το σύστημα ελέγχου να είναι αποτελεσματικό. Τη στιγμή του πρώτου ελέγχου θα πρέπει να μπορεί να διαπιστώνεται το σφάλμα. Επίσης, Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλη η διαφάνεια ε, του, της ε, διαδικασίας ε, επιστροφής. Από όσα κατάλαβα από τον κύριο Χάν, δεν γνωρίζει ακριβώς το ποσό των επιστροφών, τι επιστράφει ή τι όφιλε να επιστραφεί. Δεν είναι σαφές λοιπόν. Επομένως, θέλω να μας πείτε ποιες είναι οι προτάσεις σας, μάλλον τι προτίθεστε να κάνετε, έτσι ώστε να βελτιώσετε συγκεκριμένα όλα αυτά τα οποία σας αναφέρω. Όσον αφορά και τον κύριο Αντόρ, την προηγούμενη εβδομάδα περάσαμε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ε, για, μιλώντας για διάφορα ζητήματα οικονομικού ενδιαφέροντος. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται Ville Social, κοινωνικές πόλεις. Δέκα μικρο projects υπάρχουν. 15.000 ε, διοικητικά έξοδα οι επικεφαλείς ε, των ε, ε, προγραμμάτων πρέπει να, κάνουν, πρέπει να πληροφορούν το Βερολίνο, καθώς επίσης να δίνουν και συνεντεύξεις τύπου και μετά έχουμε διόρθωση, εδώ βλέπουμε διόρθωση των, των αναφορών τους. Το πρόβλημα γερμανογερμανικό, Λοιπόν, εδώ ή υπάρχει κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ, Χαν και Άντορ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκρέσλε, το πρώτο ερώτημά σας ε, αφορούσε στην ε, ικανότητα των ε, της αξιοποίησης των πόρων, έτσι δεν είναι. Δύο είναι οι παρατηρήσεις που θα πρέπει να έχουμε όλοι υπόψη μας. Καταρχάς, όντως σημειώνεται καθυστέρηση, ελαφρά καθυστέρηση και αυτή η καθυστέρηση οφείλεται σε δύο λόγους. Για την περίοδο μέχρι και το 2006 είχαμε παράταση των διαφόρων προγραμμάτων και σχεδίων πιο μακροχρόνια. Και τα κράτη-μέλη είχαν εστιάσει την προσοχή τους στην πλήρη αξιοποίηση των υφιστάμενων προϋπολογισμών, των υφιστάμενων κονδυλίων. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο ε, λόγο, λόγο όλων αυτών των προγραμμάτων relance και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολλοί έλεγαν, έχω ένα πρόγραμμα που μπορεί να είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση σε στοχή πλαίσιο ή μπορεί να χρηματοδοτηθεί με περιφερειακά κονδύλια. Και στο τέλος λέει όχι, προτιμούμε προγράμματα οικονομικής αναζωπήρωσης γιατί ε, είναι διαθέσιμα πιο σύντομα για δύο χρόνια. Ενώ τα κονδύλια τα περιφερειακά ε, εκτείνονται, σε 7 χρόνια, σε μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Είναι δηλαδή δύο ψυχολογικοί παράγοντες που ε, προέκυψαν και σε αυτούς οφείλεται η ελαφρά καθυστέρηση και είμαι πεπισμένος 100% ότι θα ε, ανακάμψουμε και θα καλύψουμε αυτή την καθυστέρηση μέχρι και το τέλος της προγραμματικής περίοδου. Πέρσι είχαμε πολύ πιο, συγκεκριμένη, ε, πολύ πιο συγκεκριμένο σχεδιασμό γιατί ε, είχαμε αξιοποιήσει το 100% του υφιστάμενου προϋπολογισμού. Σήμερα γνωρίζουμε σε βάθος την κατάσταση και γνωρίζουμε πότε μπορούμε να κινητοποιήσουμε κονδύλια και για ποιο λόγο. Τώρα, ως προς την ποιότητα των ελέγχων. Αυτό το οποίο, αν θέλετε, ε, διακυβεύεται είναι το ότι τα προγράμματα εκτείνονται σε πολλά και διαφορετικά έτη. Ορισμένοι έλεγχοι εξάντε εκ των προτέρων για διάφορους λόγους. Γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί ε, τα προγράμματα αυτά. Πολλές φορές οι έλεγχοι εξάντε εκ των προτέρων δεν μας οδηγούν στην ανείχνευση και ταυτοποίηση σφαλμάτων ή ανακριβιών. Ε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι με την ετήσια επαλήθευση του ελεγκτικού συνεδρίου Ε, γίνεται έλεγχος σε ένα πρώτο επίπεδο. Έχουμε τρία επίπεδα ελέγχου και επαντλήθευσεων. Και γι' αυτό έχω πει επανειλημμένος ότι ελπίζω ότι κάποια μέρα θα καταλήξουμε σε μια αποδεκτή διαδικασία μετά το οριστικό κλείσιμο της προγραμματικής περίοδου θα πρέπει να γίνεται μια επαλήθευση του συνόλου της περίοδου από το ελεκτικό συνέδριο και να διαπιστώνεται το ποσοστό των σφαλμάτων και θα πρέπει αυτά τα νούμερα να χρησιμεύσουν ως σημεία αναφοράς για την ετήσια αξιολόγηση και τους ετήσιους ελέγχους. Θεωρώ ότι για να είναι αποτελεσματικό το σύστημα αυτό θα πρέπει όλα αυτά να προβλεφθούν. Ε, θα ήταν καλό να υιοθετήσουμε κάτι τέτοιο. Θεωρώ επίσης ότι από την επόμενη χρονιά τα κονδύλια θα συμνοδεύονται από ένα ενιαίο έντυπο, αν θέλετε, ένα σύστημα έκθεσης από πλευράς κρατών μελών. Αυτό θα μας επιτρέψει να μάθουμε καλύτερα τα ποσοστά σφαλμάτων ανάλογα με το είδος του προγράμματος, ανάλογα με την περιφέρεια ή ανάλογα με τη χώρα. Θα χρειαστεί ένα-δύο χρόνια ε, μέχρι να καταλήξουμε σε ένα ικανοποιητικό ε, ποιοτικό και ποσοτικό σύστημα αξιοπιστίας ε, της αξιολόγησης. Δεν μπορούν όλες αυτές οι χώρες μέσα σε μια βραδιά να λειτουργήσουν με τον ίδιο τρόπο. Θα πρέπει να, χρησι... να περάσει κάποιο χρόνος μέχρι ότου να συμμορφωθούν και να ανέβει η ποιότητα τη δουλειά. Πρόεδρο. Ε, η κυρία Γκρέσλερ σας έκανε και μια συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με αυτή την υπόθεση του Βερολίνου. Τι μπορείτε να μας απαντήσετε γι' αυτό. Δεν έχουμε Κυρία ε, Γκρέσλε, δεν έχουμε φέρει υλικό τεκμηρίωσης για συγκεκριμένο πρόγραμμα εξατομικευμένο. Εάν θέλετε να επανέλθουμε γραπτός και να σας δώσουμε αυτές τις πληροφορίες αργότερα. Αλλά για τη σημερινή συνεδρίαση δεν έχουμε μαζί μας αυτά τα στοιχεία. Κύριε Επίτροπε, δεν ήθελα να σας ε, φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά δεν υπάρχει κάπου κάποια διάταξη η οποία λέει θα πρέπει να επαληθεύονται από την ε, ιεραρχικά προϊσταμένη αρχή ή ανακοινώσει τύπου. Κάποιος τέτοιος όρος δεν υπάρχει κάπου. Well, uh, Κοιτάξτε, είναι πολλά τα στοιχεία τα οποία είναι δημόσιου χαρακτήρα για τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της συνοχής και για προγράμματα ξεχωριστά. Δεν είναι ε, ένα θέμα για το οποίο είναι δύσκολο κανείς να αποκτήσει πληροφορίες. Εύκολα μπορεί κανείς να αξιολογήσει την κατάσταση έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Βόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ε, έκθεσή Έχω μία ερώτηση για τον Επίτροπο της ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης, ο οποίος κάνει πολύ καλή δουλειά. Νομίζω ότι η μείωση του ποσοστού σφάλματος ε, σε αυτό το θέμα από το 11% στο 5% δείχνει την πολύ καλή πρόοδο που έχει σημειωθεί. Ωστόσο, θα ήθελα να σας επεσημάνω το εξής. Ένα παράδειγμα όπου σφάλματα ίσως σημειώθηκαν εσκεμένα ε, για την ε, εταιρεία Twinings ε, τσαγιού, η οποία είχε ε, δύο εργαστάσεων στον Αμένο Βασίλειο. Μετά είχαμε μείωση θέσεων απασχόλησης, ε, σύστησε μια θηγατρική, έφτιαξε ένα καινούριο εργοστάσιο στην Πολωνία, η οποία, το οποίο εργοστάσιο έλαβε χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Και ξέρετε, ένας συνάδελφος ε, απέστειλε επιστολή στον Επίτροπο και ανέφερε το περιστατικό και ο επίτροπο απάντησε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα κατά την άποψή του, διότι η Άνιξ ήταν μικρομεσαία επιχείρηση τεχνικός, άρα ήταν επιλέξιμη ε, για τα ε, διαρθρωτικά ε, ταμεία. Μπορείτε να το σχολιάσετε, δηλαδή είναι σωστή αυτή η χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων. Πολλοί συναδελφοί υπάρχουν που έχουν άλλα παραδείγματα τέτοιου είδους. Είναι ξεκάθαρη περίπτωση μετεγκατάστασης για λόγους κόστους. Ε, δεν μπορείτε να εξετάσετε τους κανόνες, να αλλάξει η νομοθεσία έτσι ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Ο Επίτροπος Χάν, παρακαλώ. Ναι, θα, θα σας πω ότι, με πάση ειλικρινία, είναι πολύ δύσκολη η υπόθεση και ερώτηση Ναι, μπορώ να δω ότι βεβαίω υπάρχει κάποια σύμπραξη εδώ στι περιπτώσει των περιφερειών, των κρατών με το Twinings. Υπάρχει πάντω σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάθε φορά περίπτωση επιχειρήσεις να μεταθέτουν το κέντρο των επιχειρήσεών τους, της παραγωγής τους και μπορώ να σκεφτώ ένα πρόχειρο παράδειγμα μιας ε, αλυσίδας ρούχων, ε, ειδών ενδύσεως, μόδας, που είχε ένα κέντρο διανομής στο Παρίσι και αποφάσισε να κατασκευάσει ένα άλλο κέντρο διανομής εδώ κοντά στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. Και ενώ κανονικά θα περίμενε κανείς ότι απειλείται το Βέλγιο από το, οι Βρυξέλλες από το Παρίσι, όχι, ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση να μετατεθεί εδώ το κέντρο αυτό διανομής στις Βρυξέλλες. Και πάλι με ευρωπαϊκά κονδύλια, με χρηματοδότηση και με ε, απώλεια στο πρώτο κέντρο των Παρισιών δηλαδή θέσεων εργασία. Αυτό μπορώ να πω μόνο ότι εν τέλει στο σύνολο έχει παραχθεί ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία συνολικά. και δεν μπορεί κανεί να ζητήσει λογαριασμό για μια τέτοια επιλογή, γιατί υπάρχουν σαφείς κανόνες οι οποίοι τα, τηρούνται. Η μετάθεση ενό κέντρου παραγωγής, διάθεση εμπορία που μπορεί να έχει χρηματοθετηθεί πριν από μερικά χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί τώρα για ένα άλλο ε, μέρος, για μια άλλη τοποθεσία να μην είναι επιλέξιμη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει η επιλογή της επιχείρησης να αναπτύξει μια νέα μονάδα, ένα νέο κέντρο στην Πολωνία. Και από ό,τι γνωρίζω, μέχρι τώρα έχουν αξιοποιηθεί κονδύλια για μικρομεσαία επιχείρηση, τάξεως μεγέθους μικρομεσαίας επιχείρησης δηλαδή, με τρόπο απόλυτα νομότυπο. Φυσικά θα ελέγξουμε εις βάθος την υπόθεση, έλεγα πάντως εδώ στο Κοινοβούλιο για την Επιτροπή σας, ότι δεν είναι δυνατόν να επιβάλλουμε μια, ένα τέτοιο περιορισμό. Υπάρχουν περιπτώσεις που μετατίθεται μια μονάδα παραγωγής μέσα στο κράτος μέλος από τη μια περιοχή στην άλλη. Γιατί μια περιοχή είναι περιοχή ε, σύγκλησης και η άλλη ανταγωνισμού. Και άρα υπάρχει περισσότερη δυνατότητα χρηματοδότησης για την περιοχή σύγκλησης και μπορεί να αξιοποιηθεί τα κονδύλια αυτά η επιχείρηση. Και από την άλλη έχουμε μακροοικονομική ε, υποχρέωση, καλύτερα μας ενδιαφέρει μακροοικονομικά να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη αυτής της περιοχής σύγκλησης και στην προσέγγιση τέτοιου είδους επιχειρήσεων ή ε, θέσεων εργασίας. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να πω το εξή για να μην βλέπουμε τα πράγματα μόνο από πλευράς από τη σκοπιά μάλλον της εκλογικής περιφέρειας ότι βρισκόμαστε μέσα σε έναν διεθνή ανταγωνισμό. Μήπως είναι προκυμότερο όταν πρόκειται να μετακομίσει μια επιχείρηση, να μετακομίσει μέσα στην Ευρώπη και να μην πηγαίνει να εγκατασταθεί στην Κίνα ή την Ινδία. Γιατί τότε νομίζω είναι πολύ προβληματικές συνθήκες του ανταγωνισμού. Ως επιχειρηματίες λοιπόν, ως Ευρωπαίοι νομίζω πρέπει να δούμε και αυτή την πτυχή. Sorry, λίγο μιλείτε στα αγγλικά, αλλά δεν μπορώ να δώσω περισσότερες απαντήσεις. Δεν είναι απλή ερώτηση, είναι πολύ περίπλοκη. Υπάρχουν σαφείς κανόνες μετακίνησης μίας επιχείρησης μετά τα πέντε χρόνια, εφόσον δηλαδή πέντε χρόνια ε, έχουν εκκρέψει από τη στιγμή που καταβλήθησαν αυτά τα ποσά, τη στήριξη, μπορεί να μετακινηθεί. Βεβαίως είναι πολύ πιο περίπλοκη η όλη κατάσταση αλλά έχω δώσει εντολή στις υπηρεσίες μου όταν έχουμε να κάνουμε δύο κράτη να κοιτάμε πάντα το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, Ανδρέας. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση πρώτα απ' όλα προς την κυρία Καρολάιτ. Υπάρχει δυνατότητα να μετρηθεί ε, το κατά πόσον η μείωση του περιθώριου λάθους σχετίζεται με την μείωση του αριθμού των προγραμμάτων που λειτουργούν λόγω ελλείψεως της χρηματοδότησης. Ερώτηση προς τους Επιτρόπους, κύριε Άντορ και Χάν. Ποια είναι η αντίδρασή σας στο δημοσίευμα των Financial ε, Times όσον αφορά τα διαφορετικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής σύμφωνα με το οποίο ε, τα χρήματα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης καταλήγουν στα χέρια της Ιταλικής μαφίας. Κύριε Αντόρο, γιατί θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν την υποχρέωση δημοσίευσης λογαριασμών, ας πούμε, όπως οι τράπεζες. Και εν παρόδο, να συμφωνήσω με τα σχόλια του κυρίου Βόν, γιατί ξέρω και στην Ιρλανδία υπάρχουν εταιρείες όπως η Dell που ε, έφυγαν από την Ιρλανδία και πήγαν στην Πολωνία λόγω χαμηλής εταιρικής ε, ε, φορολογίας ε, και τελικά είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τελικά θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα του κοινωνικού ταμείου για την αποζημίωση των Ιρλανδών που θα έχουν χάσει τη δουλειά τους κυρία Καριλάιντε ευχαριστώ πολύ μείωση του περιθώριου λάθους και κατά πόσον εξαρτάται αυτή από την μείωση της χρηματοδότησης είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πούμε κανείς. Ε, παραμένει αρκετά χαμηλό το ποσό χρηματοδότησης ε, και το ποσοστό εξε, εκτέλεσης επίσης δεν είναι τόσο υψηλό όσο κάποια προηγούμενα χρόνια. Απ' την άλλη πλευρά ε, εν μέρη οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιες χώρες χρησιμοποιούν ακόμα χρήματα παλαιών περιόδων ε, δεν υπήρξαν επίσης ε, ε, πολλά παράπονα σχετικά με την μη διαθεσιμότητα των κονδυλίων από πλευράς της Κομισιόν και είναι γεγονός ότι παρόλα αυτά εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν παλιά χρήματα τα, οι χώρες, τα κράτη. Γενικώ είναι πολύ δύσκολο να ε, προχωρήσουμε στη διατύπωση και διαπίστωση κατά αυτή την έννοια και επίσης κατά την διάρκεια των επισκέψεων μας στις χώρες μέλη δεν διαπιστώσαμε να έχουν σταματήσει προγράμματα λόγω της αδυναμίας συγχρηματοδότησης. Βεβαίως, εάν κανείς δεν δαπανά χρήματα, προφανώς δεν θα κάνει και λάθη. Ε, αλλά, όπως είπα και στην αρχή, ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει κάποια κάποια επίπτωση αυτής της μείωσης των χρηματοδοτήσεων στη μείωση των ε, λαθών γιατί είναι γεγονός ότι κάποια σφάλματα που δεν έχουμε δει στην αρχή μπορεί στην ε, στον επόμενο έλεγχο να γίνουν σαφή. Κύριε Χαν, κύριε Επιτρόπε. Ναι. για το θέμα της μεταφοράς. Δεν είναι βέβαια θέμα της συζήτησης εδώ, αλλά στην Ευρώπη έχουμε να κάνουμε με πολύ διαφορετικά συστήματα οικονομικά και φορολογικά, που σημαίνουν βέβαια, που σημαίνουν βέβαια και διαφορετική ελκυστικότητα κάποιες περιοχές ή κάποιους, κάποιου κράτους. μια επιχείρηση. Ο φορολογικός παράγων, πέραν της ποιότητας των διαθέσιμων μέσων, είναι ασφαλώς πολύ σημαντικός παράγων στη λήψη απόφασης για την εγκατάσταση μιας επιχείρησης ε, σε μια περιοχή. Ναι, μπορεί να είναι λόγος η εξασφάλιση κονδυλίων, ενισχύσεων, αλλά και ένα πιο ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον μπορεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα επίσης. Επίσης, βλέπουμε ότι επικρίνεται το γεγονός ότι δεν διατίθεται αρκετά ποσά. Και από την άλλη, μια-δύο παραγράφεις πιο πέρα, βλέπουμε ότι φταίει η γραφειοκρατία, μάλλον ότι δεν γίνονται αρκετοί έλεγχοι για τη διάθεση των ποσών. Και μετά δύο παραγράφους πιο πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει επίκριση για την υπερβολική γραφειοκρατία. Ναι, αλλά πρέπει κάπω να ελέγχονται τα ποσά που διατίθενται και για να ελεγχθούν πρέπει να υπάρχει σχετική δομή που ονομάζεται γραφειοκρατία. Το πρόβλημα εντοπίζεται, όπω είπα νωρίτερα, ε, στο επίπεδο των κρατών μελών, όπου δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε απευθείας τον έμεσο, τον έλεγχο. Είμαστε υποχρεωμένοι να επαφεθούμε στις εκθέσεις των κρατών μελών. Κάνουμε στο βαθμό που μπορούμε τους ελέγχους, λαμβάνουμε τις σχετικέ επιβεβαιώσεις, επιβεβαιώνουμε δηλαδή και την ποιότητα του δημοσιονομικού ελέγχου τακτικά, ώστε να μην δίνεται μία λευκό επιταγή με την ε, επιβεβαίωση, την πιστοποίηση των δημοσιονομικών ελεγκτών ή των ελεκτικών αρχών. Όχι, δεν δίνουμε λευκό επιταγή, παρακολουθούμε διαρκώς την κατάσταση και προσπαθούμε να διεξάγουμε στο δυνατόν πιο πολλούς και πιο αποτελεσματικούς ελέγχους αλλά δεν είναι και σωστό από την άλλη να στιγματίζεται ένα συγκεκριμένο κράτος ως πάντα υπέτειο για τα προβλήματα της παρατυπίας. Ενδείξεις δηλαδή δεν έχω επιπλέον να δώσω. Η μόνη ένδειξη που μπορώ να σας δώσω στους ελέγχους μας είναι η μηδενική ανοχή. Αυτό είναι μια πάγια, μια σταθερά στην ε, στάση μας απέναντι στους προσωπικούς ελέγχους. Ευχαριστώ κύριο Σάντορ. Όσον αφορά τα δημοσιεύματα του Financial Times, βεβαίω είναι μια σημαντική εφημερίδα και επομένως ε, ε, το γεγονός ότι ασχολείται με το Ταμείο Συνοχής, τις πολιτικές συνοχής και τα διορθωτικά ταμεία είναι πολύ σημαντικό. Ε, τα διαβάζουμε άλλωστε τα δημοσιεύματα αυτά όλοι μας και είναι σημαντικό που ασχολείται η εφημερίδα. Όμως ε, πρέπει να πω ότι δεν θα συμφωνήσω με πολλές από τις ε, αναφορές ή ε, υπόνοιες ή και συμπεράσματα. Αυτό θα κάνω και στην προκείμενη περίπτωση. Και η συλλογή των στοιχείων αλλά και πολλά από τα συμπεράσματα οδηγούν σε εσφαλμένη κατεύθυνση και νομίζω ότι και διαβάζοντας προσεκτικά τα δημοσιεύματα δεν βλέπουμε ε, ο δημοσιογράφος να έχει ε, πολύ ισχυρά ε, στοιχεία. Σχετικά ε, με τα ευρωπαϊκά χρηματοοικονομικά εργαλεία σε σχέση με τα ιδιωτικά αντίστοιχα εργαλεία ή μέσα. Ε, νομίζω ότι δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε ακριβώς τις πρακτικές ιδιωτικών εταιριών γιατί σε αυτές η χρηματοδότηση και αναχρηματοδότηση ε, αναφέρεται και συνδέεται με την αξιοπιστία, με την φρεγγιότητα αλλά και την διάθεση ε, στην προκείμενη περίπτωση τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τα δημόσια οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθούν μια δική τους ε, πορεία. Η αναχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν βασίζεται και δεν εξαρτάται από ιδιωτικές ε, πηγές και επομένως δεν είναι απαραίτητη η δημοσιοποίηση, δημοσιοποίηση των τρεχόντων λογαριασμών από την άλλη πλευρά ε, το να προσπαθούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο θα ήταν ε, απόλυτα μεγάλη δαπάνη και στην ουσία κατασπατάληση του χρήματος των πολιτών γιατί δεν θα ανταποκρίνεται σε έναν ε, συγκεκριμένο σκοπό. Έχουμε ένα ορθό σύστημα, έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι αξιόπιστο, έχουμε συστήματα ελέγχων ε, και νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να κατανοήσουν οι φορολογούμενοι τι ακριβώς συμβαίνει με τα χρήματα. Ε, επίσης υπήρξε μια επιπλέον ε, ε, ερώτηση πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα του Ταμείου uh, της προσαρμογής του παγκοσμιοποίηση και πώς χρησιμοποιούνται σε σχέση με αυτές τις μετακινήσεις επιχειρήσεων. Στην προκείμενη περίπτωση της Ιρλανδίας η συγκεκριμένη εταιρεία έφυγε όντως από την Ιρλανδία και ε, αύξησε την ανεργία, δημιούργησε νέους ε, ανέρχους. Προχώρησε αρχικά σε μείωση της παραγωγής. Το παράδειγμα όμως δεν αποτελεί τυπικό παράδειγμα. Βεβαίως ε, ενδελεχώς μελετούμε την περίπτωση αυτή, την ερευνούμε για την ώρα δεν έχουμε βρει κάποιες ε, ατασταλίες ή ανομαλίες, ε, αλλά βεβαίως οι πολιτικές ευαισθησίες ε, είναι σημαντικές. Πρέπει όμως για μία ακόμα φορά να πω ότι δεν είναι αυτός ο συστηματικός τρόπος χρήσης των κονδυλίων του Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Αντιθέτως πρέπει να χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τους ε, ε, εργαζόμενους να προσαρμοστούν στις νέες καταστάσεις και σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Κοινοβουλίου πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους του Ελεκτικού Συνεδρίου για την πολύ καλή δουλειά τους, αλλά και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσίασή τους. Ζητώ συγγνώμη που δεν σας απευθύνω την ερώτηση κατά πρόσωπο και σας έχω γυρισμένη την πλάτη, αλλά έτσι είναι η διάταξη της αίθουσας. Πολλοί συνάδελφοι το είπαν, είναι πολύ θετικό και πολύ καλό το γεγονός ότι παρακολουθούμε και βλέπουμε μια την τάση να βαίνει μειούμενη ως προς τα σφάλματα και αυτό είναι προϊόν ε, της αποτελεσματικότητας των συστημάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ταυτοχρόνως όμως είναι κάπως απογοητευτικό να ε, βλέπουμε ότι συνεχίζονται τέτοιου είδου σχόλια και συμπεράσματα από το ελεγκτικό συνέδριο την τελευταία 15 ετία τα ίδια και τα ίδια. Όντως το ποσοστά σφαλμάτων έχει πέσει, έχει μειωθεί δραστικά συγκριτικά με το 11% της περσινής χρονιάς. Αυτά είναι τα καλά νέα Ωστόσο, μήπως αυτό έχει σχέση και με την δειγματοληψία, τον τρόπο ε, συλλογής των δειγμάτων από τις ε, χώρες μέλη. Και απευθύνω το ερώτημα και στους δύο επιτρόπους. Κύριε Χάν, θα ήθελα να σας ρωτήσω ε, κάτι που έχει σχέση και με τη γραπτή ερώτηση που σας έχω απευθύνει. Τα ασφάλματα που θα, θα έπρεπε μήπως να έχουν ανοιχνευθεί από τα κρατη και να διορθωθεί από τα κράτη-μέλη πώς ε, παρακολουθεί η Επιτροπή αυτού του είδους περιπτώσεις, τις περιπτώσεις δηλαδή όπου τα κράτη-μέλη εντοπίζουν σφάλματα και τα ανοιχνεύουν. Στην απάντησή σας προσφέρατε λεπτομερείς εξηγήσεις. Όμως ε, ε, είπατε κάτι, γράψατε κάτι στην απάντησή σας που δεν μπορώ να καταλάβω. Λέτε ότι για τις περιπτώσεις αυτές φαίνεται ότι έλεγχοι δούλεψαν μεν, αλλά δεν ήταν ικανοί να ανοιχνεύσουν το σφάλμα για την περίοδο για την οποία μιλάμε, δηλαδή το πολιετές πλαίσιο, οι έλεγχοι επιτόπου δεν ανοιχνεύουν ε, παρατυπίες ή σφάλματα σε αιτήσια βάση. Και πώς μπορούν όμως ταυτοχρόνως να μην τα εντοπίζουν. Μπορείτε να εμβαθύνετε σε αυτό το θέμα. Ποιες είναι οι δράσεις που θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να είναι πιο αποτελεσματικά τα συστήματα ελέγχου. Και δεύτερο ερώτημα. Ε, η ετήσια έκθεση ε, της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης. Υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις για τα συστήματα ελέγχου σε διάφορα κράτη-μέλη για 38 επιχειρησιακά προγράμματα και 75 εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό που ε, διακυβεύεται. Και λέει η ετήσια έκθεση ότι ο κίνδυνος ανεπαρκειών του συστήματος εκπεφρασμένος ως ποσοστό ε, για την περίοδο 2007-2013 ε, για τις προσωρινές πληρωμές για το 2009 είναι χαμηλός και σε ποσοστό είναι 1,6%. συμφωνώ είναι ε, χαμηλός συστημικός ε, κίνδυνος αν θέλετε. Ωστόσο στην ίδια έκθεση η ίδια Γενική Διεύθυνση αυτή καθ' αυτή παραδέχεται ότι ίσως ε, δεν εκφράζεται αυτό το ποσοστό του όλες τις διαστάσεις. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί που υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εντοπισμό τέτοιου είδους ελλείψεων ή ανεπαρκειών. Επίτροπε Χάν, στην έκθεσή σας φαίνεται ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης, οι εκθέσεις διαδικολόγησης για 46 προγραμμάτα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Είμαστε στο 14% σε σχέση με το σύνολο των προγραμμάτων. Είναι χαμηλό το ποσοστό αυτό και είναι αρκετά ανησυχητικό. Ε, ποια είναι τα εμπόδια, που, τα πιο βασικά που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη και τι είδους δράση έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπερπηδηθούν. Ποιοι είναι οι τομεί με τον υψηλότερο κίνδυνο ποιου έχετε εντοπίσει ω τέτοιου εσεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να υποβάλω και ένα αίτημα για κάτι που ανέφεραν και οι συνάδελφοί μου. Για να κάνουμε εμεί καλύτερα τη δουλειά μα στην Επιτροπή μα. Χρειαζόμαστε πιο συγκεκριμένα στοιχεία, πιο ακριβείς πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πληροφορίες για τις αδυναμίες αλλά και για τα ισχυρά σημεία αναπολιτικές και ανακράτη-μέλη, γιατί μόνο αν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε τα ποσοστά σφάλματος ανακράτος μέλους και να αξιολογήσουμε το κατά πόσο λειτουργεί τελικά το σύστημα και μόνο έτσι θα είμαστε σε θέση να αποφασίσουμε κατά πόσο πράγματι ε, προστατεύονται τα συμφέροντα των Ευρωπαίων ε, φορολογουμένων. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος Άντορ. Ευχαριστώ. Ως προς ε, το ερώτημα για το οποίο μιλάμε, κυρίως το πρώτο σκέλος του, δηλαδή την αποτελεσματικότητα του ελέγχου, θα ήθελα να σας πω ότι ε, μιλήσαμε όντως για περιπτώσεις όπου λειτουργήσε με το εφιστάμενο σύστημα αλλά δεν εντόπισε επαρκώς τα σφάλματα. Παραδέχομαι ότι δεν είναι αυτονόητη η εξήγηση αυτής της πρότασης ε, υπάρχει όμως αυτή η διατύπωση για να περιγράψει τις καταστάσεις ε, για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί ένα σχέδιο δράσης και θέλει να δει την εφαρμογή του. Και ε, σε πιο συγκεκριμένες περιπτώσεις είχαμε διορθώσεις από 5% μέχρι και 25%. 25% βέβαια μόνο κατεξαίρεση. Και γίνεται λόγος για περιπτώσεις όπου τα περισσότερα σφάλματα που ανοιχνεύτηκαν από το ελεγκτικό συνέδριο θα μπορούσαν να είχαν εντοπιστεί μόνο με έλεγχο επιτόπου. Και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι λειτουργούμε σε ένα πολιετές ε, πλαίσιο ε, και γίνονται έλεγχοι επιτόπου όχι απαραίτητα αμέσως μετά το κλείσιμο των κατατόπους προγραμμάτων, αλλά αργότερα, λόγω των προθεσμιών που υπάρχουν για την υποβολή εκθέσεων και απολογισμών. Επομένως, ε, υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις που η κατάσταση έχει ως εξή. Όντως λειτουργεί ο έλεγχος, αλλά δεν μπορεί να αναχνεύσει το σφάλμα. Και γι' αυτό σημασία για μας έχει να αναλύσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο έχει σχεδιαστεί το σύστημα για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά του, όπως είπα και προηγουμένως. Βεβαίως κάποια σφάλματα θα, παραμείνουν, ε, θα παραμείνει αδύνατο να ανεχνευθούν χωρίς έλεγχο επιτόπου. Αυτό είναι και το νόημα της διατύπωσης σε αυτό το σημείο της έκθεσης. Ευχαριστώ. Κύριε Σχάν, μπορώ να συμφωνήσω και εγώ σε πολλά σημεία της παρέμβασης του συναδέλφου κύριου Άντζορ. Ως προς την ε, ποιότητα, ένα σημείο, εάν εντοπίζονται το 30% δεν μπορεί να είμαστε ικανοποιημένοι με το αριθμητικό αυτό στοιχείο. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Λοιπόν, προσπαθούμε και με την κατάρτιση, με πολλά προγράμματα κατάρτισης του, του προσωπικού στι διάφορες περιοχές, να ενισχύσουμε την ποιότητα. Έχουμε να κάνουμε με περιπτώσεις όπου με την επιμόρφωση έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, έρχεται μια πολιτική αλλαγή, αλλάζουν και τα πρόσωπα που έχουμε επικεφαλής ε, σε μια υπηρεσία ε, και τα οποία έχουμε ήδη επιμορφώσει και καλούμεθα να αρχίσουμε από το μηδέν. Πάλι αυτή η προσπάθεια της επιμόρφωσης. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα δεν ξέρω αν μπορούμε να το αλλάξουμε, να το επιλύσουμε καλύτερα, αλλά προσπαθούμε τουλάχιστον με τα κράτη-μέλη στις συνομιλίες που έχουμε να εξηγήσουμε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίσουμε παγίως. Και όχι μόνο σε επίπεδο νέων κρατών μελών και τα παλαιότερα κράτη-μέλη ε, εμφανίζουν αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, εμείς χρειαζόμαστε και σταθερότητα σε επίπεδο διοίκηση. Σταθερότητα η οποία μπορεί να μας εξασφαλίσει αυτή την ποιότητα. Πάλι για τα ε, εκκρεμή προβλήματα των κοινών προγραμμάτων. Θα παρακαλώ τον κοινικό Διευθυντή κύριο Άνερ να μας πει πέντε λόγια, αν και νομίζω ότι ήδη γνωρίζετε αρκετά. Στα τέλη της ε, περασμένης χρονιάς, σε κάποια προγράμματα η αξιολόγηση όντως του συστήματος ελέγχου ήταν ε, ατελής. Δεν είχε ολοκληρωθεί. Αυτό είναι σαφές. Έκτοτε όμως, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Έξι ε, προγράμματα μένουν εκρεμή, όπου υπάρχει πρόβλημα με την αξιολόγηση του συστήματος ελέγχου και γι' αυτά δεν πληρώνουμε μέχρι στιγμής. Τα δύο ε, αφορούν στη Γερμανία και ένα-δύο στην Ιταλία. Ωστόσο, γιατί υπήρξε αυτή η καθυστέρηση. Ε, πολύ συχνά αυτό οφείλεται σε εσωτερικά προβλήματα ε, μέσα σε, κάθε, σε κάθε κράτος μέλος. Για παράδειγμα, αρμοδιότητα ε, μεταξύ περιφερειακών αρχών και κεντρικής αρχής μέσα στο κράτος μέλος. Ή ε, προβλήματα μεταξύ της αρχής διαχείρισης και της αρχής ελέγχου. Οι δύο αρχές αυτές μέσα στο κράτος μέλος δεν μπόρεσαν να συνοηθούν σωστά. Και όλα αυτά συνιστούν τις αιτίε για την πολύ ε, δυστυχή, αν θέλετε, κατάσταση που σημειώθηκε ε, πέρσι. Όμως δουλεύουμε σκληρά ε, για να ολοκληρωθεί και ο έλεγχος με αυτά τα έξι επιχειρησιακά προγράμματα. Ο κύριος Σκίνερ, σας ευχαριστώ. Αξιότιμη κύριοι Επίτροπη, σας ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Σας έχω αποστείλει διάφορες επιστολές, παρακολουθώ και τη συζήτηση και θα ήθελα να πω ότι πολλοί στην Ανατολική Αγγλία θα εξανίσταντο ακούγοντας ότι ο ορισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι και ο λόγος για τον οποίο χάσατε δουλειά τους. Μιλούμε για μια πολύ σοβαρή και πολύ μεγάλη μετεγκατάσταση εργοστασίου από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Πολωνία που μεταφράζεται σε απώλεια θέσεων απασχόλησης. Θα έπρεπε να ξέρετε ή κάποιος θα σας έχει πει ότι είναι ένα τεράστιο εργοστάσιο και όχι μια μικρομεσαία επιχείρηση, η Twinings, που φτιάχνουν τα φακελάκια τσαγιού και θα έπρεπε να ζητήσετε τα χρήματα πίσω. δεν μπορεί να λέει ένας ορισμός ότι οι νεοσυσταθήσεις επιχειρήσεις μπορεί να είναι επιλέξιμες, δηλαδή ε, αλλιώς τεράστια ε, κονδύλια και πράγματα μπορεί να μεταφερθούν από τη Γερμανία στη Τσεχία. Ίσως ε, μας πιάσανε κορόιδα και θα έπρεπε να το πούμε. Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να ταιριάζουν και να προσαρμόζονται με το βεληνικές της Τη κάθε κατάσταση. και ελπίζω να εξετάσετε το θέμα σε βάθο. Ευχαριστώ. Σα επιβεβαιώνω ότι όντω θα επαληθευτεί. Έχουμε να κάνουμε δύο κράτη και άρα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε και για το μέλλον στοιχεία για να ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Πάντω δεν έχουμε εισαγάγει κάποια όρια ή κατόφλια τα οποία να σημαίνουν περισσότερη ανοχή ή ε, ελαστική ορολογία, ημεροληπτική ορολογία ως προς τον ορισμό της μικρομεσαίας επιχείρησης. Αλλά γεγονός είναι ότι κατά την επαλήθευση της αιτήσεως στην Πολωνία, οι πολωνικές αρχές, στηριζόμενες στην εν λόγω αίτηση, έλαβαν τουλάχιστον καταρχάς τη σωστή απόφαση στο πλαίσιο του αιτήματο του σχετικού με το σχέδιο, όπως είχε κατατεθεί το αίτημα και όπως είχε περιγραφεί το σχέδιο μέσα στο αίτημα. Φαίνεται όμως ότι τα πράγματα δεν ήταν όπως φαινόντουσαν. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έδωσα εγώ την εντολή να διερευνηθεί η υπόθεση. Παρακαλώ όμως και ε, να δείξετε και κατανόηση ότι για λόγους σεβασμού προς το κράτος δικαίου, προς αρχές του δικαίου, δεν μπορώ να σας δώσω ιεσδήποτε ενδείξεις ως προς την κατάληξη αυτής της υπόθεσης. Πάντως έχουμε ευαισθητοποιηθεί και επαληθεύουμε αυτή την υπόθεση. Οι πολωνικές αρχές σας διαβεβαιώ ότι έλαβαν με βάση τα στοιχεία που τους είχαν υποβληθεί καταρχάς τουλάχιστον τη σωστή απόφαση. Ευχαριστώ. Ολμπριχτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη Επίτροπη. Επίτροπη. Διατηρώ κάποιες αμφιβολίες ως προς την ερμηνεία που δίδονται που δίδεται στα στοιχεία, τα αριθμητικά. Μετά τη μεγάλη αλλαγή στην πολιτική συνοχή, ορισμένοι εξημών δήλωσαν ότι το εγχείρημα ήταν επιτυχημένο και άλλοι δήλωσαν ότι το εγχείρημα ήταν απολύτω αποτυχημένο ε, χρησιμοποιώντας τα ίδια νούμερα, ακριβώς τα ίδια νούμερα. Και αν δεν ήταν καταστροφικό το αποτέλεσμα ή τουλάχιστον ήταν εκεί κοντά. Ε, Θέλω λοιπόν να θέσω το ερώτημα στους εκπροσώπους του ελεκτικού συνεδρίου, διότι εκείνοι διεξήγαγαν το έλεγχο. Μπορούν να μας διαφωτίσουν, να συνειδητοποιήσουμε καλύτερα τι συμβαίνει. Προσπάθησα λοιπόν να μάθω τα νούμερα. Και ξέρετε, σε αυτό τον οίκο έχω ακούσει ότι, για παράδειγμα, το 35% των σφαλμάτων σημαίνει αυτό κτλ. Το οποίο δεν ισχύει. Σημειώνω λοιπόν ότι από την ποσόστοση αν θέλετε, το 36% ε, επηρεάζεται από τα σφάλματα, ένα ή περισσότερα. Τώρα, από αυτό το 36% μόνο μέρος είναι ποσοτικοποιημένα σφάλματα. Δηλαδή δεν είναι 36% αλλά είναι για παράδειγμα το μισό του 36%. Και μετά γίνεται λόγος για το 5% ή και το 3% αν θέλετε, γιατί αυτό που είπατε εσείς είναι ότι δεν είχαμε μείωση από το 11% στο 5% αλλά 11, από το 11% στο 3%. Ε, ε, κάνουμε ένα άλμα δηλαδή από το 11% στο 3%. Ε, τι θέλει λοιπόν το ερώτημα, ποια πολιτική συζήτηση θέλετε να γίνει. θέλετε να συζητήσουμε τι συνέβη και κάναμε αυτό το άλμα από το 11% στο 3%, στο 3 ή έχουμε μη πληρωμές, κάτι το οποίο στατιστικώς δεν θα πρέπει να υπαϊσχύει. Είναι δυνατό από το 11 στο 3 ή πώς θα δούμε τελικά τι συνέβη. Ίσως το 11%, ήταν, το 11 ήταν λάθος. Μπορεί κανείς να πει ίσως να πει ότι δεν γίνονται καθόλου πληρωμές. Μιλούμε για ένα έτος. Ε, πείτε μας τι ακριβώς συμβαίνει. Ήρθα εδώ ε, θετικά διακείμενος και άκουσα πολλά αρνητικά και ανησυχώ τι συμβαίνει, μήπως, είναι, ε, μήπως κάτι πάει στραβά και έχουμε τόσο χαμηλό ποσοστό. Και από εκεί και πέρα, πώς το ελεγκτικό συνέδριο αποφασίζει ποιες περιφέρειες ή ποια κράτη θα ε, ερευνήσει, αν θέλετε, θα ελέγξει. Ε, κατά τύχη υπάρχει ειδική μεθοδολογία. Δώστε μας τα στοιχεία. Πώς, ποια είναι τα κριτήρια. Είναι πολιτική απόφαση. Ε, ότι να πάρουμε το χειρότερο δυνατό σενάριο, όσους έχουν τις χειρότερες επιδόσεις ή όσους έχουν τις καλύτερες ή να διαβουλευτούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποφασίσουμε ποιους θα ελέγξουμε. Δηλαδή του χρόνου μπορείτε να πείτε δεν είναι 3 αλλά είναι 5% γιατί θα έχετε αλλάξει ε, αυτό το συντελεστή των σφαλμάτων αν θέλετε. Κάτι πάει λάθος επίσης με το θέμα των ε, δημοσιών ή κρατικών προμηθειών. Εκεί παραμένουν τα προβλήματα. Τι ακριβώς γίνεται εκεί. Ε, σημειώνεται απουσία, έλλειψη ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ε, διαπράττονται λάθη από πλευράς κρατών μελών ή σημειώνονται σφάλματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ τα κάνουν σωστά οι, ε, τα στελέχη των κρατών μελών. Ακούμε στοιχεία από διαφορετικές πηγές και έχουμε την εντύπωση ότι ο, καθένας έχει διαφορετικές διαφορετικά στοιχεία στη διάθεσή του για το θέμα των δημοσίων προμηθειών. Και ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να αποφθύνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως δεν μπορεί να μας απαντήσει σήμερα, ωστόσο θα το θέσω. Μιλούμε για τις ανακτήσεις των κονδυλίων και εμείς στη δική μας επιτροπή δεν είχαμε το νούμερο που μας αναφέρατε, τα 700 εκατομμύρια, αλλά πολύ περισσότερο, ένα νούμερο πολύ μεγαλύτερο. Άρα επανέρχομαι στο πρώτο ερώτημα πώς ερμηνεύονται τα αριθμητικά στοιχεία που παρουσιάζει το ελεγκτικό συνέδριο, πώς επιλέγει πού θα κάνει ελέγχους το ελεγκτικό συνέδριο και τι γίνεται με τις δημόσιες προμήθειες. Αυτά είναι η περίληψη των ερωτήσεών μας. Η κυρία Λάιντ, σας ευχαριστώ ε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να εξηγήσω την κατάσταση. Ε, Ήθελα να κάνω αυτό το σχόλιο και πριν, ότι το αποτέλεσμα εξαρτάται και από τον τρόπο με τον οποίο έχει συλλεχθεί το δείγμα. Ε, το ελεγκτικό συνέδριο μπορεί να ελέξει ε, τις πληρωμές που έχουν δηλωθεί και τις προσωρινές και τις ε, τελικές μετά και τις επιστροφές. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις προκαταβολές. Επομένως, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε ποιος έχει δηλώσει τι, πόσα πολλά επιχειρησιακά προγράμματα, το ύψο όλων αυτών, 10, 20, 30 δις κτλ. Αυτό δεν μπορούμε να το λέξουμε καθόλου. Κάθε ευρώ που δαπανάτε το προσθέτουμε και με τελείως τυχαίο τρόπο διαλέγουμε 180 ε, συναλλαγές αν θέλετε. Ε, καταρχάς ε, επιλέγουμε χ αριθμό επιχειρησιακών προγραμμάτων και μέσα σε αυτά τα επιχειρησιακά προγράμματα επιλέγουμε ψ αριθμό ε, προγραμμάτων. Και γι' αυτό είχαμε 20% πριν από κάποια χρόνια, 11% πέρσι και 3% ε, Έχετε δίκιο. Είναι συγκρίσιμα αυτά τα αριθμητικά στοιχεία. Όλα αυτά είναι προϊόντα της ίδιας μεθοδολογίας. Δεν διαβουλευόμαστε με κανέναν. Έχουμε ένα τυχαίο δείγμα, απολύτως τυχαίο δείγμα, αλλά μόνο από τις πληρωμές για τη δεδομένη χρονιά. Επομένως, αν είχαμε χαμηλό όγκο πληρωμών τη συγκεκριμένη χρονιά, ίσως ε, το δείγμα τελικά είναι λιγότερο αντιπροσωπευτικό για το σύνολο της περίοδου. Το είπα και στην εισαγωγική μου ομιλία. Ε, για κάποια χρονιά μπορεί να υπάρχουν διάζοντα χαρακτηριστικά. Εάν, για παράδειγμα, ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα ε, διοχετεύει ε, λιγότερα κονδύλια ή λιγότερα κονδύλια, υπάρχουν επιστροφές λιγότερες, είναι πιο δύσκολο να ελεγχθούν οι δηλώσεις. Γι' αυτό και δυσκολεύομαι να σας δείξω πώς έχει επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Επιμένω όμως, η δειγματοληψία γίνεται με τελείως τυχαίο τρόπο και στο παρελθόν και στο παρόν και στο μέλλον. Η, η συνθήκη μας επιβάλλει κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά ελέγχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπ' αυτή την έννοια δεν έχει σημασία ποιο κράτο μέλο ελέγχουμε. Πάντοτε με τυχαίο τρόπο λαμβάνονται τα δείγματα και αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε. Τώρα, ω προ τι ε, δημόσιες προμήθειε. Ε, τα ασφάλματα που εντοπίσαμε, συμφωνούμε και η Επιτροπή και εμείς και η ομάδα ελέγχου στο τέλος συμφωνούν τα ευρήματά μας. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά. Εάν το σφάλμα δεν είναι σοβαρό ή δεν είναι ποσοτικοποιημένο λόγω απουσίας στοιχείων, το ελεγκτικό συνέδριο δεν θα το ποσοτικοποιήσει, άρα δεν θα έχει επίπτωση στο ποσοστό σφαλμάτων, στο συντελεστή αν θέλετε σφαλμάτων. Εάν είναι σοβαρό θα ποσοτικοποιηθεί 100%. Τώρα, το σύστημα ποσοτικοποίησης που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διαφορετικό, γιατί ως Επιτροπή αυτοί θέλουν να διαχειριστούν τις δαπάνες. Όταν εμείς ε, υιοθετούμε την εξή θέση και λέμε εάν το σφάλμα ήταν σοβαρό στις δημόσιες προμήθειες το 100% είναι μη επιλέξιμο, στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να υιοθετήσει την εξή άποψη. Ακόμα και αν αγόρασαν κάτι χωρίς τη σωστή διαδικασία, κάποια χρήματα ξόδεψαν. Μπορεί να το πήραν πιο φτηνά, αλλά ε, για λόγους φάλματος μπορεί να ζητήσουν ανάκτηση. Αυτή είναι οι μάνατζερ, αυτοί είναι αυτοί που διαχειρίζονται, επομένως έχουν διαφορετική προσέγγιση. Εμείς είμαστε οι ελεγκτές. Ελπίζω να ε, διευκρίνησα και να ήμουν σαφής στις εξηγήσεις μου. Αν θέλετε, ε, συνεχίζουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χάν. Ναι, επιβεβαιώνω καταρχήν αυτά που είπε η κυρία Καριολάιντ όσον αφορά τις ε, διαφορετικές ερμηνείες. Όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες, ε, το ελεγκτικό συνέδριο έχει όντως αυτήν την άσπρο-μαύρο αντιμετώπιση και προσέγγιση, ενώ εμείς έχουμε μία προσέγγιση λίγο διαφορετική. Δεν είναι ναι όχι άσπρο-μαύρο, εμείς έχουμε ε, αξίες ε, διόρθωσης 2, 5, Η πεποίθησή μας ε, είναι λίγο διαφορετική και ο μηχανισμός διόρθωσης εφαρμόζεται σύμφωνα με τις αντιλήψεις μας. Βεβαίως, σε βάθος χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε πολύ διαφορετικούς υπολογισμούς. Πέραν τούτου, το θέμα των δημοσίων προμηθειών παραμένει σημαντικό πρόβλημα. 85% ε, των λαθών αφορούν ακριβώς τις δημόσιες προμήθειες και η πολιτική συνοχή ε, στην ουσία είναι λίγο καπανέας για τους άλλους ε, τομείς. Άλλοι αποφασίζουν, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστούν οι υπόλοιπες πολιτικές και εμείς αντιμετωπίζουμε και την ευθύνη των αποτελεσμάτων βέβαια ε, και από καιρού εις καιρών σκοντάφτουμε σε κάποιο πρόβλημα και ο κύριος, ο Βανία και εγώ ο ίδιος έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας που ασχολείται ακριβώς με αυτά τα προβλήματα και βλέπουμε κατά πόσον ε, είναι δυνατόν να βελτιώσουμε την ε, κατάσταση και βεβαίως θα ήθελα να γίνει μια πιο διαρθρωμένη συνεργασία με το ελεγκτικό συνέδριο έτσι ώστε ώστε από την πλευρά τους να μας δώσουν ε, κάποιους τρόπους ή κάποιες ιδέες γιατί πιστεύω ότι είναι προς όφελος όλων να οργανωθούν τα πράγματα με τρόπο τέτοιο ώστε οι, οι, αυτές οι απαιτήσει των δημοσίων προμηθειών να γίνονται ε, σωστά και προς όφελος τελικά της εσωτερικής αγοράς. Ε, μερικές φορές ε, υπερβάλλουμε, προχωράμε υπερβολικά μακριά. Ε, λόγω εσφαλμένης ερμηνείας φτάνουμε σε πολλαπλασιασμό λαθών που εμείς θέλουμε να μειώσουμε. 7,7 δις για τις δύο περιόδους 94-2006 είχαμε 23 ε, εκατομμύρια ε, επικάλυψη. Όσον αφορά ε, τα υπόλοιπα αποθεματικού είναι μέχρι το 2006 αλλά δεν έχουν ακόμα ε, ε, ε, καταχωριστεί και θα δούμε πώς θα κλείσουν οι λογαριασμοί στα πλαίσια των συζητήσεων με τα κράτη-μέλη. Αλλά βεβαίως θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Κύριε... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. ερώτηση υπαριθμών 28 για τα περιφερειακά ταμεία και για τα σφάλματα τα οποία έχουν ήδη επιβεβαιωθεί και τις πάυσεις πληρωμών ε, για τα περιφερειακά ταμεία. Στην απάντησή σας διαφαίνεται η περιπλοκότης του ζητήματος που ούτως ή άλλως καταδεικνύεται και από τον πίνακα. Αλλά βεβαίως εξαρτάται πολύ και πώς, πώς ερμηνεύει κανείς, πώς διαβάζει και πώς ερμηνεύει τις, τους πίνακες. 2,7 δις διαβάζω εδώ, διορθωτικά ποσά και ένα δις ε, για χρήματα επιπλέον. Αλλά αυτά είναι πάρα πολλά χρήματα. Εγώ θα ήθελα δύο λεπτά να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Διορθωτικά, εάν αν καταλαβαίνω καλά, αυτό ε, αφορά την, ε, τη διαπραγμάτευση που έχει γίνει με τα κράτη-μέλη και εν πάση περιπτώσει αυτό που είναι διατεθειμένα τα κράτη-μέλη να δεχτούν ή τέλος πάντων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι θα πρέπει να το δεχτούν. Πώς γίνεται ο διάλογος αυτός, πώς φτάνει κανείς σε αυτά τα ποσά, σε αυτά τα, τα στοιχεία, ποια είναι η πρόταση των κρατών μελών, ποια είναι η αντιπρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πώς επιτυγχάνεται αυτός ο συμφωνημένος ε, αριθμός, το ποσό των 2,7 δις. Θα θέλαμε να ξέρουμε λίγο επίσης να δούμε πώς καλύπτεται η απόσταση ανάμεσα στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ε, διάθεση των κρατών μελών. Πόσο δρόμο έχει διανύσει η μία και η άλλη πλευρά μέχρι να φτάσουν σε αυτό το συμφωνημένο ποσό. Επίσης, εάν δεν κάνω λάθος, έχουμε 43 παύσεις πληρωμών. Εγώ ήθελα να καταλάβω πώς λαμβάνουν χώρα αυτές οι παύσεις, ε, ε, ε, δηλαδή πώς, πώς γίνεται ακριβώς αυτή η παύση και επίσης ποιες είναι οι αρχές που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ερώτηση που έχω υποβάλει και γραπτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν, πρέπει, όταν αποφασίζει ότι θα προχωρήσει σε διακοπή ή παύση πληρωμών, ποια στοιχεία ακολουθεί μου φάνηκε ότι κατάλαβα ότι υπάρχει μια τεχνική διαδικασία και μια πολιτική διαδικασία. Εγώ θα ήθελα να ξέρω ποια είναι τα κριτήρια που εφαρμόζει τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ποιες περιπτώσεις και σε ποια, και σε ποια ποσά. Θα ήθελα κάποια αποσαφήνιση από αυτού. Ερώτηση 29 για τις ε, εθνικές δηλώσεις. Και εδώ να σταθούμε λίγο. Υπόθηκε ότι δεν μπορούν να υποχρεωθούν τα κράτη-μέλη να ε, υποβάλουν αυτή τη δήλωση. Όμως, πριν από έξι χρόνια, καμία χώρα δεν το ήθελε. Ήδη έχει αλλάξει αυτό. Έχουν αλλάξει οι νοοτροπίες. Έξι χώρες έχουν μείνει οι οποίες δεν δέχονται έστω και αν δεν μπορεί να υπάρξει ε, υποχρέωση, το να επιβληθεί υποχρέωση στα κράτη-μέλη, πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια μέσα πίεσης. Ε, ε, ώστε να λάβουν τις ευθύνες τους τα κράτη. Και ίσως την επόμενη φορά να διαπιστώνουμε ότι δεν είναι μόνο τέσσερα, έξι μπορεί να είναι, ακόμα και οχτώ, τα οποία το τηρούν. Τι είδους λοιπόν στρατηγική έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να θέσει σε εφαρμογή αυτό το θέμα. Απάντηση. Καταρχάς για το δείγμα. Σημαντικό νομίζω είναι να γνωρίζουμε ότι το 2009 έχουμε περίπου 2 τρίτα των εξαστικών περιπτώσεων που τήρησαν τις προδιαγραφές. Αυτή είναι η υπαγωγή ε, για την όλη δημοσιονομική περίοδο. Τώρα για τη διόρθωση. Πρόκειται για έκφραση ή αποτέλεσμα του προγράμματος δράσης και των νέων κανονισμών. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα τέτοιο μέσο στη διάθεσή μας, την διακοπή που προηγείται, την διακοπή μάλλον προηγείται της παύσης. Σημαίνει ότι ο αρμόδιος δημοσιονομικός διαχειριστής που είναι ο Γενικός Διευθυντής βλέπει νόμιμο έρισμα θεωρεί ότι είναι θεμητό δηλαδή ορισμένες περιπτώσεις ανεξαρτήτως ποσού, γιατί δεν πρόκειται για ένα μικρό, για ένα μεγάλο ποσό πάντα, ανεξαρτήτω ποσού, επαναλαμβάνω, ακόμα και για 2 ευρώ ή για 200 εκατομμύρια ευρώ, σφάλμα να το καθιστά σαν περίπτωση περίπτωση παραδειγματισμού. Φυσικά πάντα υπάρχει μια στάθμιση. Λέμε ότι δεν μετράει το ποσό, αλλά πάντα υπάρχει μια στάθμιση ε, του πώ χειριζόμαστε την κάθε περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, σημαντικό είναι να γνωρίζουμε, πέραν αυτής της, αυτού του περιθωρίου κρίση του Γενικού Διευθυντή, ότι δεν υπάρχει πολιτική πίεση, αλλά είναι γεγονός το ότι το ελεγκτικό συνέδριο και εμείς έχουμε μία στάση ως ελεκτικές αρχές έναντι του κράτους το οποίο ελέγχεται στο οποίο διαπιστώνονται κάποιες παρατυπίες, το οποίο θα έρθει να απαντήσει μετά να πει όχι δεν έχει συμβεί αυτό. Υπάρχουν συζητήσεις, αντιπαραθέσεις μπορεί να προσπαθήσει να μας πει στο κράτος μέλος Φερρυπίν ότι δεν είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα ή ότι έχει διαφορετικά στοιχεία πάνω στα οποία στήριξε τις εκτιμήσεις του. Η προσωπική αυτή επικοινωνία και η ανταλλαγή εγγράφων μερικές φορές ε, αποδεικνύει, γιατί η ανταλλαγή εγγράφων μερικέ φορέ πρέπει να περάσουμε από τη μετάφραση κτλ. Αποδεικνύεται ίσω ανεπαρκή και άρα η προσωπική επικοινωνία ίσω είναι πιο αποτελεσματική αποτελεσματική και ως προς το να αξιολογήσουμε τον βαθμό στον οποίο θα γίνει η διόρθωση. Αυτό, επαναλαμβάνω, το πρόκειται για διόρθωση συστημικών σφαλμάτων, όπου ε, επιβάλλουμε ένα flat rate, ένα συγκεκριμένο ποσό, χωρίς να θέλω να δώσω συγκεκριμένες ε, ενδείξεις. Ξέρετε τι σημαίνει ακριβώς σαν ιδέα το να διακόπτεται η καταβολή κάποιων ποσών στην υπόθεση αυτή. Έτσι λοιπόν έχουμε προσεκτική στάθμιση των υπέρ και των κατά, βάσει των οποίων λαμβάνεται η απόφαση από τη σχετική την αρμόδια υπηρεσία και βεβαίως το κράτος μέλος πρέπει να δεχθεί αυτή την κρίση, μερικές φορές δεν την δέχεται οπότε καταλήγουμε στο δικαστήριο και ίσως αυτό να μην είναι και χειρότερο τελικά, διότι ένας ανεξάρτητος τρίτος παράγων λαμβάνει την απόφαση. Ας περιπτώσει εμείς αυτό, ακόμα και αν θέλουμε να αποφεύγουμε γενικά τη δικαστική αντιπαράθεση, δεν το βλέπουμε σαν πρόβλημα να καταλήξουμε στο δικαστήριο. Ίσως ε, αν επιτρέπετε να δώσει και ο Γενικός Διευθυντής ορισμένες πρακτικές ενδείξεις για το πώ λειτουργεί αυτή η διαδικασία. Πάντως, για να δώσουμε την αποτελεσματικότητα αυτής ε, της μεθόδου, για εφέτος έχουμε προβεί σε 23 διακοπές καταβολής, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο Γενικό Διευθυντή Διευθυντής, εάν θεωρεί ότι δεν είναι ικανοποιημένο από μία ε, δήλωση, μπορεί να προκαλέσει, να θέσει εκείνη σε αυτή τη διαδικασία της διακοπής. Και Εάν μέσα στο εξάμεινο διευκρινιστεί η κατάσταση, διαλευκανθεί η κατάσταση, τότε έρεται αυτή η διακοπή και συνεχίζει η καταβολή. Εάν μέσα στους έξι μήνες δεν δοθεί ικανοποιητική ε, απάντηση, ως λογική συνέπεια αυτού του προβλήματος, κατά κατατίθεται μάλλον ως αίτημα στο συλλογικό όργανο της Επιτροπής το αίτημα της παύσης χωρίς προθεσμία των καταβολών αυτών. Πρόκειται και ένα μέσο το οποίο φαίνεται τόσο αποτελεσματικό ώστε μέχρι τώρα δεν χρειάστηκε να φτάσουμε μέχρι το αίτημα για την πάυση. Και μάλιστα η διακοπή ήταν μέχρι τρίμηνη στις καταβολές αυτές. Είπαμε 43 μέχρι τώρα και δεν έχουμε ε, παρατείνει πάνω από 16 διακοπές. 43 ήταν περιπτώσει που ερευνήσαμε, 16 ήταν αυτέ τι οποίε δόθηκε, επευλήθη μάλλον η διακοπή. Αποτελεσματικό λοιπόν το, το όργανο αυτό, το μέσο αυτό και νομίζω επιτρέπει και επιβάλλει ουσιαστικά τη βελτίωση των δημοσιονομικών ελέγχων. Ο κύριο Άνερ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν τρεις πηγές στις οποίες θα ήθελα να βασιστώ. Πρώτη πηγή οι επιχειρησιακές ομάδες οι οποίες καθημερινά είναι σε επαφή με τις περιφέρειες και πολύ συχνά κάνουν αποστολές, ε, βλέπουν την κατάσταση και επιστρέφουν με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία έχουν συλλέξει. Έχω επίσης και τη δική μου ομάδα ελέγχου, η οποία μεταβαίνει στην περιφέρεια και κάνει ελέγχους. Και η προσέγγιση που ακολουθούμε είναι μια προσέγγιση που εξαρτάται από το κίνδυνο Πηγαίνουμε δηλαδή κατά κύριο λόγο στις περιφέρειες ε, για τις οποίες η ανάλυση κινδύνου που έχουμε κάνει ε, επισημαίνει ε, προβλήματα. Και τρίτη πηγή είναι έξωθεν πηγές, π.χ. το ελεγκτικό συνέδριο, τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια τις δικές τους εκθέσεις, ενδείξεις που έχουμε συλλέξει. Βεβαίως πολλά πρέπει να τα ελέγξω πριν λάβω μέτρα. Και πρέπει να επιβεβαιώσω, να επαληθεύσω ότι, για παράδειγμα, αυτό το οποίο λέγεται σε μια επιστολή που λαμβάνω, όντως απεικονίζει την πραγματικότητα. Για τις περιπτώ... περισσότερες περιπτώσεις ε, συλλέγουμε στοιχεία από τις δικές μας ομάδες, με τις δικές μας αποστολές ελέγχου και μετά μου υποβάλλονται εκθέσεις που επισημαίνουν ενδεχομένως προβλήματα. Με αυτή τη βάση και πάνω σε αυτή τη βάση ακολουθούμε μια εσωτερική διαδικασία, ε, κάνουμε σύσκεψη με όλους τους συναδέλφους που εργάζονται και έχουν ως αντικείμενο αυτή τη συγκεκριμένη περιφέρεια, από κοινού αναλύουμε την κατάσταση και αποφασίζουμε ε, κατά πόσο δεν υπάρχει αξιοπιστία αν θέλετε, υπάρχει έλλειμμα αξιοπιστίας, αξιοπιστίας. και αν συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό όντως αναστέλλονται, διακόπτονται οι, πληρωμές μέχρι να διευκρινιστεί η κατάσταση από πλευράς κράτους μέλους. Σε πολλές περιπτώσεις ε, εφαρμόζεται σχέδιο δράσης στο εν λόγω κράτος μέλος ή στην εν λόγω περιφέρεια και μετά από κάποιους μήνες ξεκινούμε και πάλι τις πληρωμές εκ νέου. Ε, πολύ συχνά αυτό είναι ο λόγος για τις 43 παύσεις ας πούμε που έκανα φέτος. Στις 25 ή 30 φορές από τις 43 έτσι έχει η κατάσταση. Εάν τώρα δεν συμφωνήσουμε ότι κάτι πάει στραβά με το συγκεκριμένο κράτος μέλος, υπάρχει επίσημη, πολύ καλά προκαθορισμένη διαδικασία καθόμαστε γύρω από ένα τραπέζι σε σύσκεψη με δικούς μας εμπειρογνώμονες, με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Όταν υπάρχει λοιπόν ε, διαφωνία με το κράτος μέλος, ε, ακολουθείται μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία και μετά ε, λαμβάνεται απόφαση κατά πόσο θα γίνουν διορθώσεις, θα ανασταλούν, θα πάυσουν οι πληρωμές Σε πολλές περιπτώσεις η εμπειρία μου δείχνει ότι πολύ γρήγορα λύνεται το θέμα. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης αυτές οι διακοπές. Λειτουργούν ε, ενθαρρυντικά ώστε να υπάρξουν γρήγορα συμπεράσματα, να κλείσει γρήγορα η περίπτωση. υπόθεση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω κι εγώ μια ερώτηση προς την Επιτροπή, συγκεκριμένα στον Επίτροπο Με μεγάλη προσοχή διάβασα τις απαντήσεις σας και ε, συνδέοντάς με, το σημερινό, με τη σημερινή συζήτηση βλέπω ότι στην Ιταλία τουλάχιστον, αλλά φαντάζομαι και σε άλλες χώρες, οι μεγαλύτερες αριθμίες παρουσιάζονται στις ε, δημόσιες προμήθειες. δεν αναφέρομαι τώρα ε, μονάχα στο δημοσίευμα των Financial Times γιατί ε, αναφέρεται σε πράγματα τα οποία δυστυχώς γνωρίζουμε καλά και εσείς αναφερθήκατε εις στους ε, ασθενείς. Ναι, αλλά ξέρετε ότι αν η ασθένεια προχωρήσει τότε δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα θεραπείας. Είναι γεγονός λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα της ε, ε, του οργανωμένου εγκλήματος και της πρόσβασης ε, των χρημάτων εκεί. Ξέρετε ότι στο Αμπρούτσο έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο ζήτημα για τις 550 εκατομμύρια ευρώ σχετικά με την χρήση των χρημάτων αυτών για, τις, για την ανοικοδόμηση της περιοχής αυτής μετά το μεγάλο σεισμό. Ακόμα και ο Γενικός Εισαγγελέας Τη της Ιταλίας για το θέμα αυτό ανέφερε ότι εδώ και πολύ καιρό δυστυχώς το οργανωμένο έγκλημα, η μαφία στην Ιταλία έχει απλώσει τα πλοκάμια της ε, στα ευρωπαϊκά χρήματα που φτάνουν στην χώρα. Ε, το έχουμε συζητήσει αυτό και στην Επιτροπή και με τον ε, Επίτροπο κύριο Μπαρνιέ. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να ενισχυθούν τα μέσα και τα εργαλεία του αρχικού ελέγχου και πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχυθεί και η συνεργασία με τα κράτη-μέλη, κυρίως δε με, ε, τα αρμόδια σώματα ελέγχου, ελεγκτικά συνέδρια κλπ. Έτσι ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε ε, εσφαλμένη ή εγκληματική χρήση του δημοσίου χρήματος. Γιατί αυτό εμποδίζει βεβαίως και αμαυρώνει την ε, εικόνα της Ευρώπης. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Και θα σας παρακαλούσα να μας διαθέσετε και όλη την εμπειρία που έχετε συλλέξει στο παρελθόν ως προς τις ε, δυνατότητες προληπτικών ελέγχων. Γιατί, όπως φαίνεται μέχρι τώρα η κατάσταση, λειτουργούν τα συστήματα. Εάν όμως υπάρχουν ενδείξει ότι υπάρχουν παρόλα αυτά κάποιες ε, περιπτώσεις να αντιπαρέλθει κανεί τα συστήματα, τότε θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τα συστήματα αυτά, να τα θωρακίσουμε. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να βελτιώσουμε την ποιότητα των ελέγχων. Διότι δεν μπορούμε να αποσυρθούμε αλλά ή να αφήσουμε σε κάποιον άλλον τη ρύθμιση, της, ε, την αντιμετώπιση κατάστασης, πρέπει ε, να μεριμνήσουμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε εμείς την κατάσταση στην κάθε περιοχή. Γιατί αυτό είναι καθήκον της περιφερειακής πολιτικής. Και ως πρέπει να είμαστε εξίσου καλοί και επαρκείς και διαφανείς σε κάθε περίπτωση. Αυτό σημαίνει και προκαταβολικό αποκλεισμό των περιπτώσεων καταχρήσεων. Γι' αυτό λοιπόν θα σας παρακαλέσουμε να μας δώσετε οποιοδήποτε στοιχείο έχετε. Ο κύριος Σοντή, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ε, και εγώ να, να στηρίξω την άποψή σας ε, για την ενίσχυση της Όλαφ και λυπούμε που διάφορες ε, χειραγωγήσεις ε, και κινήσεις της Βελικής Προεδρίας ε, απομάκρυναν από την Προεδρία έναν πολύ ικανό υποψήφιο. Ευχαριστούμε πολύ την εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου για όσα μας είπε. Με απασχολεί λίγο αυτή, αυτός ο συσχετισμός ανάμεσα στον αριθμό των ελέγχων 180 και τον αριθμό των πληρωμών, τον οποίο αγνοώ. Ε, δηλαδή, τον ε, συνολικό αριθμό πληρωμών για το Ταμείο Συνοχής, έτσι ώστε να ξέρουμε, να βεβαιωθούμε ότι το μέγεθος του δείγματος είναι ορθό σε σχέση με τις διεθνείς πρακτικές ε, οικονομικού ελέγχου προτάθηκε η ιδέα μιας μικρής, μιας μίνιντας στους έξι μήνες. Μήπως, εάν δεν είχαμε ο έλεγχο, θα μπορούσαμε σε επίπεδο δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής να έχουμε μια μαξιντάς, που θα αφορά δηλαδή και τις, ε, ε, τις δημοσιονομικές ε, προοπτικές. Δηλαδή, μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε μία ε, γενικευμένη αξιολόγηση για όλη την περίοδο 6-9 έτσι ώστε να ξέρουμε τι συνέβη ακριβώς και ποια είναι τα λάθη τα οποία ε, παρατηρήθηκαν. Τελευταίο σχόλιο ή μάλλον δύο τελευταία σχόλια όσον αφορά τις ε, μεταφορές έδρας ε, επιχειρήσεων. Ε, άκουσα για την επιχείρηση αυτή η οποία έφυγε από την Ιρλανδία και εγκαταστάθηκε στην Πολωνία. Αυτό καταδεικνύει ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε να μην χρηματοδοτούμε πράγματα τα οποία τελικά θα αποβούν κατά της δημοφιλίας μας και της δημοτικότητάς μας. Και δεύτερον, πιστεύω ότι πραγματικά θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ζητήματα τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τους στην Ευρώπη κινήσεις οι οποίες θα είναι εντός αγωγικών φιλοευρωπαϊκές. Τελευταία παρατήρηση πλέον κύριε Πρόεδρε. Διαπιστώσατε ότι όταν υπάρχει αλλαγή κυβέρνηση αλλάζουν ε, και οι υπάλληλοι που ασχολούνται με τους μηχανισμούς ελέγχου σε εθνικό επίπεδο. Ε, αν ε, όντως ε, υπάρχει αυτό ε, και όσον αφορά τους ελέγχους ε, και όσον αφορά τον οικονομικό έλεγχο τελικά θα κατανοήσουμε αυτό που επανειλημμένα έχουμε πει ότι προφανώς δεν είναι ανεξάρτητες αυτές οι αρχές ελέγχου και επομένως ενισχύεται η θέση μας για συνδιαχείριση. Πρόεδρος, νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Θα δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου και μετά να κλείσουμε. Ευχαριστώ. Μία σύντομη απάντηση. Η μεθοδολογία του ελεγκτικού συνεδρίου έχει υποστεί το peer review, την αναθεώρηση ομολόγων, αλλά έχει εγκριθεί και από διεθνεί εμπειρογνώμονε. Συμφωνούμε με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και λογιστικά πρότυπα. Όλα αυτά έχουν επαληθευτεί από διάφορου συναδέλφου. Ω προ τι δημοσιονομικέ προοπτικέ, αποφασίσαμε για το, τα διαρθρωτικά ταμεία και για την περιφερειακή ανάπτυξη να έχουμε αυξημένο δείγμα για να έχουμε καλύτερη εικόνα της κατάστασης. Για τις δημοσιονομικές προοπτικές θα πρέπει να έχουμε υπομονή. Είχαμε σταδιακή εξάλληψη συγκεκριμένων διαπανών και σταδιακή εισαγωγή νέων διαπανών, phase out και phase in αναλόγως. Έχουμε συγκεκριμένες εβδομάδες ελέγχου ανά έτος ε, είναι σωστή μεθοδολογία αλλά είναι και πολύ δαπανηρή. Εξετάζουμε πώς θα αντιληφθούμε καλύτερα ε, τις πληρωμές που κλείνουν, αλλά είναι πολύ τεχνική αυτή η συζήτηση και αν θέλετε να την κάνουμε εκτός εθούσης μετά, στο τέλος της συνεδρίασης. Ε, κάτι άλλο ήθελα να πω. Με χαρά άκουσα τον εισηγητή να μιλά για τις εκθέσεις ε, που συνοδεύονται και από την, ε, τα σχόλια για τη διαχείριση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για πρώτη φορά άκουσα ότι όντως επηρεάζεται αυτή η συζήτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό δείχνει ότι τα στοιχεία έχουν βελτιωθεί, η ποιότητα των στοιχείων που συλλέγουμε. Υπάρχουν δύσκολες περιπτώσεις, αυτό είναι αληθές, ωστόσο πιστεύω ότι όλοι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος Χάν. Και εγώ, ε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να πω το εξής. Συμφωνώ απολύτως με ό,τι έχει λεχθεί και δεν θέλω να επαναλάβω πράγματα που έχω ήδη πει. Καλό θα ήταν να συμφωνήσουμε όλοι ε, πάνω σε αυτό. Αυτό το maxi dash, αυτή η μέγιστη αν θέλετε εξέταση της δήλωσης αξιοπιστίας, ίσως θα ήταν κάποια λύση μόνο εάν συμφωνήσουμε πάνω στη μεθοδολογία, αν θα ασχοληθούμε με το 1 τρίτο π.χ. με κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει αναγνωρίζονται τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού συνεδρίου. Αν μπορούσε το ίδιο το ηλεκτρικό συνέδριο να το κάνει αυτό θα ήταν ιδανικό. Να ασχοληθεί δηλαδή με το Maxi Dash και θα είχαμε ένα αυξημένο επίπεδο ως προς την ε, ποιότητα των στοιχείων. Τώρα, ως προς το σύστημα της των πληροφοριών. Δηλαδή έχουμε τις εκθέσει. έχουμε τη δήλωση αξιοπιστία. Όλα αυτά οδηγούν στο εξή αποτέλεσμα. Εθελούσια όλο και περισσότερα κράτη-μέλη θα προσχωρήσουν σε αυτό το σύστημα εθνικών δηλώσεων. Κατα... Θα έχουν αυτή τη βούληση δηλαδή και αυτό είναι καλό. Η σταθερότητα, ε, τα ακράδαντα, ο χαρακτήρας του ακράδαντος στα στοιχεία αυτά θα σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη δεν θα έχουν πρόβλημα να τα υποβάλουν. Θα είναι οι που ήδη θα διαθέτουν. Δηλαδή, σιγά-σιγά θα αυξήσουμε την αξιοπιστία των εθνικών στοιχείων. Βήμα-βήμα. Ε, Και όλο και περισσότερα μέλη θα προσχωρήσουν σε αυτή, κράτη-μέλη θα προσχωρήσουν σε αυτή την εθνική δήλωση αξιοπιστίας. Πίστευω κραδάντος ότι είμαστε σε καλό δρόμο και αυτά θα επαληθευθούν του χρόνου, θα φανούν και στην πράξη. Κατά τα λοιπά, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ, Επίτροπος Άντορ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι μπορούμε όντως να συζητήσουμε περαιτέρω για τη φύση και για τις συνέπειες της τυχαίας δειγματοληψίας, του τυχαίου στη συλλογή των δειγμάτων. Ωστόσο, το σημαντικό είναι να εστιάσουμε την προσοχή μας στη δουλειά που κάνουμε και στο πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε έτσι περαιτέρω. Αυτό το οποίο πιστεύουμε είναι το εξής. Πέρα από τη βελτίωση των στοιχείων, Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εστιασμένες προσπάθειες και αυτό φαίνεται. Έχει βρει νέες μεθόδους συνεργασίας με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά και με τις εθνικές αρχές και τους κρατικούς φορείς. Και αυτό είναι καλό. Έχουμε την πρακτική των διακοπών και παύσεων ή αναστολών, αν θέλετε, πληρωμών και αυτό είναι επίσης καλό. Η απειλή απώλειας κονδυλίων είναι αποτελεσματική σε επίπεδο κράτους μέλους, όμως θα πρέπει να είναι το απότατο εργαλείο, το τελευταίο μέσο που να χρησιμοποιήσουμε. Ε, θα είναι καλό να έχουμε αναλογική ανταπόκριση, αναλογική απάντηση, να μην υπερβάλλουμε στα σφάλματα που ενδεχομένως μπορεί να σημειώνονται, στα λάθη που μπορεί να διαπράττονται. Αυτά έχουν αντίκτυπο και στην ετήσια εικόνα, αλλά βελτιώνουν και την διαχειριστική ικανότητα, αλλά και τους, τον ποιοτικό έλεγχο ε, που διενεργούν οι εθνικές αρχές. Μένει λοιπόν ε, να βελτιώσουμε ε, τις επιδόσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εγώ βεβαίως σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία και προσδοκώ στη συνέχιση της ανταλλαγής απόψεων με εσάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, υπήρξε ε, με εξαιρετικά επικοδομητική η συζήτηση και πριν ολοκληρώσουμε την συζήτηση θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Χατσμαρκάκη, τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή η οποία ήρθε εδώ απόλυτα προετοιμασμένη ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον ε, κύριο Σμέτα ο οποίος ε, είναι υπεύθυνος για συγκεκριμένα θέματα. Μιλήσατε αγαπητή κυρία Κάλιου για την πλευρά του ελέγχου, από πλευράς ελεγκτικού ε, συνεδρίου. Ε, νομίζω ότι βρισκόμαστε ε, σε καλό δρόμο, μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό. Οπωσδήποτε ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όπως λέει και η παλιά ασιατική παροιμία ε, στόχος ε, είναι ο δρόμος επομένως μας ενδιαφέρει αυτός ο δρόμος προς την αλλαγή του συστήματος. Μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε τα βήματα απλούστευσης για το 2011 και χαιρόμαστε που ακούμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Πάντως όσον αφορά την απαλλαγή δεν ξέρω αν θα έρθει τόσο εύκολα. Θα ήθελα να πω και στον κύριο Χάν ότι φτάνουμε σε ένα πρόγραμμα δράσης ε, με την έννοια μιας εθνικής τοποθέτησης αλλά και γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε τα πράγματα πολύ καθαρά. Ε, υπάρχουν ήδη κάποιες χώρες οι οποίες έχουν δώσει όλα τα στοιχεία, ε, είναι άλλες οι οποίες βρίσκονται σε καλό δρόμο και περιμένουμε, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο πρέπει οπωσδήποτε να ασκήσουμε πιέσει στα κράτη-μέλη. Και θεωρώ πολύ θετική τη στάση σας προς του αυτοματισμού. Έχετε ήδη εξηγήσει ότι δεν υπάρχουν αυτοματισμοί ως προς τη διακοπή ή την πάυση των πληρωμών, έχει, των καταβολών μάλλον, έχετε επισημάνει τη, τα, τα, τα, στοιχεία τα σχετικά με τη ρύθμιση, έχετε καταστήσει σαφές ότι δεν πάει πλέον έτσι και έχετε πολύ καλή και ανοιχτή στάση απέναντι στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά. Απλώ θα πρέπει να μα βοηθήσει αυτή η στάση να ασκήσουμε περισσότερε πιέσει. Δεν μιλήσαμε αρκετά για του μηχανισμού ε, πίεση για το πώ μπορούν να διατεθούν τα κονδύλια. Ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε το πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Πάντως το πώς βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα δεν το έχουμε συζητήσει. Και αυτό πρέπει να είναι ο στόχος της δουλειάς μας. Αποτελεσματικά μέσα, εργαλεία με τα οποία να μπορούμε από κοινού να ε, φέρουμε εις πέρας τη δουλειά μας, την πολιτική μας, αλλά νομίζω ότι έχουμε μπει στο σωστό δρόμο. Οι δημοσιονομικές προοπτικές που έχουμε μπροστά μας τώρα είναι πιστεύω χρήσιμες και για αυτόν τον λόγο μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε, μπορείτε και εσείς να τις αξιοποιήσετε. Ε, συνάδελφοι εδώ, όπως η κυρία Γκρέσλε, ο κύριος Γκάιντ, είναι μέλη στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών και μπορείτε να αξιοποιήσετε τη δική τους βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ και καλή δουλειά από εδώ και εμπρός. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και περάμε στο σημείο 5 της ημερησίας διατάξεως. Δήλωση αξιοπιστίας 2009, αποτελέσματα και τάσεις. Και θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Καλιουλάιντ, ε, εξ ονόματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Παρακαλώ, κυρία Καλιουλάιντ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω μια επισκόπηση των ε, στοιχείων που συνεδεύουν ε, τη δήλωση του Συμβουλίου. Θα ήθελα να επαναλάβω καταρχάς το βασικό μήνυμα του Προέδρου Καλδέιρα για την αξιοπιστία των λογαριασμών. Το ελεκτικό συνέδριο για τρίτη συνεχή χρονιά έχει αποφανθεί ότι οι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζουν μια δίκαιη εικόνα, αν θέλετε, ε, της ε, οικονομικής θέσης και τα αποτελέσματα των ε, συναλλαγών και των ταμιακών ροών. Τώρα, ως προς ε, την νομιμότητα και την ε, κανονικότητα των συναλλαγών θα ήθελα να σας μιλήσω για τα σφάλματα. Στις 1040 συναλλαγές που ελήφθηκαν ως δείγμα για όλες τις ε, πολιτικές, το ελεγκτικό συνέδριο εντόπισε 690 σφάλματα, 170 των οποίων ήταν ποσοτικοποιημένα τα ποσοτικοποιήσιμα σφάλματα είναι αυτά που συμβάλλουν στο συντελεστή σφάλματος. Συνολικά ε, τα σφάλματα είναι παρεμφερή με το, τα στοιχεία στην ετήσια έκθεση για το 2008 του Ελεκτικού Συνεδρίου. Ο αντίκτυπός τους όμως είναι διαφορετικός σε σχέση με το 2008 ε, λόγω ε, του διαφορετικού εύρους και λόγω των αξιολογήσεων της λειτουργίας των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου. Πράγματα δηλαδή που είναι γνωστά ως ε, τα φανάρια αν θέλετε. Δηλαδή, το δεύτερο μήνυμα που θέλω να σας ε, στείλω είναι ότι οι συνολικές δαπάνες επηρεάζονται ουσιοδός από τα ασφάλματα και για αυτή τη χρονιά. Η συχνότητα είναι σταθερή μεταξύ ποσοτικοποιήσιμων και μη ποσοτικοποιήσιμων σφαλμάτων. Δηλαδή, η συχνότητα σοβαρών ποσοτικοποιήσιμων σφαλμάτων, όσα ξεπερνούν το 2%, έχει αυξηθεί, ωστόσο η συχνότητα των περιορισμένων ποσοτικοποιήσιμων σφαλμάτων από μισό μέχρι 2% έχει αυξηθεί. Τι σημαίνει αυτό με δύο λόγια. Ότι παρόλο που ο αριθμός των ποσοτικοποιήσιμων σφαλμάτων παραμένει σταθερός, ο αντίκτυπός τους είναι χαμηλότερος το 2009 συγκριτικά με αυτό το 2008. Αξίζει τον κόπο να δούμε ε, ποια σφάλματα εντοπίζονται κατά κύριο λόγο. Ως προς την ομάδα πολιτικής γεωργία και φυσική πόρη, ε, το είδος σφάλματος έχει να κάνει με την ακρίβεια. Δηλαδή, οι δαπάνες έχουν υπολογιστεί εσφαλμένα είτε από τον δικαιούχο είτε από οποιοδήποτε έχει επεξεργαστεί αυτές τις πληροφορίες στη συνέχεια. Αντιθέτως, για τη συνοχή, το ελεγκτικό συνέδριο βρήκε ότι τα σφάλματα που σχετίζονται με τη μη τήρηση των κανόνων για τις δημόσιες προμήθειες είναι και αυτά που απαντώνται πιο συχνά. Το τρίτο μήνυμα που απέστειλε ο πρόεδρος Καλμπέιρα είναι το εξής. Οι εκτιμήσεις για το πιο πιθανό σφάλμα σε θέματα δαπανών, για θέματα συνοχής αν θέλετε, ήταν σημαντικά χαμηλότερες από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Η σημαντική διαφορά ουσιαστικά αντιστάθμισε ε, λειτουργήσε αντισταθμιστικά με τη μικρή αύξηση ε, στο συντελεστή σφάλματος για τη γεωργία και τους φυσικούς πόρους. Δηλαδή, σε σχέση με το σύνολο του προπολογισμού, οι συνολικέ εκτιμήσει για τα επίπεδα των σφαλμάτων δεν είναι μόνο χαμηλότερε το 2009 από το 2008, αλλά κυμαίνονται για πρώτη φορά από το 2 μέχρι το 5%. Εκεί εντοπίζονται και όχι παραπάνω. Θα ήθελα τώρα να ε, επισημάνω ένα συγκεκριμένο θέμα που έχει να κάνει με τις οικονομικές διορθώσεις ή τις ανακτήσεις. Είναι διαφορετικά πράγματα. Οι ανακτήσεις έχουν να κάνουν με άτυπες πληρωμές που έχουν γίνει σε ατομικούς δικαιούχους, σε ξεχωριστούς δικαιούχους, οι οποίοι πρέπει να επιστρέψουν ε, τα χρήματα που έχουν λάβει κακώς. Επομένως είναι ένας μηχανισμός διόρθωσης φαλμάτων. Ενώ οι χρηματικές οικονομικές διορθώσεις έχουν να κάνουν με αδυναμίες στο σύστημα διαχείρισης. Δηλαδή η Επιτροπή αποσύρει κονδύλια από τα κράτη-μέλη από τρίτες χώρες και ε, για να μην υπάρχουν συνέπειες που θα βαρύνουν τον Ευρωπαίο ε, φορολογούμενο. Ε, εμείς ως ελεγκτικό συνέδριο εστιάζουμε την προσοχή μας στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει αυτούς τους διορθωτικούς μηχανισμούς. Και ε, σημειώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε γενικές γραμμές αναφέρει αξιόπιστα στοιχεία όσον αφορά τις δικές της δραστηριότητα. Ωστόσο, τα στοιχεία των κρατών μελών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι πλήρη και δεν είναι ακριβή στο σύνολό τους. Το 2009 σχεδόν το 90% των επιβεβαιωμένων ποσών και σχεδόν το 80% των εφαρμοσμένων ε, ποσών είχαν να κάνουν με τις διορθώσεις. Καταρχήν, εάν υπήρχαν ε, ολοκληρωμένα και ακριβή στοιχεία για το ύψος των ανακτήσεων από πλευράς κρατών μελών και από την Επιτροπή ως προϊόντα των σφαλμάτων που έχουν ανοιχτευθεί σε συγκεκριμένα έτη, τότε αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ένας πραγματικός δείκτης που να ε, αποδεικνύει την αποτελεσματική λειτουργία ε, των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου. Εξού και έρχομαι στο τέταρτο μήνυμα ε, του ελεκτικού συνεδρίου. Παρά τις βελτιώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι πληροφορίες που έχουμε για τις ανακτήσεις και τις διορθώσεις δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένες και ε, ακριβής. Θα ήθελα να ε, μιλήσω στο τέλος της ομιλίας μου για το μέλλον. Εμείς έχουμε ε, λάβει τα αιτήματα των διαφόρων ενδιαφέρων μελών και θα τα εντάξουμε στις αιτήσει εκθέσεις που θα συντάξουμε στο μέλλον. Βεβαίως έχουμε περιορισμένους πόρους και θα πρέπει να σεβαστούμε και να τηρήσουμε συγκεκριμένα στάνταρ και πρότυπα ελέγχου. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο εφαρμόζουμε την προσέγγισή μας. Για την επόμενη χρονιά θα εμβαθύνουμε στις ομάδες πολιτικής για τη γεωργία και τους φυσικούς πόρους, αλλά και για τη ε, συνοχή. Και θα αυξήσουμε το δείγμα των συναλλαγών που θα ελέγξουμε για να έχουμε πιο συγκεκριμένες αξιολογήσεις για κάθε ένα από αυτούς τους τομείς για το εγχείρημα της δήλωσης αξιοπιστίας για το έτος 2011. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κύριε Ευχαριστούμε και κύριοι βουλευτέ. Θα ήθελα να ευχαριστώ την κυρία Καριολάιτ για την εκτεταμένη αυτή ενημέρωση, την ανάλυση της κατάστασης και την παρουσίαση του κεφαλαίου υπαριθμών 1 του ΙΣΕΚΤΕΣ 2009 του Ελεγκτικού Συνεδρίου καταρχάς με ικανοποίηση σημειώνουμε ότι υπάρχει, επισημαίνεται καλή διαχείριση των κονδυλίων, επισημαίνεται ότι οι ακαταπώνητες προσπάθειές μας έχουν φέρει καρπούς και ιδιαίτερα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού βλέπουμε ότι 95% συνολικά των πληρωμών που κατεβλήθησαν σε κάθε μορφή διαχείρισης ήταν νόμιμα και νομότυπα ποσά. Επίσης, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω για τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταπολεμήσει, να αντιμετωπίσει και να καταπολεμήσει κάθε είδους εναπομείναν πρόβλημα και να εξασφαλίσει τους μηχανισμούς ε, διαχείρισης. Η κυρία Κάλιου Λάιτερ επισήμανε ήδη τη γεωργία και τη συνοχή ως κύριους ε, τομείς, ο οποίος επισήμανε δυσκολίες ως προς την ακρίβεια στις ε, ε, στην ακρίβεια και την διαχείριση. Από πλευρά μα, λαμβάνονται τα μέτρα αντιμετώπισης αυτών των αδυναμιών. Όσον αφορά τη γεωργία έχουν θεσπιστεί μέσα ε, σχέδια δράσης και επιβαλλονται στα κράτη εκείνα στα οποία έχουν ε, εντοπιστεί προβλήματα το 2009 και έχουν οδηγήσει σε σχετικές επιφυλάξεις από την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων από τις σχετικές γενικές διευθύνσεις. Για τα άλλα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2009 ε, έλεγξε τα συστήματά τους, τα βρήκε αποτελεσματικά. Υπάρχει όμως ακόμη περιθώριο για βελτίωση και αυτό το χτένισμα των εισαγωγικών θα το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην συνεργασία με τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη. Επίσης, διαδικασίες ε, Εκαθάριση χρησιμοποιούνται για τον αποκλεισμό από την κοινοτική χρηματοδότηση όποιου δεν τηρεί τους κοινοτικού κανόνες, όπως ορίζεται δηλαδή για τη διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ως προς τη συνοχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη στο ελεγκτικό της έργο έχει ενσωματώσει σφάλματα στις δημόσιες προμήθειες από πλευρά των κρατών μελών σε επίπεδο Άλλα βήματα έχουν ληφθεί όπως σε παραδείγματι η εξειδικευμένη επιμόρφωση για τις διαδικασίες για, ε, τις δημόσιες προμήθειες και ε, καθοδήγηση ή οδηγίες προς τις αρμόδιες αρχές. Πιστεύω ότι έχετε ήδη συζητήσει με τους συναδέλφους Χαν και Άντζορ τα θέματα αυτά. Και με χαρά σημειώνω ότι το ενεκτικό συνέδριο διαπιστώνει βελτίωση του πεδίου και της ενημέρωσης των εθνικών διορθώσεων, όπως καταγράφονται στους λογαριασμούς του όλο του 2009. Όντω δεν είναι, όπως επισημαίνει και το ελεγκτικό συνέδριο, επακριβή, απόλυτα ακριβή και σωστά ή πλήρη τα στοιχεία που προσφέρουν τα κράτη-μέλη στον έλεγχο. Ωστόσο, οι δημοσιονομικές διορθώσεις δεν μπορούν να συγκριθούν απευθεία με το ποσοστό του σφάλματο. Υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες διόρθωση ανάλογα με τη νομική βάση ή τον τρόπο διαχείριση. Και πρώτον, οι δημοσιονομικές διορθώσεις είναι ευθύνη διαφόρων παραγόντων κατά περίπτωση. Στην απευθείας διαχείριση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκομίζει τα ποσά, εξασφαλίζει στην επιστροφή είτε με carry out είτε με ε, διακοπή των μεταγενέστερων πληρωμών των ποσών από τον δικαιούχο. Στην μεικτή διαχείριση περίπου δηλαδή το 80% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, την διόρθωση την κάνει το κράτος μέλους. Και τη δημοσιονομική διόρθωση μπορεί να την επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά έχει να αντιμετωπίσει συστημικά ασφάλματα ή αδυναμίες στο επίπεδο των κρατών μελών και όχι σφάλματα συγκεκριμένα στο επίπεδο του δικαιούχου. Τρίτον, δεν υπάρχει πάντα η αδυναμιες στο επιπεδο των κρατων μελων και οχι σφαλματα συγκεκριμενα στο επιπεδο του δικαιουχου τριτον δεν υπαρχει παντα δυνατοτητα να, να ακτιθούν τα χρήματα. Στη συνοχή επιτρέπεται οι πόροι οι οποίοι ε, απελευθερώνονται λόγω κάποια δημοσιονομική διόρθωση να αξιοποιηθούν σε άλλο πρόγραμμα. Και επιπλέον, συμπληρώνω ότι η διόρθωση είναι μια διαδικασία μακροχρόνια και ένα σύστημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί μακροπρόθεσμα. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με πολυετή συστήματα ελέγχου. Πολλά ασφάλματα τα οποία εντοπίζονται από το ελεκτικό συνέδριο σε ένα συγκεκριμένο έτος θα έπρεπε ή θα μπορούσαν να έχουν εντοπιστεί από τα διορθωτικά ε, συστήματα της Επιτροπής σε μεταγενέστερα έτη. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη στιγμή του κλεισίματος ενός προγράμματος που αποδεικνύει ότι έχει, ότι έχει χαμηλότερο ποσοστό εκτέλεση από την περίοδο εφαρμογής ε, μπορεί να εντοπιστούν τα σφάλματα. Το ίδιο είδαμε στα προγράμματα 94-99. Ενδείξεις δηλαδή ότι αφού έγιναν οι δημοσιονομικές διορθώσεις ή έκλεισαν οι λογαριασμοί, το ποσοστό του σφάλματος μειώθηκε σημαντικά. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει τα κράτη-μέλη της ε, τα καθήκοντά τους. Ιδιαίτερα δε μετά το άρθρο 317 της ε, νέας συνθήκης, το σχετικό με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να καταθέτουν πλήρεις και αξιόπιστες πληροφορίες για τα ποσοστά απορρόφησης και ανάκτησης και βεβαίως με το νέο σύστημα που έχουμε μπορούμε να αποστέλουμε σε μηχανογραφημένη μορφή, σε ψηφιακή μορφή, στοιχεία σχετικά με την ανάκτηση τεκοπιτών πληρωμών. Η Επιτροπή όχι μόνο προσφέρει βοήθεια προς τα κράτη-μέλη, επιπλέον τους ζητεί να βελτιώνουν την ποιότητα των πληροφοριών που προσφέρουν, πέραν και αυτών που απαιτεί ο ίδιο ο κανονισμό. Να βελτιώνει ακόμη περισσότερο την ποιότητα των πληροφοριών. Και αν χρειαστεί, η Επιτροπή θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο του ελέγχου του δημοσιονομικού ελέγχου και την καταγραφή των διορθώσεων. Ασφαλώ αυτή η έλεγχη θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική και ουσιαστική εφόσον τα κράτη-μέλη και οι αρχέ του υποχρεωθούν να καταθέτουν κάθε χρόνο την σχετική ε, δήλωση αξιοπιστία με την πιστοποίηση ενό ανεξάρτητου ελεγκτικού οργάνου, όπω είχε ζητήσει στο Δημοσιονομικό Κανονισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, σκοπεύω, σε συνεργασία με του ε, συναρμόδιου επιτρόπου, να εξετάσω πώ μπορούμε να βελτιώσουμε στην τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο τη λειτουργία των ε, συστημάτων δημοσιονομικού ελέγχου και να βελτιώσουμε τα ποσοστά σφάλματος. Και πριν κλείσω, θα ήθελα, να μου επιτρέπετε, να ε, καλέσω το ελεγκτικό συνέδριο για το 2010 να επεκτείνει το πεδίο έρευνας για το πιστοποιητικό ε, για τη βεβαίωση αξιοπιστίας και, στο και στην ε, γεωργία και τη συνοχή αλλά και το περιβάλλον. Πιστεύω ότι θα δει πολύ καλά αποτελέσματα εκεί. Και η διαδικασία απαλλαγή του 2009 θα ήθελα να πω ότι είμαι βέβαιος πως θα αποδειχθεί χρήσιμη για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Χρειάζεται τώρα μια και δεν έχουμε πια πολύ χρόνο να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατό μέσο για να βελτιώσουμε την απορρόφηση και την ποιότητα χρήσεως των ευρωπαϊκών κονδυλίων γιατί προετοιμάζουμε έτσι το μέλλον και πιστεύω ότι πρέπει να δούμε σημαντικά ζητήματα όπως απλούστευση, προσθέμενη αξία των δαπανών, αποτελεσματικότητα και στρατηγική ελέγχου που στηρίζεται στον κίνδυνο τώρα για να ετοιμάσουμε το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χατζημάρκα, εξωσυγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και καταρχάς ε, θα ήθελα να επισημάνω την κύρια δήλωση του, του κεφαλαίου υπαριθμών 1 ότι το ελεγκτικό συνέδριο διαπιστώνει ότι για 16η χρονιά σημειώνονται σημαντικές ελλείψεις ως προς τις ε, καταβολές κονδυλίων από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι το κύριο στοιχείο και γύρω από αυτό το πρόβλημα περιστρέφονται τα πάντα. Εδώ θα επιμείνω και ευχαριστώ τον Επίτροπο Σμέτα που μίλησε για, την, ε, για το θέμα της εθνικής δήλωσης που βέβαια μας απασχόλησε και στη συζήτηση με τους Επιτρόπους Άντορ και Χάν και είμαι βέβαιος ότι θέλετε και εσείς να ασκήσετε πίεση γιατί είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, ένα θέμα στο οποίο θέλουμε την υποστήριξή σας και στο οποίο θα πρέπει και εσείς να ασκήσετε περισσότερη πίεση προς τα κράτη-μέλη ιδιαίτερος δεδομένων των άρθρων ε, που, του άρθρου μάλλον που αναφέρθηκε από τη συνθήκη. Η έκθεση λοιπόν του Ελεκτικού Συνεδρίου ακολουθεί τον ίδιο μύτο της Αριάδνης, ότι δηλαδή δεν είναι αξιόπιστα τα στοιχεία. Επανέρχεται διαρκώς αυτή η εποδός. Δεν μπορούμε να στηριχθούμε στα στοιχεία, στοιχεία που μας δίνουν τα κράτη-μέλη. Δεν είναι παρκώ ακριβή τα στοιχεία τα συστήματα επιτήρησης, το 3% δεν λέει τίποτα. Η κυρία Καρκουλάιτ μας λέει ότι χρειάζεται περισσότερα δείγματα για να είναι αξιόπιστα τα στοιχεία αυτή. Πολύ καλά. Πλην όμως διερωτώμεθα γιατί το ελεγκτικό συνέδριο δεν πιέζει περισσότερο για, περισσο... για να, να αξιοποιήσει, να αξιοποιήσει συγγνώμη, την πραγματογνωμοσύνη, την εμπειρία, τη γνώση των εθνικών ελεγκτικών συνεδρίων. Γιατί δεν κοιτάτε περισσότερο τα εθνικά και περιφερειακά σε ορισμένε περιπτώσει ελεγκτικά συνέδρια, ώστε να, τους, να τα καλέσετε και αυτά να συμμετάσχουν στον έλεγχο. Θα ήταν πολύ πιο αξιόπιστα τα, τα στοιχεία εάν είχαμε μη τι άλλο φερειπίν κοινέ αρχέ. Ξέρω ότι προσπαθεί το ελεγκτικό συνέδριο. Ξέρω ότι οργανώνει σεμινάρια. Έτσι ώστε να προσδοριστούν κοινέ αρχέ. Εν πάση περιπτώσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν δημιουργήθηκε προχτέ. Γιατί λοιπόν δεν υπάρχουν αυτά τα κοινά συστήματα ακόμα. Γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι κοινέ αρχές. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η συνεργασία. Και γιατί δεν έχουμε περισσότερη επιτυχία τελικά ως ελέγχου. Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω το ελεγκτικό συνεδρίο, αλλά και να το καλέσω να τοποθετηθεί στον τομέα για το θέμα της γεωργίας. Ακούστηκε ότι υπάρχουν τριμερείς συνομιλίες για την συνοχή. Για την ερμηνεία δηλαδή ορισμένων ζητημάτων που καλείστε κυρία Κάλιου Λάιτ να ερμηνεύσετε συζητείτε Φερρυπίν για την, για την συνοχή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς κρίνετε τα θέματα αυτά. Πολύ καλά. Υπάρχουν διάφορα σημεία στα οποία χρειάζεστε την πραγματογνωμοσύνη τη Επιτροπή, την αξιολόγησή τη, τι παρατηρήσει τη. Στον τομέα τη γεωργία όμω αυτό δεν υφίσταται. Και έτσι, το 2009 το αποτέλεσμα ήταν ότι ο τομέας που ήταν πράσινος μέχρι τώρα ήλθε στο χρώμα κίτρινο. Αυτό προκύπτει από την τριμερή ε, συνομιλία ή μάλλον θα μπορούσε να είχε αντιμετωπιστεί αν υπήρχαν οι τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Κομισιών Ελεκτικού Συνεδρίου και Κρατών Μελών. Αυτό νομίζω πρέπει να το λάβουμε υπόψη για το μέλλον στον τομέα τη γεωργία. Ή, εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να μα πείτε γιατί ακόμα δεν έχει εξασφαλιστεί μια βελτίωση. Ξέρουμε ότι είναι βέβαια τα ποσά διαφορετικά. Στη συνοχή είναι μεγαλύτερα τα ποσά από ό,τι στη Γεωργία. Υπάρχει κάποιο τρόπο όμω ε, να διαπραγματευτείτε τα θέματα αυτά ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση για τι δημοσιονομικέ διορθώσει που ανέφερε ο κ. Επίτροπο. Θα ήθελα να επισημάνω και επανέρχομαι στον τομέα της ε, γεωργίας, ότι εδώ ε, ισχύει ο 50-50. Δηλαδή, ένα κράτος μέλος το οποίο αδικαιολόγητα έχει κάνει κάποια πληρωμή, με τήρηση του κανόνα 50-50, θα έχει σε συνέπεια ότι θα πρέπει να ε, ανακτηθούν τα 50, το, το μισό δηλαδή των ποσών από τα ε, εσφαλμένω καταβληθέντα, αλλά το άλλο 50% είναι ποινή, τιμωρία. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι φορολογούμενο τιμωρείται διπλά. Και δεν εκτελείται το πρόγραμμα και τελικά έρχεται η ανάκτηση δηλαδή των ποσών, το πρώτο μισό, και το άλλο μισό είναι η ποινή. Άρα η επιβάρυνση για τον φορολογούμενο είναι διπλή, είναι πολύ μεγαλύτερη. Έχετε αναλογιστεί μήπως υπάρχει διαφορετική λύση για το θέμα αυτό. Το ελεγκτικό συνέδριο έχει κάποιες προτάσεις. Μήπως θα έπρεπε να ανατραπεί τελικά αυτός ο κανόνας. Γιατί νομίζω ότι τελικά το αποτέλεσμα είναι ακόμη πιο επιβλαβές για τον, Ευρωπαϊκό, για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Και για το ενέκτηση του ελεγκτικού συνεδρίου θα ήθελα να πω ότι ναι είναι κωδικοποιημένη η ορολογία που χρησιμοποιείται. Η κυρία Γκρέσλε στην Ολομέλεια ε, κατεφέρθη κατά της ε, κρυπτογραφικής αυτής ε, μεθόδου που χρησιμοποιείται στην έκθεση. Αλλά νομίζω ότι μαζί με το μεγάλο εγχειρίδιο για τα δημοσιονομικά του ελεγκτικού συνεδρίου μπορούμε να παρακολουθήσουμε την έκθεση και κυρίως να καταλάβουμε ποια κράτη εννοείται. Αν και πιο καλό για μας φυσικά θα ήταν να μην είστε τόσο ε, συμβιλική στα όσα λέτε και να είναι πολύ πιο ξεκάθαρα λέτε τα σίκα σίκα. Εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει συζήτηση κύριε Σεμέτα, κύριε Επίτροπε, τα μέσα τα οποία παρουσιάσατε εσείς ως ανεκτό κίνδυνο σφάλματος, tolerable risk error, δεν μπορεί να είναι ανεκτό ποσοστό για το μέλλον. Και το λέω αυτό και να με ακούσει το ελεγκτικό συνέδριο, διότι πιστεύω ότι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί σωστά δεν επιτρέπεται ούτε καν να αυξάνει φυσικά τον κίνδυνο του, σφάλμακος, του σφάλματος, αλλά ούτε και να καθυστερεί τη του. Γιατί έτσι παραμένουν συστημικά προβλήματα, προβλήματα τα οποία έχουμε εντοπίσει ήδη. Χαίρομαι διότι το ελεγκτικό συνέδριο με τρόπο σχετικά ανοιχτό, με ανοιχτό πνεύμα, γιατί το είχαμε την ευκαιρία ως Επιτροπή του Ελέγχου του Προπολογισμού να επισκεφθούμε και το Λουξεμβούργο, αλλά και εδώ να συζητήσουμε με τους εκπροσώπους του ελεγκτικού συνεδρίου. Έχει λοιπόν μια ανοιχτή θεώρηση ως προς το θέμα αυτό της ερμηνείας και των αρχών που ακολουθεί. Πιστεύω ότι και εμείς ως βουλευτές ακολουθούμε την ίδια αρχή, ότι δηλαδή η ιδέα, η αρχή της, ε, του αποδεκτού κινδύνου σφάλματος είναι για μας απαράδεκτη. Την εξετάσουμε μάλλον με αρνητικό πνεύμα. Ευχαριστώ πολύ. Αν θέλετε να απαντήσετε κυρία μου παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή ε, για τα ευγενικά του λόγια και για τις παρατηρήσεις. σχετικά με το τι κάνουν τα περιφερειακά δικαστήρια και οι εθνικές ε, ελεγκτικές αρχές. Πρέπει να σας πω ότι σε γενικές γραμμές ε, το κοινό αίσθημα δεν είναι ε, προς την συνεργασία. Ο καθένας ε, ελέγχει, αυτό γίνεται στον ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον, ο καθένας ελέγχει από την πλευρά του. Τώρα η συνεργασία γίνεται μέσω επιτροπών στις οποίες, οι οποίες διέπονται από εθελοντική συνεργασία και εθελοντικές βάσεις πώς μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας. Η μεθοδολογία μας είναι γνωστή και τα κράτη-μέλη ε, τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα θα πρέπει ε, να δουν κατά κάποιο τρόπο ε, πώς μπορούν να βελτιώσουν το περιθώριο λάθος τους. Ίσως θα πρέπει να δουν τι κάνουμε κι εμείς κατά κάποιο τρόπο ο καθένας ε, έχει την δικιά του μέθοδο ε, σαν μια διαδικασία benchmark. Το ίδιο συμβαίνει και στον τομέα των ε, ταμείων συνοχής. Τώρα, όσον αφορά... But indeed, in cohesion we established the Όσον αφορά τώρα την ε, μορφή. Αυτή η συζήτηση θα λάβει χώρα αύριο. Το σημαντικό είναι να ε, χρησιμοποιήσει καλή σωστά τα ευρήματα ε, της, του, του οικονομικού ελέγχου. Και βεβαίως για μερικές περιπτώσεις όπως ας πούμε στις, στην περίπτωση των δημοσίων προμηθειών πρέπει κανείς να βλέπει τι γίνεται και στο, σε εθνικό επίπεδο και ενδεχομένως να προσφεύγει και στο ε, δικαστήριο. Τώρα γιατί οι συνάδελφοι της ε, Γεωργίας ε, δεν θεώρησαν κάτι τέτοιο απαραίτητο, μα γιατί οι δαπάνες όσον αφορά την Γεωργία μπορεί να είναι αντιφατικές, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέποντας, διαπιστώνουμε από τις επισκέψεις μας ότι και εδώ αν πρέπει να εκφέρω την δικιά μου άποψη είναι ότι ε, και τα κράτη-μέλη και η πλευρά των, ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, δεν αντιδρούν τόσο πολύ όσον αφορά τα ευρήματά μας. Σέβονται περισσότερο τα ευρήματα που έχουμε ακριβώς επειδή εμείς δεν έχουμε τριμερείς συναντήσεις ενδεχομένως παραμένουν κάποια ανοιχτά ζητήματα και προβλήματα. Πάντως το δείγμα μας, έστω και αν ε, μεθοδολογικά είναι σωστό, είναι μικρό ε, και επομένως δεν μπορούμε να, ε, είμαστε, να έχουμε πάντα το πιο αντικειμενικό και καλό αποτέλεσμα. Αλλά πάντως μην πυροβολείτε τον αγγελιοφόρο εάν δεν σας αρέσει το μήνυμα. Αυτό είναι σαφές. Ε, από τα υπόλοιπα που είπατε είναι πιο πολύ πολιτικές σκέψεις, τις οποίες θα πρέπει να κάνετε εσείς κυρίως. Τέλος, ε, η αναφορά στα κράτη τα οποία ε, ελέγξαμε, το πρόβλημα για μας είναι ότι είναι δύσκολο να πούμε ακριβώς ε, πού πήγαμε και τι κάναμε, ε, γιατί δεν κάνουμε ε, κάθε χρόνο τις ίδιες, τους ίδιους ελέγχους. Δεν αποφεύγουμε να δημοσιοποιήσουμε τα στοιχεία αυτά, γιατί εμείς δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο σχήμα. Ο Επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ. Τα περισσότερα ερωτήματα αφορούσαν το ελεκτικό συνέδριο, αλλά θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια όσον αφορά την ε, διαχείριση δηλώσεων. Ξέρετε ότι μας απασχόλησε το θέμα αυτό και ε, στο θέμα των ε, πολιετώ, του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και του δημοσιονομικού κανονισμού. Εγώ προσωπικά οποτεδήποτε επισκέπτομαι τα κράτη-μέλη, ε, θέλω να συναντώ εκπροσώπους του ελεγκτικού συνεδρίου των κρατών αυτών και ε, λέω πάντα ενδιαφέρομαι να μάθω τι κάνει, ε, ποια είναι η εργασία και τα αποτελέσματα στα οποία καταλήγει το ελεγκτικό ε, συνέδριο. Αλλά βεβαίως ε, θα πρέπει ε, να είναι ανεξάρτητες αρχές έτσι ώστε και ο έλεγχος να είναι ανεξάρτητος. Ταυτοχρόνως εμείς θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τις εθνικές δηλώσεις. Αυτή τη στιγμή τελειοποιούμε την εργασία σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές, δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν οι δηλώσεις αυτές να γίνονται έτσι ώστε να δώσουν θέμενη αξία στην εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι η παρούσα ποικιλομορφία και οι φυστάμενες διαφοροποιήσεις των δηλώσεων δεν επιτρέπουν την ορθή χρήση αυτών των δηλώσεων. που κάνουν τα κράτη-μέλη, τουλάχιστον ορισμένα κράτη-μέλη. Όσον αφορά το θέμα του επίπεδου ενοχής, ε, όσον αφορά ε, τα λάθη, πιστεύω ότι έχει ήδη λάβει χώρα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στην Επιτροπή σας εδώ και ε, ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε την ανταλλαγή απόψεων και τον διάλογο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμφωνήσουμε καταρχήν μεταξύ μας όσον αφορά ε, την ε, ε, αντίληψη που έχουμε για τον οικονομικό έλεγχο. Πρόκειται περισσότερο για μια αντίληψη διαχείρισης που θα μας επιτρέψει να έχουμε σημεία σύγκρισης και αναφοράς για, την, για, σε αιτήσια βάση. Και βεβαίως να έχουμε και ένα σημείο αναφοράς και σύγκρισης και για τα υπόλοιπα ποσά, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να έχουμε όσο γίνεται σαφέστερη εικόνα, να ξέρουμε πώς έχει η κατάσταση, ποια είναι η περούσα κατάσταση, πώς ήταν πριν, τι μπορούμε να βελτιώσουμε, τι βελτιώθηκε, έτσι ώστε να εξαγάγουμε κάποια γενικά χαρακτηριστικά του προγράμματος. Αυτή νομίζω ότι είναι η κεντρική ιδέα της αντίληψης ε, για το ανεκτό επίπεδο λαθών. Ε, κινδύνου, συγγνώμη για το 50-50 ο, κανένας, ο κανόνας του 50-50 ε, κατά την άποψή μου δεν είναι κυρωτικός για τα κράτη-μέλη. Εάν τα κράτη-μέλη δεν ε, ε, πάρουν τα χρήματα, τότε αυτός ο κανόνας του 50-50 αρχίζει να εφαρμόζεται. Όμως, δεν επιτρέπει στα κράτη-μέλη να σταματήσουν την διαδικασία. Αντιθέτως, ε, τους επιτρέπει να συνεχίσουν τη διαδικασία ανάκτησης. Στην ουσία δηλαδή πρόκειται για ε, επιπλέον κίνητρο. Uh, uh, Αυτά σε σχέση με τις ε, ερωτήσεις που έκανε ο εισηγητής. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκρέσλερ. Ε, Θα ήθελα και μια άλλη φορά να επισημάνω ότι βεβαίως είναι πολύ σημαντικά το όσα μας λέτε, ότι πληροφορίες μας δίνει το Ελεκτικό συνέδριο και δεν συμφωνώ σήμερα ότι μπορεί κανείς να παραπεμφθεί σε άλλα 4-5 διαφορετικά έγγραφα και να έχει επαρκή ενημέρωση. Όχι, σε αυτό δεν συμφωνώ. Και το θέμα επίσης είναι πόσα κονδύλια έχουν απορροφηθεί από το, το Ταμείο Συνοχής. Ο κύριος Καλτέρα μας είπε 30%, οι Financial Times λένε 10%, και ο επίτροπο επίση μα είπε 10%. Επομένως, ποια είναι τα σωστά νούμερα. Σε ποιο βαθμό γίνεται αυτή η διάθεση των κονδύλων. Για τελικά αυτό θέλουμε. Θέλουμε να διατεθούν όπως πρέπει τα κονδύλια στα κράτη-μέλη. Πάση περιπτώσει, τις πληροφορίες θα τι παίρνουμε πάντοτε από τον τρόπο, από την έκθεση σχετική με την εκτέλεση του προπολογισμού της κάθε χρονιάς. Και έτσι θα ήθελα να παρακαλέσω του εκπροσώπους του Ελληνικού Συνεδρίου να μας δίνουν πάντοτε πληροφορίες ανάλογα με αυτό που ζητούμε και να, μας, και τα όσα λένε κατά τρόπο πιο προσεκτικό. Για τη τελευταία ανάλυση εμάς υπηρετεί το ελεγκτικό συνέδριο. Εδώ, αυτό το έγγραφο που έχουμε με την συγκριτική εξέλιξη της δημοσιονομικής διαχείρισης, αυτό το έγγραφο με τα χρώματα, βλέπω ότι έλαβε χώρα συλλογική ψηφοφορία μέσα στο ελεγκτικό συνέδριο ε, για το αν θα περιληφθεί ή όχι το σχετικό έγγραφο μέσα στην ενημέρωσή μας. Το καταλαβαίνω αυτό και με λυπεί πολύ. Ναι, βεβαίως και είναι στιγμιές καταγραφές της κατάστασης τέτοιου είδου έγγραφα και βεβαίω θα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη ω μόνιμες καταστάσεις κλπ. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί κανείς πρέπει να κάνει την επιλογή αντί για μένα και να αποφασίσει να μην μου διαθέσει τη σχετική πληροφορία. Δεν είναι σωστό. Επιτρέψτε μου, δεν είναι fair. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πια πρέπει να συζητήσουμε εις βάθος ορισμένα θέματα και σε σχέση με το ελεγκτικό συνέδριο και ως προς το εάν και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν κάποιες πληροφορίες, εάν και πώς διατίθενται στο Κοινοβούλιο ορισμένες πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Καλιουλάιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως, αυτή τη στιγμή που το ελεγκτικό συνέδριο είδε ε, βελτίωση των, ε, της ε, ποιότητας ε, πληροφόρησης ε, όντως από τον, ε, την διαχειριστική αρχή μείωσε ε, τη, το, τις διαπιστώσεις ε, λάθους. Όμως υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία ε, κάποιες επικρίσεις λείπουν από το φετινό έγγραφο. Τώρα, τα αποτελέσματα δειγματοληπτικών ελέγχων αφορούν ε, κυρίως ε, στοιχεία τα οποία πήραμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχουμε κάνει επιπλέον ε, οικονομικό έλεγχο, αλλά βεβαίως μερικές φορές είναι καλύτερα να έχει κανείς ένα τεύχος πιο μεγάλο με 500 σελίδες παρά 2-3 από 200 ή 300 σελίδες σχετικά με τις επικρίσεις αυτές μπορώ να πω για το 2010 ότι εάν υπάρξουν πληροφορίες πολύ σημαντικές οι οποίες θα πρέπει να αναφερθούν στα εγκάρσια κεφάλαια τότε και για τις ομάδες πολιτικών ε, αυτό ε, θα πρέπει να αναφερθεί και το έχουμε καταγράψει και εγώ η ίδια αλλά και άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι ασχολούνται με τον τομέα της συνοχής. Θέλετε να προσθέσετε κάτι? Όχι. Ο κύριος Χατζημαρκάκης ε, όχι. Επομένως μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, σημείο 6 που αφορά τη συνέχεια στην άρνηση χορήγησης απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία ε, για το οικονομικό έτος 2008 και θα δώσω αμέσως το λόγο στη συνάδελφο Ματιού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα της άρνησης απαλλαγής το 2008, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η συζήτηση για την απαλλαγή για το 2009. Λυπούμε γι' αυτό, αλλά ε, με πάσα ειλικρίνεια θα σας λέω ότι και η συγγήτρια και ο σκιώδης η συγγήτρια πολύ θα ήθελα να έχει κλείσει αυτό το θέμα αλλά έχει τόσο πολύ καθυστερήσει και έχει μπει στα συρτάρια που τελικά θα καταλήξει σύριαλ. κύριος Μποφίλ, διευθυντής και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αλλά και υπάρχει, και υπάρχει εδώ και εκπρόσωπος του Ελεκτικού Συνεδρίου και τη επιτροπή και ελπίζω να ακούσουμε και την άποψή σας. Ο, ο κύριος Μαρίνη είναι εδώ δηλαδή και με, με μεγάλο ενδιαφέρον θα περιμένω την παρέμβασή σας. Ο κύριος Μποφίλ. Καταρχάς, θα θέλαμε να μάθουμε το εξή. Έχει σχέση με το ελεγκτικό συνέδριο δηλαδή το ερώτημα. Ε, να το πω αλλιώς, να το θέσω αλλιώς. Διαπιστώσαμε διάφορα ε, σφάλματα για ποσά καθόλου αμεληταία και μιλούμε για διορθώσεις οι οποίες εκτείνονται σε βάθος ετών και Ε, εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για το 2008 244.000 ε, για παράδειγμα ευρώ ε, για το 2008 αυτά δημοσιεύθηκαν τον Ιούλιο γιατί δεν έθεσε επιφύλαξη το ελεγκτικό συνέδριο και μιλούμε και για διορθώσεις για ένα εκατομμύριο ευρώ και πάνω πρόκειται για αποκατάσταση των πλεονασμάτων του 2007 που δεν έτυχαν αναγνώρισης ή είναι υπερβολική εκτίμηση για τα εισοδήματα. Πολύ τεχνικά είναι τα ερωτήματα που έχω να θέσω υπόψη του κυρίου Μποφίλ. Δεν θέλω να ε, χρονοτριβήσουμε γιατί είναι ήδη 6 και 5. Είναι πολύ τεχνικές οι ερωτήσεις και πολύ συγκεκριμένες. Και μάλιστα η λογιστική υπηρεσία του Κοινοβουλίου έθεσε υπόψη μου ε, τα θέματα αυτά. Θα σας τις υποβάλω γραπτό στις ερωτήσεις αυτές για να έχουμε και γραπτή απάντηση. Έτσι απλουστεύεται η διαδικασία και θα έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια. Μπορείτε ωστόσο τώρα να μας απαντήσετε για τις διορθώσεις. Για τι σημαίνουν, γιατί γίνονται το 2010 για τις προηγούμενες χρονιές. Και τέλος, ποια είναι η οικονομική κατάσταση της υπηρεσίας. Μπορείτε να μας την περιγράψετε. Πού βρίσκεται σε επίπεδο προϋπολογισμών. Στη σελίδα 8 διαβάζουμε ότι ε, το κεφάλαιο είναι μείον πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ στις 31 Δεκάτου του 2009. Ισχύει αυτό. Και γιατί η υπηρεσία δεν έχει τηρήσει αυτή την αρχή ε, της ε, ε τήρησης του προϋπολογισμού, τόσο ώστε να μην έχει αρνητικό πρόσημο. Και κάτι που μας ενδιαφέρει επίσης σήμερα είναι οι πιστώσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί για ιδιωτικές δαπάνες. Ο ανεξάρτητος εξωτερικός έλεγχος που έγινε για τις ιδιωτικές δαπάνες εκτιμά ότι το ύψος του είναι 42.800 λίρες. Διαφορετικά είναι τα στοιχεία που έχει υποβάλει η υπηρεσία. 19.000 περίπου λίρες. Ποιος είναι ο αντίκτυπος στον προπολογισμό και πώς ε, εξηγούνται αυτές οι διαφορές. Να, σας, ε, να σταματήσω από εδώ για να απαντήσετε. Καλώς. Να δώσουμε το λόγο αν θέλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι προφανώς. Θα ήθελα πρώτα να απαντήσει, λέει η κυρία Ματιώ, να απαντήσει ο κύριος Μπόμφη. ε, ε γιατί ε, έθεσα συγκεκριμένα ερωτήματα στον κύριο Μπόμφη, ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο και μετά στην Κομισιόν και μετά στους συναδέλφους, αν συμφωνείτε κι εσείς. Εξαιρετικά κύριε Πρόεδρε, εξαιρετικά μέλη του Κοινοβουλίου. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Τη Ευρωπαϊκή Σχολή Αστυνομίας, του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Αστυνομία. Ε, ευχαριστώ πολύ που μας έχετε δεχθεί εδώ και ελπίζω ότι θα μπορέσω να σα δώσω συγκεκριμένε απαντήσεις σε ερωτήσεις. Όπως γνωρίζετε, ανέλαβα τα καθήκοντα στις, του Διευθυντού στι 16 Φεβρουαρίου εφέτο. Η κληρονομιά που πήρα, παρέλαβα, είναι μια περίπλοκη πρόκληση. Διαχείριση σημαίνει και μεγάλη ε, στράτευση, πολλή δουλειά, αλλά και επαγγελματικότητα, επαγγελματισμό πλευρά όχι μόνο δικής μου, αλλά όλου του προσωπικού της σχολής. Με λύπη ενημερωθήκαμε ότι αποφάσισαμε εδώ στην απαλλαγή το Κοινοβούλιο για το έτος 2008. Ε, αποδέχομαι φυσικά την ε, απόφαση, αντιλαμβάνομαι τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν, πλην όμως θα ήθελα να πω ότι ο τρέχον διευθυντή, ο τωρινό διευθυντή, στα καθήκοντα που έχει αναλάβει, έκανε ό,τι μπορούσε με βάση τους δημοσιονομικού κανονισμού και κανόνες να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα απέτρεπε το Κοινοβούλιο από το να χορηγήσει απαλλαγή. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σα δώσω μια σύντομη επισκόπηση εν προκειμένου και μια σύντομη απάντηση στα όσα είπε η κυρία Ματσιού. Ω ανταπόκριση στο νόμιμο ε, θεμητή προσδοκία μάλλον του Κοινοβουλίου. Πεβάλαμε, υποβάλαμε τις προτάσεις μας, οι οποίες είχαν λάβει την έγκριση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του εσωτερικού δημοσιονομικού λόγου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την επιβεβαίωση από το Διοικητικό μας Συμβούλιο που συνομενόταν. Ένα δεκαετές λοιπόν πρόγραμμα δράσεως, το οποίο υπέβαλα ακριβώς για αυτό το λόγο, για να εγκριθεί. Ένα σχέδιο το οποίο στοχεύει να παρακολουθήσει την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Σχολής Αστυνομίας και είναι παρεξήγηση και παρερμηνία της λειτουργίας της σχολής, ότι δηλαδή θα παραμείνει μόνο σε λειτουργία για τα τέσσερα χρόνια της θητείας του ευθυντή. Το πολιετές πρόγραμμα δράσης υπευλήθη εγκαίρως στις 6 Ιουνίου του 2010 και μάλιστα πριν από την προθεσμία, την καταληκτική προθεσμία που οριστεί, μετά την κατάθεση του πολιετούς προγράμματος δράσεως. Κατέθεσα και δύο εκθέσεις προόδου ως προς την υλοποίηση του σχεδίου προς το Κοινοβούλιο. Στη διάθεσή σας. Η εσωτερική, ο εσωτερικός δημοσιονομικός έλεγχος παρακολούθησε την εφαρμογή και αιτιολόγησε το περιεχόμενο, δικαιολόγησε μόνο το περιεχόμενο της δεύτερης έκθεσης, λέγοντας ότι αυτά που σας αναφέρω ήταν ορθά. Ο, επίσης, δεύτερον, ο εσωτερικός έλεγχος λέει ότι έχουν προχωρούν ικανοποιητικά οι διαδικασίες της υλοποίησης. Και φαντάζομαι ότι η Επιτροπή σας θα μπορεί να επαληθεύσει τα στοιχεία αυτά αν ρωτήσει τους δημοσιονομικούς ελέγκτες. Υπευλήθη λοιπόν στρατηγική, ε, Επιτροπή Στρατηγικής στις 25 Νοεμβρίου, στη ΣΥΠΟΛ δηλαδή η σχετική έκθεση και τώρα ε, μέχρι τις 8-9 Δεκεμβρίου θα έχει φτάσει στο Διοικητικό Συμβούλιο που θα την εξετάσει τότε η πρόοδος στους τελευταίους εννέα μήνες είναι απτή και θα ήθελα να δηλώσω ότι είναι νόμιμη, λειτουργική και νομότυπη η δράση της σχολής. Οι παρατηρήσεις που έχουν να κάνουν με κατάχρηση στοιχείων, ε, όπως ανέφερε η κυρία Ματσιέ, επαληθεύτηκαν από την εξωτερική ε, εταιρεία δημοσιονομικού ελέγχου ένα ποσό 42.800 λιρών που ήταν αντικείμενο κατάχρησης, ένα, ένα ποσοστό σχετικά χαμηλό έχει αποδοθεί, έχει επιστραφεί και σε αυτό συμφωνούμε με την ε, διαπίστωση του ελεγκτικού συνεδρίου, το ποσοστό δηλαδή ανάκτηση είναι πολύ χαμηλό και ότι δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί το πραγματικό πεδίο της κατάχρησης. Διότι δεν είναι επαρκής η τεκμηρίωση που άφησε πίσω της η προηγούμενη διοίκηση και διαχείριση της σχολής. Οι κύριες απώλειες εντοπίζονται στην αγορά επίπλωσης. 14.388 ε, ευρώ που πωλήθηκε κατόπιν συστάσεως της, ε, ε, του ελεκτικού συνεδρίου με έσοδο που έφερε αυτή η πώληση 500, 500 λίρες. Δεν θα ήθελα να σας εξηγήσω λίγο περισσότερο την ε, κατάσταση, γιατί δεν καταλάβετε. Η κατάσταση αυτή σχετική με την αγορά των επιπλώσει είναι του 2007, όχι του 2008. Οι διαδικασίε, λοιπόν οδήγησαν, οι διαδικασίε αυτέ του 2007 έδωσαν οδήγησαν το κοινοβούλιο στο να δώσει απαλλαγή, ενώ ήταν γνώση αυτή τη αγορά επίπλωση. Εφέτος όμως φαίνεται ότι ε, κατηγορούμε πως αρνήθηκα την ε, ε, απόδοση ποσών σε 13 διαφορετικές περιπτώσεις, ατομικές επιστροφές. Ωστόσο, εγώ όταν ανέλαβα τα καθηκοντά μου βρήκα στον προπολογισμό του 2008 70 περιπτώσεις προβληματικές. Τις διερεύνησα όλες, τις επέλυσα όλες και ο το προπολογισμό του 2008 τώρα είναι καθαρός. Δεν υπάρχει ερωτηματικό εκκρεμότητα δηλαδή για τον προπολογισμό του 2008. Άλλο ένα πολύ σημαντικό θέμα που ήθελα να επισημάνω είναι ότι από ό,τι εγώ γνωρίζω από αυτή την εξωτερική ε, ελεγκτική δραστηριότητα, τον εξωτερικό δημοσιονομικό έλεγχο, αποδεικνύεται ότι δεν προκύπτουν ποινικέ ευθύνε. Δεν έχει κινηθεί δηλαδή ποινική διαδικασία. Γι' αυτό λοιπόν καλό το Κοινοβούλιο να ζητήσει από την Όλαφ τη σχετική έκθεση και να ρωτήσει την Όλαφ γιατί δεν εκκίνησε ποινική διαδικασία για κατάχρηση κατά του προηγούμενου διευθυντή. Για κατάχρηση, για διαφθορά, για οικονομικό έγκλημα. Όχι, όχι, δεν το έπραξαν. Διαφορά Ποιος είναι ο λόγος που εμφανίζεται αυτή η διαφορά. Η σχολή δεν ήταν σε θέση και σε αυτό δεν μπορώ να δώσω απάντηση γιατί δηλαδή συνέβη, γιατί δεν είχα εγώ να λάβει κάτι κοντά ακόμα, δεν ήταν σε θέση να δώσει ε, εκτεταμένη έκθεση, συνολική έκθεση εμείς τώρα όμως δώσαμε κάθε δυνατότητα πρόσβαση στους δημοσιονομικούς, δημοσιονομικούς ελεγκτές, συνεργαστήκαμε στενά μαζί τους, προκειμένου να ευκολύνουμε να καταλήξουν στην αλήθεια. Η τωρινή ηγεσία δεν έχει κανένα συμφέρον να συγκαλύψει ή οδήποτε περιστατικό κατάχρησης ή κακοδιαχείρισης από το παρελθόν. Έχει κάθε συμφέρον να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου και θέλουμε να στηρίξουμε το μελλοντικό κολέγιο αστυνομία σε μια ισχυρή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η διόρθωση λοιπόν των σφαλμάτων ε, που αναφέρονται στους τελικούς λογαριασμούς του 2009 στις αρχές Μαρτίου μεταξύ 8 και 11 Μαρτίου έγινε ο προσδιορισμός της δημοσιονομικής ε, δήλωσης της ε, ε, σχολή στις 12 του μηνό Μαρτίου πάλι, την επομένη δηλαδή έκανα συνάντηση με τους εκπροσώπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου που μου, εν, ε, που με ενημέρωσαν ότι δεν ήταν η προσωρινή αυτή δήλωση αξιόπιστη και οι λοιποί λογαριασμοί. Μου εξηγήθηκαν κάποιες άλλες δυσκολίες που είχα να αντιμετωπίσω και γι' αυτό λόγο έθεσα σε κίνηση μια ειδική ε, εργασία, λειτουργία εκαθάρισης όλων των τεχνικών, δηλαδή λογιστικών σφαλμάτων στους λογαριασμούς. Και έτσι εκεί αποκαλύφθηκαν πολλά μεγάλα σφάλματα διοικητικού χαρακτήρα, αυστηρά διοικητικού χαρακτήρα και χωρίς να τολμώ να αστιευτώ θα το πράξω στο παρελθόν το 2 συν 2 σήμαινε 6 στους λογαριασμούς της σχολής. Τέτοια σοβαρά σφάλματα δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει εντοπίσαμε πολλά τεχνικά σφάλματα στους λογαριασμούς ως τον προπολογισμό, στους λογαριασμούς μας. Ενημερώσαμε για τα σφάλματα αυτά, δώσαμε ιδέες για ε, λύση των προβλημάτων αυτών στην Επιτροπή, στην Γενική Διεθνή των Προπολογισμών και διαβεβαιώσαμε για απόλυτη ε, διαφάνεια ενάντια και του ελεγκτικού συνεδρίου. Το ελεγκτικό συνεδρίο λοιπόν ξαναήρθε. Ε, τέλη Ιουνίου μέχρι τις 2 Ιουλίου ήταν στην ε, σχολή μας ολοκλήρωσε τη δήλωσή του και με χαρά μπορώ να σας πω ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της ΣΥΠΟΛ όπου έγιναν έγινε δεκτός ο, ο, ο ισολογισμός μας από το Ελεκτικό συνέδριο χωρίς καμία παρατήρηση. Αυτό καταγράφεται στην έκθεση. Σημειώνει δηλαδή το Ελεκτικό συνέδριο όλες τις διορθώσεις τις οποίες ε, ε αιτιολογούσαν τα ε, σχετικά έγγραφα, η σχετική τεκμηρίωση αλλά είναι αυτά διορθώσεις που δεν έχουν να κάνουν με τον προϋπολογισμό. Ε, βέβαια, ο συλλογισμό δηλαδή αποτελεί αντικατοπτρισμό του προπολογισμού. και ως εκ τούτου θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικές εφαρμογές στον προϋπολογισμό αυτών των διορθώσεων. Κυρίε και κύριοι, πιστεύω ότι έδωσα απαντήσεις στις ε, ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ματιέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα το ελεγκτικό συνέδριο να πάρει το λόγο και να μας απαντήσει στο εξής. Γιατί ε, δεν έθεσε επιφύλαξη για το 2008, γιατί το αποθεματικό ήταν αρκετά σημαντικό βάσει του ύψους προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Μπορεί να μας εξηγήσει, να μας απαντήσει το ελεγκτικό συνέδριο σε αυτό το ερώτημα. Απάντηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ελεγκτικό συνέδριο δεν εξέφρασε επιφύλαξη αυτή καθ' αυτή ή αν θέλετε ο σωστός όρος είναι δεν παρουσίασε χαρακτηρισμό ε, των λογαριασμών για το 2008. Σας υπενθυμίζω Ε, εξέδωσε αυτό το οποίο ονομάζουμε «An emphasis on matter» ε, λόγω συγκεκριμένων προβλημάτων που προέκυψαν ε, ως προς την ποιότητα των λογαριασμών αυτών. Γιατί δεν εκφράσαμε επιφύλαξη. Δεν ήμασταν σε θέση. Η απάντηση είναι απλή. Και είναι κάτι που είπε και ο ίδιος ο κύριος Μπάνφι. Δεν είχαμε στοιχεία στα χέρια μας για να είμαστε σε θέση να δούμε ποια είναι η ποσότητα των σφαλμάτων αυτών, πόσα πολλά είναι και πού υπάρχουν, ε, σε, σε ποιους τομείς. Και γι' αυτό εκφράσαμε αυτό το emphasis of matter. φαινόταν ότι τα σφάλματα περιορίζονταν σε συγκεκριμένους τομείς. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχαμε ε, στο εσωτερικό του ελεκτικού συνεδρίου, αποφασίσαμε αντί να τα χαρακτηρίσουμε, γιατί χαρακτηρισμός γίνεται μόνο όταν έχουμε ακριβή ποσοτικοποίηση των σφαλμάτων, προτιμήσαμε λοιπόν αντί να κάνουμε κάτι τέτοιο, να επιλέξουμε αυτή την άγουσα που σας παρουσίασα, το έμφαση σωμάτερ, ακριβώς για να εφιστήσουμε την προσοχή στο θέμα. Ε, και όπως το είπε και ο κύριος Μπάνφη, στη συνέχεια, ε, το 2007, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία αυτή ανέλαβε δράση και ε, αποκατέστησε, αν θέλετε, τους λογαριασμούς αυτούς, έγιναν διάφορες προσαρμογές, πολύ ενεργητική ήταν η καινούργια διοίκηση και έτσι, σήμερα απεικονίζεται καλύτερα η οικονομική πραγματικότητα της ΕΠΟΛ, της υπηρεσίας αυτής. Ε, πολλά στοιχεία είναι παρουσιάσιμα και έχουν γίνει και ε, προσαρμογές, ρυθμίσεις κάποιων σφαλμάτων στις εκτιμήσεις, τις ορευτικές. Και άλλωστε ως προς αυτό οι προηγούμενες εκτιμήσεις δεν ήταν καθόλου ακριβείς. Όλα αυτά έχουν επανεξεταστεί ε, κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης πραγματικά κομάντο ε, που έχει εκτελεχθεί από τότε που ανέλαβε ο κύριος Μπάνφι τα ε, δράση. Η κυρία Ματιέ, συγγνώμη κυρία, αλλά εγώ σας ρώτησα για το 2008 και όχι για το 2009 που έχει αναλάβει καθήκοντα ο κύριος Μπάνφι. Ε, το 2007 υπήρχαν ήδη προβλήματα. Και εσείς προσωπικά είσαστε αρμόδιος, έτσι δεν είναι. Η συγητή της ε, προηγούμενης χρονιάς είχα, είχε ήδη προτείνει άρνηση. Και ε, παραλίγο να εγκριθεί για τέσσερις ψήφους. Όλα αυτά που μας λέτε, σε ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι σαν να μας κοροϊδεύετε. τι θα, απαντήσετε. Γιατί αυτό ακριβώς κάνετε, ε, έτσι το χαρακτηρίζω. Ε, θα έλεγα ότι είναι γκροτέσκο να μην έχετε επιφύλαξη για τους λογαριασμούς για το 2008 και να λέτε ότι δεν είχατε στοιχεία. Ζητώ συγγνώμη, αλλά να σας υπενθυμίσω ότι ε, το 2007 διακόπτει πάλι η κυρία Ματιέ. Κοιτάξτε, υπάρχουν διορθώσει για 2005, 6, 7 αλλά και 8 για 300.000 ευρώ. Και δεν εκφράσατε επιφύλαξη στο ελεκτικό συνέδριο για καμία από αυτέ τι χρονιές. Πώς χαρακτηρίζετε αυτή τη δράση σας. Δεν μιλώ για τον κύριο Μπάμφη. Δεν έχει καμία σχέση. Ε, μιλώ για τον κύριο Γκόρενσον και μα είπατε ότι οι λογαριασμοί ήταν μια χαρά και ότι δεν είχε λόγο το ελεγκτικό συνέδριο να εκφράσει επιφυλάξει. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω κάνει λογιστική, δεν έχω σπουδάσει λογιστικά, αλλά ε, δεν χρειάζεται κανείς να είναι ορκωτός ελεγκτής για να καταλάβει αυτά τα νούμερα και αυτή την κατάσταση. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή εμπέζεται τη δική μας Επιτροπή. Να σας υπενθυμίσω, λέει ο μιλητής, ότι όπως, είπε, όπως το υπενθύμισε και ο κύριος Μπάνφη, κάθε χρονιά το ελεκτικό συνέδριο εξέφρασε επιφύλαξη για ε, τους λογαριασμούς της ΕΠΟΛ κάθε χρονιά. Το 2007, το 2008, ε, το 2006, ε, αν δεν απατώμε, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, έχουμε επισημάνει τα σφάλματα αυτά. Το 2008 μόνο, αντί για επιφύλαξη, έχοντας συζητήσει στο εσωτερικό ε, του οργάνου μας ε, τα διάφορα επιχειρήματα που πρόβαλε η υπηρεσία, προτιμήσαμε να ε, συνοδεύσουμε τη γνωμοδότησή μας, αν θέλετε, όχι με το χαρακτηρισμό της επιφύλαξης, αλλά με το χαρακτηρισμό του emphasis on matter. Κάθε χρονιά έχουμε φυστήσει την προσοχή σε συγκεκριμένα προβλήματα που απεικονίζονται στους λογαριασμούς, των ισολογισμό, αν θέλετε, της ΕΠΟΛ. Τώρα, έχει αναδιοργανωθεί η υπηρεσία αυτή το 2009 έχει ενισχύσει ε, το οπλοστάσιο της. Η κυρία Ματιέ διακόπτει πάλι. Συγγνώμη, δεν είμαστε στο 2009. Μην επανέρχεστε σε αυτό. Ε, ο καθένας εύχεται η υπηρεσία αυτή να λειτουργήσει σωστά. Εγώ δεν ε, έχω τίποτα εναντίον της ΕΠΟΛΟΥ, ούτε εναντίον του κυρίου Μπανφή. Ε, μιλήστε για το 2008 παρακαλώ. Απάντηση. Ναι, είχαμε αυτό που σας λέω, το χαρακτηρισμό έμφαση ο μάτερ για να εφιστήσουμε την προσοχή σε μια σειρά προβλημάτων. Τώρα, το ελεγκτικό συνέδριο θεώρησε ότι όντω είναι καλύτερα να έχουμε έμφαση στο και όχι επιφύλαξη το προτιμήσαμε αυτό όντω. Ε, μέσα στο εσωτερικό του οργάνου μας, του θεσμικού οργάνου. Είναι θέμα εκτίμησης αν θέλετε. Ε, αξιολόγησης των στοιχείων που είχαμε επιτάπητος. Διάφορα στοιχεία των λογαριασμών της ΣΕΠΟΛ αποκαταστάθηκαν, σκιές παρέμεναν ε, σε ορισμένα από αυτά τα βάλαμε λοιπόν στη ζυγαριά και θεωρήσαμε ότι είναι επαρκή αυτός ο χαρακτηρισμός του έμφαση of matter. Είναι θέμα εκτίμησης, είναι θέμα άποψη. Η κυρία Ματιέ. Θα ήθελα να θέσω ρωτήσει στον ε, πρόεδρο του Governing Bond, ε, του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε του λογαριασμού τη ΕΠΟΛ. Μπορείτε να μα εξηγήσετε πώ έγινε κάτι τέτοιο, πώ πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο η θέση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνη, ομόφωνος ενέκριναν τους λογαριασμούς. Ε, βασίστηκαν σε εξωτερικό ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος είπε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξαιρετική ισχύ συγκριτικά με το Διευθυντή. Πώς το ε, αξιολόγησαν αυτό Αντίθετα με τις άλλες υπηρεσίες, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει το Διευθυντή όχι κατόπιν πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποιο ήταν το κριτήριο λοιπόν για να επιλεγεί ο συγκεκριμένος Διευθυντής και γιατί ε, δεν υπήρξε αντίδραση ε, στους κόλπους του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς τις δυσκολίες που ε, είχαν προκύψει όλα αυτά τα χρόνια και τις οποίες παρουσιάσαμε τόσο εκτενώς. Παρακαλώ, εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει το λόγο. Ναι, ναι. Ε, κοιτάξτε, εμείς έχουμε ήδη απαντήσει κατά τη διάρκεια της Βελγικής Προεδρίας ε, στα ερωτήματα αυτά. Έχουμε, έχουμε βάλει και ένα πίνακα ε, βαθμολόγηση, ένα scoreboard. Ε, νομίζω ότι έχουμε ήδη απαντήσει, δεν υπάρχει λόγος να τα ξαναλέμε. Δεν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, ευχαριστώ. Όχι, ευχαριστώ. Ε, ε, νομίζω ότι απάντησα σε όλα. Ωραία λέει η κυρία Ματιά, από το καλό στο καλύτερο. Επομένως, ε, πότε ξεκινήσατε να δραστηριοποιήσετε στα πλαίσια του ΣΕΠΟΛ και πότε αναλάβατε τη λειτουργία. Ε, πότε ξεκίνησα τη θέση μου στο ΣΕΠΟΛ. Εγώ εργάστηκα εκεί και εργάζομαι κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Βελγικής Προεδρίας ε, στόχος μας ε, είναι να ε, έχουμε ένα τελικό ισορροπημένο αποτέλεσμα. Βεβαίως βρίσκεται ακόμα αυτή η δοκιμασία σε δοκιμαστικό επίπεδο. Και το όνομά σας κύριε? Jean-Marie Van Bronte. Κυρία Ματιέ, γιατί λοιπόν όταν κλικάρουμε πάνω στο site ε, του ΣΕΠΟΛ δεν βλέπουμε το όνομά σας αλλά το όνομα του κυρίου Μιλερτ Επίσης, όταν, ε, όταν λαμβάνουμε κάποια υπομνήματα ε, από την πλευρά του ΣΕΠΟΛ, ε, υπογράφει ο κύριος Μίλερτ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει εμπλακεί σε διάφορες περιπτώσεις κατάχρησης και η Υπουργό Δικαιοσύνης του Βελγίου θέλησε να τον αποσύρει και ότι επίσης τα συνδικάτα της αστυνομίας δεν δεν ήθελαν, μάλλον σκανδαλίστηκαν από την ε, απόφαση να πάρει τη θέση αυτή. Απάντηση. Ο κύριος ε, Μίλλερτ, από ό,τι ξέρω, ε, δεν ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, εξεφράστη ενώπιον του Βελγικού Κοινοβουλίου μίλησε για όλα τα ζητήματα. Πριν από τέσσερα χρόνια ξεκίνησε όντως μία ε, έρευνα ε, για τον κύριο Μίλλερ, τον εν λόγω κύριο Μίλλερ, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Επομένως δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση, δεν έχει αποδειχθεί κάτι Τώρα, ε, το συνδικάτο, υπάρχει ένα συνδικάτο της αστυνομίας, είναι ένα αναγνωρισμένο συνδικάτο το οποίο ανακοίνησε ε, το θέμα, αλλά δεν νομίζω ότι εκεί έγκυται η ουσία ε, της σημερινής συζήτησης αφορά τον κύριο Μιλάρτα. Κοιτάξτε, εγώ λέει η κυρία Ματιό, δεν έχω κανένα λόγο να είμαι κατά του κυρίου Μίλερτ. Απλώς εγώ διαβάζω, ας πούμε, δημοσιεύσει του τύπου σε Πολ δύο τελίτσες, η υπουργό Δικαιοσύνης ε, ε, αποσύρει τον κύριο Μίλλερτ κτλ. Εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με όλα αυτά, ο κύριο Μίλλερτ δεν έχει κανένα λόγο ε, να, έχει τη θέση αυτή στο ΣΕΠΟΛ. Από την άλλη πλευρά, εάν κλικάρουμε πάνω στον ιστότοπο του κύριου Μίλλερ, του, του ΣΕΠΟΛ, συγγνώμη, βλέπουμε τον κύριο Μίλλερτ. Και από την άλλη πλευρά, εγώ τον έχω δει τον κύριο Μίλλερτ. Είναι μια χαρά άνθρωπο, ευγενέστατο και συμπαθητικό, τον έχω δεχτεί και στο γραφείο μου. Από την άλλη πλευρά δεν έρχεται ο κύριο Μίλλερ, το οποίο εμφανίζεται στα χαρτιά. Έρχεστε εσεί. Φαίνεται ότι δεν έχετε καμία απολύτω διάθεση να απαντήσετε στι ε, ερωτήσει σα. Από την άλλη πλευρά δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Εμένα στο γραφείο μου ήρθε ο κύριο Μίλλερ. Από την άλλη μεριά διαβάζω ότι η Υπουργό Δικαιοσύνη τον καθαίρεσε από την ε, θέση του. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται στο Βέλγιο. Με ενδιαφέρει ότι όλη αυτή η ιστορία κάπου μυρίζει και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να δώσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή και το, το, και το ε, ελεγκτικό συνέδριο απαλλαγή. Και εν πάση περιπτώσει δεν δεχόμαστε για μια υπηρεσία η οποία υποτίθεται ε, ότι αποτελεί το φυτόριο για του ε, αξιωματούχου τη Ευρωπαϊκή Αστυνομίας. Αυτό που θα θέλαμε είναι περισσότερη διαφάνεια σε αυτήν την Ακαδημία και θα θέλαμε τα ονόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να αναφέρονται σαφώ στον ιστότοπο τη υπηρεσία. Το ζήτησαν και οι συνάδελφοι, το ζητήσαμε 36 βουλευτέ τη ολομέλεια, το ζήτησαν στην Ολομέλεια και όταν ρώτησα τον κύριο Μπάμφη γιατί δεν αναφέρονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο, στη σελίδα του, της Ακαδημίας μας, ε, η, μας απήντησε ότι ε, δεν θέλησαν, αρνήθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να δημοσιευτούν τα ονόματά τους. Ρωτώ λοιπόν γιατί δεν το θέλετε. Thank Ευχαριστώ Πρόεδρε και επιτρέψτε μου να διευκρινίσω εγώ την κατάσταση. Και γιατί απαντάτε εσείς και όχι ο εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί απαντάτε εσείς. Εσείς μιλάτε εξ ονόματο του διπλανού σα. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε, μου ζητήθηκε, μου ζήτησε να απαντήσω εγώ. Ναι. Μπορώ. Ναι, ευχαριστώ. Δεν θέλω να καταστροφέ. ότι δεν είναι υπάλληλο τη ΣΥΠΟΛ. Ο κύριο αυτό είναι διαχειριστή σχεδίου, project manager, που έχει ορίσει η Βελγική Προεδρία. Κανείς, κανένα σώμα, όργανο της ΣΥΠΟΛ δεν, το έχει, δεν τον έχει προσλάβει ή διορίσει. Αυτό πρέπει να καταστεί απολύτως σαφέ κατάλογο του διοικητικού, των ονοματών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απάντησή μου είναι ακριβώς η προσεχής. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε την δυνατότητα αυτή και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ούτε στη Europol, ούτε στη Frontex, ούτε σε κανένα άλλο διοικητικό συμβούλιο υπάρχει θέμα δημοσίευση των ονομάτων των μελών. Υπάρχει ζήτημα, υπάρχει κάποια μέρη ασφαλείας όταν καταψήφισαν παραδείγματι τη δημοσίευση των ονομάτων του στα μέλη αυτού διοικητικού συμβουλίου, το πράττουν διότι κάποια εξ αυτών είχαν στο παρελθόν ε, δραστηριοποιηθεί σε δραστηριότητες κατά της τρομοκρατίας ή άλλες δραστηριότητες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την προσωπική τους ασφάλεια και αυτό δεν είναι δική μου γνώμη, είναι γνώμη των ιδίων των μελών. Πρόεδρος, ε, είναι ήδη 18 και 35. Έχουμε όμως και τρεις βουλευτές που θέλουν να θέσουν ερωτήματα. Φιέλ, Γκρέσλερ και Γκέγερ εάν συμφωνεί η συνάδελφος Ματιέ, ε, να πάρουν το λόγο οι συνάδελφοι, να θέσουν τα ερωτήματα που επιθυμούν. Ωραία. Ναι, Πρόεδρε. Πολλά υπόθηκαν ήδη. Πολύ στο μόνο θέλω να προσθέσω το εξή. Ότι όντω το Κοινοβούλιο είχε προσωπικά είχε δώσει την απαλλαγή με πολύ μικρό περιθώριο όμως δεν ξέρω πώς έγινε Είχε αρνηθεί μάλλον την απαλλαγή, αλλά με πολύ μικρό περιθώριο. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί συνέβη αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει συμβεί και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να έχουμε τώρα πράγματι μια σαφή εικόνα της κατάστασης. Ποιο είναι υπεύθυνο γιατί μέσα στη διοίκηση αυτή τη σχολή, εν πάση τη Ακαδημία. Απαιτείται κάτι τέτοιο. Και ναι, έχει προχωρήσει η ώρα, Πρόεδρε, και ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε διεξοδικά, αλλά είναι απαραίτητο να μα δοθεί ο χρόνο να συζητήσουμε διεξοδικά το θέμα αυτό και πρέπει να είναι παρόν και το Διοικητικό Συμβούλιο και να αναλάβει τι ευθύνε του, εν πάση περιπτώσει. Γκρέσλε. Η κυρία Χολμάιερ. Πρόεδρε. Κυρία Ματσιέ, Πρόεδρε, και σε αυτό συμφωνούμε. Ε, αγωνίστε πάνω απ' όλα να μην δοθεί η εντύπωση ότι η ανώτατη αυτή σχολή ε, αστυνομίας αποτελεί καταφύγιο όποιου θέλει να παραμείνει σε ατιμορρησία τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να το συστήσουμε το θέμα αυτό. Η συζήτηση δεν μπορεί να κλείσει σήμερα πολλά από τα ερωτήματα που την απασχολούν έχουν μείνει αναπάντητα ή έλαβαν πολύ ε, περιορισμένη απάντηση. Δεν είναι ικανοποιητική απάντηση που δόθηκε σε αυτά. Και γι' αυτό λοιπόν όταν έχουμε ζήτημα κατάχρησης, όταν κάποιος διώκεται για κατάχρηση, θα πρέπει να δοθούν οι απαντήσεις ιδιαίτερα από τις αρχές του κράτους που έχει προβεί στα σχετικά μέτρα. Είναι πολύ δυσάρεστη η θέση της συγχυτρίας. Είμαι βέβαιη ότι έχει μπροστά της μια πολύ δύσκολη έκθεση και γι' αυτό παρακαλώ να δώσουμε ένα περιθώριο και σύντομα να επανέλθουμε θα μας την ημερήσια διάταξη για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα, να δούμε εκπροσώπους της Ακαδημίας, να δούμε ανθρώπους από την Επιτροπή που να είναι προετοιμασμένοι να δώσουν απαντήσεις στο θέμα αυτό, γιατί είναι πραγματικά επώδυνη αυτή η κατάσταση που ζούμε. Και σε τελευταία ανάλυση και το ελεγκτικό συνέδριο ε, για την υπόθεση αυτή σήμερα δεν είπε και τίποτα. Γκάιερ. Εγώ έχω μια διαφορετική αντίληψη της κατάστασης. Άκουσα την έκθεση του κυρίου Μπάνφη, ο οποίος δίνει απαντήσεις σε αρκετές από τις ερωτήσεις μου. Δεν βλέπω γιατί έχει τέτοια αντίληψη η εισηγήτρια, 90.000 ευρώ, εκεί όπου ο κύριος Μπάνφη μιλάει για 80.000 ευρώ. Πού βρίσκεται η διαφορά, γιατί μιλάμε για διαφορετικά νούμερα. Πρώτον. Δεύτερον. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δεν καταλαβαίνω πού πάει αυτή η συζήτηση. Εγώ θέλω βεβαίω να διευκρινιστεί όλη η κατάσταση σχετική με τη ΣΕΠΟΛ, με την Ακαδημία, η προηγούμενη ηγεσία. Πώ είναι δυνατόν τώρα σε μια προφορική μου ερώτηση, κυρία Βάλστρομ, ερώτηση την οποία είχα διατυπώσει προκειμένου να αντιληφθώ τι, ίδιους, τι είδους επιπτώσεις ε, προκύπτουν για την Επιτροπή. Στι περάσματα καταλήγει η Επιτροπή από αυτήν την κατάσταση. Και μου απαντάει η κυρία Βάστρο μου ότι βεβαίω ο Διευθυντής έχει να αναλάβει τι σχετικέ ε, επιπτώσεις. Ο Διευθυντής όμω του, ε, περίοδου μέχρι το 2008 δεν είναι πια στη θέση αυτή, άρα τι είδου επιπτώσει θα αναλάβει. Το ΔΕ Διοικητικό Συμβούλιο, λέει, επίση θα πρέπει να αναλάβει τι σχετικέ ε, ε Μα δεν είναι σε τελευταία ανάλυση κάποια συνομωτική ομάδα του Διοικητικού Συμβούλου έχει έρθει εδώ στο Κοινοβούλιο, έχει, δώσει, έχει αποδώσει λογαριασμού, ξέρουμε αν υπάρχει και αν δεν υπάρχει σε ΣΕΠΟΛ και πώ λειτουργεί. Και πρέπει ασφαλώ η διοίκηση να λάβει στα σοβαρά υπόψη το Κοινοβούλιο και τις ευθύνε του. Δεν μπορεί να, δεχθούμε να μας ε, βάλουν στο παιχνιδάκι Κομισιόν και Διοικητικό Συμβούλιο. Η ΜΕΝ Κομισιόν να μας λέει φταίει το Διοικητικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο να μας λέει τις ευθύνες φέρει η Κομισιόν. Δεν γίνεται αυτό. Φτάνει πια. Και επιπλέον, πείτε μας παρακαλώ Πού βρίσκεται η εντολή για την απαλλαγή 2008. Ποιο την έχει, γιατί εμεί είμαστε διατεθειμένοι να το διαπραγματευτούμε το θέμα αυτό. Αλλά υπάρχει εισηγητή για την απαλλαγή τη ΕΠΟΛ και των λοιπών υπηρεσιών του 2009 και εντωμεταξύ και εμείς και εσείς κυρία Ματσιέ έχουμε ανασχοληθεί με τώρα με, τις, με τα στοιχεία του 2007 που δεν έχει δοθεί απαλλαγή και του 2008 και ακούσαμε από το διευθυντή τη ε, Ακαδημία κάποια στοιχεία που θα ήθελα να επαληθεύσω για άλλη μια φορά φυσικά, αλλά που εν πάση δεν με κάνουν και να πηδάω από την καρέκλα μου. Ερωτώ λοιπόν, εφόσον ναι, υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να συστήσουμε, με ποιον πρέπει να τα συστήσουμε. Ήθελα να επισημάνω ότι η εντολή για την απαλλαγή για το 2009 είναι ε, έκθεση της δικής μας ομάδας και πρέπει να την αναθέσουμε και μάλιστα πολύ σύντομα στον αρμόδιο συνάδελφο. Κυρία Γκρέσλε. Ναι, την εντολή βεβαίως θα την αναλάβουν ε, την είχαν μάλλον αναλάβει και με τον κύριο Φλιέρνερ οι σοσιαλιστές του 2007. Αυτό είναι και κομμάτι του προβλήματος. Γι' αυτό το επαναλαμβάνεται τώρα. Δεν νομίζω ότι η Βερονίκη έχει τίποτα να κερδίσει από αυτήν την έκθεση. Πρόκειται να εμείνει μέχρι τελευταία ρανίδο, Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και πρέπει να προχωρήσει η έκθεση, θέλουμε να δούμε αυτή η ιστορία να κλείσει με κάποιο τρόπο. Δεν συνεχίζεται έτσι αυτή η υπόθεση. Προπολογισμό του 2008 πρέπει να κλείσει νομότυπα όπως πρέπει από τη Βερονίκη. Και γι' αυτό θέλω στην επόμενη συνεδρίαση να περιμένουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λάβουμε τις σχετικές απαντήσεις, για να λάβουμε την, ε, τις απαντήσεις που θέλουμε, για να μπορέσουμε να κλείσουμε την υπόθεση αυτή, για να δοθεί απαλλαγή του 2008. Δεν υπάρχει προηγούμενο εδώ στην έκθεση και δεν προσπαθούμε να σφετεριστούμε την έκθεση της επόμενης χρονιάς ή να πάρουμε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω μας. Όχι. Θα μπορούσαμε να είχαμε προχωρήσει νωρίτερα. Δεν ξέρω. Ίσως αν είχαμε απαντήσεις. Δεν θα φτάσουμε, δεν θα κουμπίσουμε την έκθεση για το 2009 ούτως ή άλλως. Αυτό δεν είναι δική μας δουλειά. Σας διαβεβαιώ. Αλλά θέλω αυτή η υπόθεση το 2008 να κλείσει από τη Βερονίκ και να φτάσουμε στο σημείο στο οποίο μπορούν να κλείσουν αυτοί οι λογαριασμοί όπως πρέπει. Ας κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε μέχρι την προσεχή συνεδρίαση και ελπίζω να μπορέσει και η υπηρεσία και το Διοικητικό Συμβούλιο να μας δώσουν τις σχετικές απαντήσεις. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αλλάζει κάθε εξάμεινο. Είναι μέρος του προβλήματος Γι' αυτό το λόγο λειτουργεί όπω λειτουργεί αυτή η υπηρεσία. Γιατί αλλάζει κάθε εξάμεινο το Διοικητικό Συμβούλιο. Και ένα δείγμα εμπιστοσύνη σε τελευταία ανάλυση είναι το να παρουσιάζονται τα ονόματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα ε, ε, επί του διαδικτύου τέλο πάντων. Και ο κύριο Μίλλερ έχει υπογράψει έγγραφα. Γιατί τα έχει υπογράψει, με ποια ιδιότητα. Εάν ε, η Ματιέ. Ακούσαμε την κυρία Χολμάγερ. Ε, με όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα, ε, νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι ότι δεν μπορούμε να αποφανθούμε οριστικά. Ε, ορισμένες απαντήσεις δεν δόθηκαν. Και μάλιστα καθόλου δεν απαντήθηκαν κάποια ερωτήματα και επομένως θα πρέπει να ξαναβάλουμε το θέμα αυτό στη μέση και να το εμβαθύνουμε έχοντας περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Συμφωνείτε? Ωραία. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε ένα κοκτέιλ έξω. Ευχαριστώ.